So, colleagues, I, I would suggest that we start. Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Καθίστε παρακαλώ. Θα μ, μας παρουσιαστούν δύο μελέτες για την εκπρόπηση γυναικών και ανδρών στα νομικά επαγγέλματα στην Ένωση. Οπότε να δώσω απευθείας το λόγο στο στην Γιούτε Γιούτελάντ, που είναι η μόνιμη εισηγήτρια για τα θέματα εσόδας ανδρών γυναικών. Παρακαλώ Γιούτε, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ όλους ε, που είστε εδώ για το mainstreaming field. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντες εμπειρογνώμονες. Χαίρομαι που έχουμε διακεκριμένους ομιλητές που θα μας κάνουν διακεκριμένες ομιλίες. Η Μόνικα Νάτερ από το SPE Consulting της Βιέννης θα μας παρουσιάσει μια μελέτη για την εκπροσώπηση των γυναικών στα νομικά επαγγέλματα στην Ένωση και η κυρία Λίζα Ερουίν από το Πανεπιστήμιο Queens του Belfast θα συζητήσει επίσης ε, την ίδια μελέτη. Και έχουμε και την κυρία Jane Ellis από ε, την Ένωση Δικηγορικών Συλλόγων που θα μας παρουσιάσει επίσης το θέμα αυτό και χαίρομαι ιδιαίτερα που η γραμματεία μας εργάστηκε σκληρά για αυτό το σεμινάριο και για το ότι εκπώνησε και το Κοινοβούλιο αυτή τη μελέτη και συνεργαστήκαμε και με την Επιτροπή Γυναικών για αυτό το θέμα και κάναμε σημαντικό έργο. <clears throat> Στο άρθρο 8 του, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρονται τα θέματα mainstreaming φύλου και λέγεται ότι είναι οριζόντια προτεραιότητα. Σε όλε τι δραστηριότητε τη, λέει η Ένωση, να προσπαθήσει να καταργήσει τι ανισότητε και να προωθήσει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι λοιπόν θεμελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και χαίρομαι ιδιαίτερα και είμαι περήφανη που εμείς, ε, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, είμαστε στην πρωτοπορία της προώθησης των στόχων αυτών. Υπάρχει μάλιστα και ένα σχέδιο δράσης που εγκρίναμε τον περασμένο Μάρτιο όπου αναφέρουμε διάφορα θέματα μεταξύ των οποίων είπαμε ότι πρέπει πρώτα να δούμε τα του οίκου μας. Σε όλους τους τομείς της εργασίας των Επιτροπών τονίσαμε πρέπει να υπάρξει κατάρτιση των μελών της γραμματείας αλλά και των μελών και βασική και περαιτέρω κατάρτιση και για τις πολιτικές ομάδες και τους βοηθούς για τα θέματα αυτά. Είπαμε ότι θα κάνουμε ακροάσεις, ε, συζητήσεις ε, και άλλες εκδηλώσεις για τα θέματα αυτά, ούτω ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα γίνει κάθε αναγκαία προσπάθεια, ούτω ώστε να διασφαλίσουμε οι ομιλητές και οι που μας επισκέπτονται να είναι ισότιμα άνδρες και γυναίκες. Και επίσης για τους διορισμούς και την κατανομή εκθέσεων και γνωμοδοτήσεων οι πολιτικές ομάδες στην Επιτροπή μας. Άρα και εμείς οι ίδιοι πρέπει να το έχουμε κατά νου. Όλοι λοιπόν πρέπει να προσέχουμε ούτω ώστε να εκπροσωπούνται ισότιμα, ανάλογα δηλαδή και με τη σύσταση της Επιτροπής μας, τα δύο φύλλα. Επίσης όταν επιλέγουμε τους συνεργάτες μας, τα μέλη του προσωπικού, Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τα θέματα επίσης ισότιμη εκπροσώπησης των δύο φύλων σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει λοιπόν να ε, φροντίσουμε ούτω ώστε εμεί οι ίδιοι να τηρούμε αυτά τα οποία διακηρύσουμε. Και επίσης στην πολιτική μας δουλειά. Τονίζουμε ότι είναι σημαντικό σε ακροάσεις, ανταλλαγές απόψεων επίσης να υπάρχει ισότιμη εκπροσώπηση. και να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα από αυτού. Και στις αποστολές επίσης θα πρέπει να διδασκόμεθα από τις βέλτιστες πρακτικές επί του θέματος αυτού. Δεν θέλω να πω πολύ περισσότερα για να δώσω το λόγο στους ομιλητές μας. Αλλά πριν το κάνω, να ευχαριστήσω και τη Διεθνή Ένωση Δικηγορικών Συλλόγων για τη μελέτη αυτή που εξεπώνησε, η οποία με ενεθάρρυνε και με ενέπνευσε. Τι συνάγω εγώ από την μελέτη αυτή. Οι γυναίκες έχουν φτάσει σε πολύ ψηλό επίπεδο ικανοτήτων και κατάρτισης. Έχουν όλα τα αναγκαία προσόντα, ούτω ώστε να εκπροσωπούνται ισότιμα στα νομικά επαγγέλματα. Αλλά υπάρχουν ε, δομές που περιορίζουν τη συμμετοχή τους. και δεν μπορούν ε, να προχωρήσουν στη σταδιοδρομία τους και πολλές φορές αλλάζουν κατεύθυνση. Και όταν βλέπουμε ποια είναι η εκπροσώπηση στα υψηλότερα επίπεδα του νομικού, των νομικών επαγγελμάτων, πιστώνουμε ότι υπάρχουν περισσότεροι άνδρες. Αυτό είναι πρόβλημα. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι το συζητάμε θα μας βοηθήσει να το αλλάξουμε. Ευχαριστώ επίσης ε, όλους ε, όσοι εργάστηκαν για τη μελέτη του Κοινοβουλίου. Εξακολουθούν, ε, διαπιστώνει η μελέτη αυτή, να υπάρχουν προκαταλήψεις που παρεμποδίζουν την επαρκή πρόσληψη γυναικών. οι οποίες γυναίκες έχουν και προβλήματα συνδυασμού της προσωπικής με την επαγγελματική ζωή γιατί πρέπει να εργάζεται κανείς πολλές ώρες. Δεν υπάρχει επίσης διαφάνεια στους διορισμούς και τις προαγωγές. Δεν υπάρχουν επίσης αρκετοί για να στηρίζουν και να συμβουλεύουν τους νέους υπαλλήλους και δεν, έχουμε και επαρκής, δεν υπάρχει επαρκής ορατότητα των γυναικών ε, σε ανώτερες θέσεις στο νομικό επάγγελμα για να ε, χρησιμεύουν ως πρότυπα. Αλλά να σταματήσω εδώ. Αλλά θέλω να τονίσω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή την εκδήλωση και να σας δώσω το λόγο, η Πρόεδρος. Ξέρω, Γιούτε, πόσο ε, αγωνίζεσαι για το θέμα αυτό πόσο σε απασχολεί, πόσο χρόνο αφιερώνεις. Λοιπόν, να έχουμε τώρα τις δύο παρουσιάσεις των δύο μελετών. Πρώτα απ' όλα την ε, μελέτη από το δικό μας τμήμα πολιτικής ΣΥ και να, να δώσω κατευθείαν το λόγο στην κυρία Μόνικα Νάτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κυρίες και κύριοι, Αξιότιμοι κύριοι ευρωβουλευτές, θα μοιραστούμε την παρουσίασή μας εγώ με τη συνάδελφο. Θα σας δώσω στοιχεία για την μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε και για τα γενικά μας πορίσματα. Η συνάδελφος Λίζα Ερβάιν θα σας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά στοιχεία για συγκεκριμένα νομικά επαγγέλματα και θα ολοκληρώσω την παρουσίασή μας με συστάσεις ε, περί πολιτικής ώστε να, αυξηθεί, να βελτιωθεί η ισορροπία των φύλων στα νομικά επαγγέλματα. Ξέχασα να αναφέρω ότι κάθε μία σας έχει 10 λεπτά. 20 στο σύνολο. Εγώ προέρχομαι από την ε, συμβουλευτική εταιρεία OSB που έχει την έδρα της στη Βιέννα της Αυστρίας. Ασχολούμαστε με την απασχόληση, την κοινωνική πολιτική και την ισότητα των φύλων. Η συνάδελφος Λίζα Ιρβάιν προέρχεται από το Πανεπιστήμιο Queen's του Belfast που είναι μεταξύ των πρώτων πανεπιστημίων, στο 1% των πρώτων πανεπιστημίων σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Λίζα εργάζεται στο κέντρο για την προώθηση των γυναικών στην πολιτική εντός του τμήματος πολιτικής του Πανεπιστημίου. Μπορείτε να δείτε τα ονόματα των 7 ειδικών που εκπώνησαν αυτή τη μελέτη σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια. Ο στόχος ε, της μελέτης ήταν να δώσουμε μια εικόνα της ισχύουσας κατάστασης των φύλων στις διάφορα ε, επαγγέλματα στα κράτη-μέλη και να εντοπίσουμε και να εξετάσουμε τους λόγους για την υποδέστερη εκπροσώπηση των γυναικών στα νομικά επαγγέλματα. Η μεθοδολογία μας ε, ήταν να εξετάσουμε την υπάρχουσα ε, τεκμηρίωση, να διαβολευθούμε με τους ε, ενδιαφερόμενους φορείς και να συλλέξουμε δευτερογενή στοιχεία. Θέλω να αναφέρω κάποιες από τις μεθοδολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε. Τα τελευταία στοιχεία που ήταν συγκρίσιμα ήταν από το 2014 θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τα στοιχεία υπόκειται στην ερμηνεία των ερωτήσεων που θέτουν οι ερευνητές και, και καλύτερη ε, στοιχεία έχουμε από τα διάφορα κρατημέλη και δεν είναι πάντοτε απολύτως συγκρίσιμα ανάμεσα στα κρατημέλη. Ας πούμε, το θέμα του Ρέξ πλέγει δεν μπορούμε να το βρούμε αυτό σε όλες τις χώρες. Τώρα, υπάρχει έλλειψη ε, συνέπεια στις πληροφορίες, τα στοιχεία κάποιες φορές δεν υπήρχαν ή δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν και, εν πάση περιπτώσει, δεν υπήρχαν ε, για μια σειρά συναπτών ετών. Δεν έχουμε αρκετά στοιχεία όσον αφορά τους ε, δικηγόρους και δεν έχουμε και πλήρη στοιχεία για όλα τα νομικά επαγγέλματα. Η συλλογή των στοιχείων καλύπτει τους καθηγητές νομικών μόνο στην κατηγορία κοινωνικών επιστημών και σε σχολές όπως είναι η ψυχολογία, η οικονομία, οι πολιτικές επιστήμες. Οπότε τα στοιχεία δεν είναι απόλυτα όσον αφορά τους καθηγητές νομικής ή δικαίου. Τα βασικά προβλήματα που είχαμε να κάνουμε να αντιμετωπίσουμε ήταν ότι υπάρχει ενδο, μάλλον, κρυφή, κρυφή προκατάληψη στον αφορά τα φύλλα και αυτό σημαίνει ας πούμε για παράδειγμα την υπόθεση ότι οι άνδρες θεωρούνται ικανοί ενώ οι γυναίκες χρειάζεται επανειλημμένα να αποδείξουν τις ικανότητές τους Επίσης, πολύ συχνά συνδέεται για τις γυναίκες η μητρότητα με την έλλειψη προσήλωσης ή αφοσίωσης. Και οι γυναίκες εξάλλου θεωρούνται εξαιρετικά ήπιες ή εξαιρετικά σκληρές συχνά, ότι έχουν ε, λιγότερο, χαμηλότερες προδιαγραφές από ότι οι άνδρες και ότι δεν είναι εύκολο να δουλεύει κανείς με αυτές. Ε, ενώ υπάρχουν ε, δίκτυα ανδρών που παρέχουν υποστήριξη, μεν στους δε, από την τεκμηρίωση προκύπτει ότι για τις γυναίκες συχνά δεν υπάρχουν τέτοια δίκτυα υποστήριξης. Επίσης υπάρχει μια τάση να αναπαράγεται το ίδιο σύστημα ε, σημαίνει δηλαδή ότι περισσότερο οι άνδρες προτιμούνται για τις πιο ορατές ε, και τις πιο ψηλές θέσεις. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω την έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τις διαδικασίες ε, διορισμού είναι προφανές σε όλα τα νομικά επαγγέλματα, ιδιαίτερα στις υψηλότερες θέσεις, ότι οι γυναίκες δεν ε, ε, υποαντιπροσωπεύονται, αλλά σε διάφορους βαθμούς. Η συνάδελφος Λίζα Ερβάιν θα μπει στις λεπτομέρειες των συγκεκριμένων επαγγελμάτων. Με την άδεια της Προέδρου θα ήθελα να της δώσω το λόγο, παρακαλώ. Η ποσοτική πτυχή αυτής της μελέτης ε, στην ουσία βασίστηκε στη συλλογή στοιχείων από τις στατιστικές υπηρεσίες των ε, κρατών μελών. Έχουμε στοιχεία για το δικαστικό κλάδο, εισαγγελικό ε, προσωπικό, αλλά και προσωπικό των δικαστηρίων. Τα στοιχεία αυτά που έχουμε ε, δεν είναι απόλυτα ανεξάρτητα, ε, ε, μάλλον δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρα. Και εδώ έχουμε και στοιχεία από τη Eurostat όσον αφορά τους φοιτητές στις διάφορες σχολές νομικών. Κατά μέσο όρο επικρατεί πλειοψηφία στους δικαστές σε αυτό το επίπεδο κατά 59% το 2014. Ας πούμε για στα πρωτοδικεία, Ενώ εν γέννη επικρατούν οι άνδρες, οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία πάνω από το 60% σε αρκετές χώρες. Για τους δικαστές του Δικαστηρίου αλλάζει η εικόνα. Δύο τρίτα άνδρες και ένα τρίτο γυναίκες. Ε, Λετωνία, Λουξεμβούργο, Ρουμανία και Σλοβακία μόνο ε, έχουν πλειοψηφία γυναικών το 2014. Οι ε, γυναίκες δηλαδή κάπου χάνονται στη διαδικασία αυτή. Είναι καλύτερα εκπροσωπούμενες στα χαμηλότερες βαθμίδες και πολύ λιγότερο εκπροσωπούνται στις ψηλότερες βαθμίδες του δικαστικού σώματος. Παρόμοια εικόνα για τους εισαγγελείς. Στα πρωτοδικεία, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 41% κατά μέσο όρο, ε, ε, οι άντρε το 41% και οι γυναίκες το 59%. Αυτό σε όλες τις χώρες εκτός από τη Σλοβενία. Εκεί οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 74% των εισαγγελέων πρωτοδικών. Και στη Γερμανία έχουμε περισσότερους άντρες από την άλλη μεριά. Σε επίπεδο του δικαστηρίου έχουμε υπερεκπροσώπηση των ανδρών στους εισαγγελές. Πάνω από 60% είναι άνδρες. Το Βέλγιο ε, έχει ένα προφίλ που είναι αποκλειστικά άνδρες. Στη Σουηδία από την άλλη μεριά οι άνδρες εισαγγελείς μειώνονται ως ποσοστό τα τελευταία χρόνια από το 60% στο 38%. Στη Δανία αυτό το ποσοστό των γυναικών έχει αυξηθεί και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 77%. Στο Λουξεμβούργο επίσης έχουμε μια πλειοψηφία 62% γυναικών εισαγγελέων στο Ανώτατο Δικαστήριο. Μια μικρή πλειοψηφία βρίσκουμε στη Σλοβενία και στη Λετωνία επίσης. Για το μη δικαστικό προσωπικό που εργάζεται στα δικαστήρια έχουμε πολλά επαγγέλματα και ένα μεγάλο αριθμό υπαλλήλων. speaker, ε, τεχνικό, διοικητικό προσωπικό, γραμματής κλπ. Εδώ έχουμε ίση περίπου εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών, ε, ενώ έχουμε περίπου ίση, ίση εκπροσώπηση στις χαμηλές βαθμίδες ε, για το δικαστικό προσωπικό, εδώ έχουμε κυρίως γυναίκες. Μόνο στο Λουξεμβούργο έχουμε περισσότερους άνδρες από ό,τι γυναίκες. στοιχεία για τις γυναίκες δικηγόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η, μιλούμε για τους δικηγόρους όπως αυτοί, αυτοί αναγνωρίζονται σε κάθε χώρα. Έχουμε σταδιακή αύξηση του ποσοστού των γυναικών δικηγόρων. Μεγαλύτερο η ποσοστία αύξηση στην Βουλγαρία κατά 18%, Ελλάδα 17% και Σλοβενία 16%. Εκεί έχουμε εξασφαλίσει την ισότητα στην εκπροσώπηση των δύο φύλων. Στις χώρες του Common Law ε, έχουμε κυρίως άνδρες, δικηγόρους 75%. Σε Έχουμε όμως μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις χώρες. 11 κράτη-μέλη, κυρίως της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ε, έχουμε περισσότερε περισσότερες ε, γυναίκες συμβολιογράφους, ε, για παράδειγμα Πολωνία, Λιθουανία κλπ. Στη Δυτική Ευρώπη, την άλλη μεριά, οι συμβολιογράφοι είναι κυρίως άντρες. Στην Αυστρία 91% των συμβολιογράφων είναι άντρες και 82% στη Γερμανία. Μόνο στο Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και τη Σλοβενία έχουμε περίπου ίση εκπροσώπηση των δύο φύλων ε, σπουδές, ε, ε, νομικές σπουδές ήταν κυρίως ε, ψηλής εκπροσώπησης γυναικών ε, τα τελευταία χρόνια. Στη Βαλτική, στις Βαλτικές χώρες και στην Κροατία είναι 70% γυναίκες, 30% άνδρες αυτοί που παίρνουν πτυχίο νομικής. Όμως στα διδακτορικά η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική. Στις περισσότερες ε, χώρες περισσότεροι άνδρες παίρνουν διδακτορικό το 2015 τουλάχιστον. Ε, Βουλγαρία, Αυστρία, Ουγγαρία και Σλοβενία είναι μόνο μόνοι χώρες που υπάρχουν, έχει πλειοψηφία γυναικών. Να δώσω, αν με επιτρέπετε, το λόγο στη συνάδελφό μου ξανά. Τα δεδομένα της μελέτης ε, δείχνουν μια ανισορροπία στις ψηλές βαθμίδες ε, και μια οριζόντια διάκριση σε αυτά τα επαγγέλματα. Ε, το διοικητικό προσωπικό στα δικαστήρια είναι περισσότερο γυναίκες για παράδειγμα. Χρειάζεται λοιπόν να αλλάξουμε λίγο την οτροπία και τις πρακτικές έτσι ώστε να, διατηρήσουμε, να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ένα περιβάλλον όπου τόσο γυναίκες όσο και άντρες θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για να κάνουν σταδιοδρομία. ε, συστάσεις για το άμεσο μέλλον που προκύπτουν οι εξής. Πρώτον, ε, η γενίκευση καλών ε, πρακτικών ε, για την ενθάρρυνση των ε, κρατών ε, μελών να ξεκινήσουν προγράμματα για την εξασφάλιση ισότητας των δύο φύλων στα νομικά επαγγέλματα. Χρειάζεται μια θετική προσέγγιση με, μέσω σχεδίων δράσης αναχώρα μαζί με την Επιτροπή ΦΑΜ και την Γενική Διεύθυνση Justice της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την δημιουργία μιας ε, μεθόδου παρακολούθησης ε, της εξέλιξης, των εξελίξεων ε, στα νομικά επαγγέλματα. Η συζήτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει και την ενθάρρυνση των κρατών μελών να θέσουν χρονοδιαγράμματα και στόχους. ωστόσο θα μπορούσε να είναι ένα από τα εργαλεία που θα χρησιμοποιούν τα κρατη Ε, κίνητρα για την ε, δημιουργία δικτύων ισότητας ε, των δύο φύλων στα νομικά επαγγέλματα και δικαστικά επαγγέλματα και αντικειμενικές και μη μεροληπτικές διαδικασίες πρόσληψης ιδιαίτερα στις χώρες του αγγλοσαξονικού δικαίου. Κάποιες άλλες συστάσεις για τα δεδομένα. Τα δευτερογενή δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν δεν ήταν πάντοτε ε, συνεπή μεταξύ τους. Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα, χρειάζεται, αυτό το φαινόμενο, χρειάζεται ένα ενιαίο πλαίσιο για την ε, συλλογή στατιστικών στοιχείων που θα λαμβάνει υπόψη τις ε, διαφορές ανάμεσα στα επαγγέλματα και τις ε, χώρες. Πιο εμπειρικά δεδομένα είναι επίσης απαραίτητα. Χρειάζεται επίσης ε, συλλογή περισσότερων δεδομένων για συγκεκριμένα ε, ζητήματα όπως οι αμοιβέ ή θέματα διάκρισης ε, φύλου, οριζόντιας διάκρισης φύλου, ε, η, εξειδίκευση σε διάφορους τομείς, αριθμό ανδρών και γυναικών στα διάφορα, στα, στα, βαθμίδες, χρόνους προαγωγής κλπ. Η απουσία ε, δεδομένων αναφύλω για, τους, ε, το πάγγελμα του καθηγητή στη μέση και ανώτερη εκπαίδευση είναι επίσης πρόβλημα. Η Επιτροπή Νομικών ε, Θεμάτων, Νομικών Υποθέσεων θα μπορούσε να συζητήσει με την Κομισιόν ε, για το θέμα της ε, αναφύλω ε, κατανομής των δεδομένων που ήδη υπάρχουν σε, στο, για για τους καθηγητές ε, δικαίου. Συστάσεις για την νομική εκπαίδευση περιλαμβάνουν ε, ανάπτυξη συστάσεων για ένα κοινό πλαίσιο ορολογίου εκπαιδευτικού προγράμματος, συστηματική συμπερίληψη του φύλου ε, ως οριζόντιο θέμα στις νομικές ε, σπουδές. Τα θέματα του φύλου μπορούν, μπορούν να συμπεριληφθούν ως οριζόντιο μάθημα σε όλες τις δραστηριότητες των νομικών σπουδών. Ευχαριστώ πολύ για την ε, προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Πριν περάσω ερωτήσεις, θα πρότεινα να ακούσουμε και τη δεύτερη έκθεση και μετά να δώσουμε το λόγο για Έχουμε την κυρία Τζέιν Ellis που είναι διευθυντής δημοσίων σχέσεων στην Διεθνή Ένωση Δικηγορών Συλλόγων και θα μας μιλήσετε για τις γυναίκες που ασχολούνται με το εταιρικό δίκαιο ως δικηγόροι. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να συζητήσω την εκθεσή μας την οποία ελπίζουμε να δημοσιεύσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Αρχές Δεκεμβρίου το αργότερο κάναμε λοιπόν μία μελέτη φέτος που στείλαμε σε όλα μας τα μέλη όπου θέλουμε πληροφορίες για το πώς οι δικηγόροι αποχωρούν και επανέρχονται στις, ε, στα δικηγορικά γραφεία που ασχολούνται με το εταιρικό δίκαιο. Κάνουμε μια σειρά από μελέτες Μελετήσαμε και την έκθεση που μόλις ε, μας στείλατε. Ευχαριστώ πολύ. Και τα πορέσματά μας βασίζονται σε όλα αυτά που ψάξαμε. Οι περισσότερες απαντήσεις ήρθαν από γυναίκες που ασχολούνται με το εμπορικό δίκαιο. Πολλές προφορίες λοιπόν που έχουμε ασχολούνται με γυναίκες που εργάζονται σε δικηγορικά γραφεία, όχι, όχι γυναίκες. Να το έχουμε λοιπόν αυτό υπόψη μας. Με συγχωρείτε εάν ε, μιλάω πολύ γρήγορα. Πείτε μου να, ε, να μιλήσω πιο αργά. Πολλοί λένε ότι γίνεται όλο και πιο θηλυκό ε, ε, θηλυκός ο κόσμος που εργάζονται ε, σε νομικά επαγγέλματα αλλά αυτά είναι ανοησίες ε, μόνο στα πολύ κατώτερα επίπεδα υπάρχει κάτι τέτοιο από όλα όσα λάβαμε μόνο 30% είπαν ότι είναι συνδιοκτήτε, αλλά μόνο 14% από τι γυναίκε στα δικηγορικά γραφεία είπαν ότι συμμετέχουν και στο μετοχικό κεφάλαιο των δικηγορικών γραφείων. Και θα σας δώσω μια σειρά από λόγους γι' αυτό. Το πρώτο που προέκυψε και από τη δική μας μελέτη, αλλά και από τις, ε, τα στοιχεία που συλλέξαμε, είναι ότι δεν λειτουργεί σωστά η δομή των δικηγορικών γραφείων και ο τρόπος λειτουργίας τους. Ε, δεν υπάρχουν, για παράδειγμα, ελαστικές μορφές απασχόληση. Γιατί παίζει ρόλο και θα ήθελα να ακούσω περισσότερα. Οι γυναίκες εισέρχονται στον τόπο εργασία των ανδρών που λειτουργούσαν καλά για τους άνδρες. Άρα οι γυναίκε πρέπει να προσαρμοστούν ε, στην δομή τη εργασία. που έργα που επιβάλλονται ε, από άτομα που δεν ξέρουν πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα, δεν συμμετέχουν. Αν θέλουμε να βελτιωθεί η συμμετοχή των γυναικών, τότε θα πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά πώς λειτουργούν τώρα οι δομές και οι συνήθειες, οι εργασιακές συνήθειες. Να δούμε ποια είναι τα προβλήματα. Δηλαδή, οι πολιτικές για να προωθήσουμε τις ε, γυναίκες είναι απλώς για να βολέψουμε τις γυναίκες, αλλά το θέμα δεν είναι Είναι πολύ δύσκολο να σα παρακολουθήσουν οι διερμηνεί. Α, ωραία, θα επιβραδύνω. Λοιπόν, δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των πολιτικών για την πολυμορφία γίνονται για να απλώς βολευτούν, προσαρμοστούν οι γυναίκες στις υπάρχουσες συνθήκες. Όπως έμπαιναν όλο και περισσότερες γυναίκες στο νομικό επάγγελμα, στα νομικά επαγγέλματα, τα νομικά επαγγέλματα, οι δικηγορίες συγκεκριμένα, άλλαζαν πολύ από επιχειρήσεις ε, νομικών θεμάτων τα μεγάλα δικηγορικά γραφεία έγιναν στην ουσία νομικές επιχειρήσεις με διεθνή παρουσία. Αυτό σημαίνει ότι για παράδειγμα εργάζονται πολύ περισσότερες ώρες τις οποίες χρεώνουν στους πελάτες. Για παράδειγμα στα 1990 τα αμερικανικά δικηγορικά γραφεία πρότειναν ότι ε, θα έπρεπε το πολύ να κάνουν 1.300 ώρες εργασίας ε, οι δικηγόροι. Και μετά πέρασαν στις 1.800 και τώρα στις 2.200. Χωρίς να έχει διπλασιαστεί ο χρόνος, ε, ο αριθμός των ωρών ενός έτους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρεώσεις 40 ώρες τη βδομάδα. Το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να εργαστεί 50, 60 ή 70 ώρε για να επιτύχει να χρεώσει 40. Και η τεχνολογική πρόοδο και οι ευέλικτε μορφέ εργασία ε, σημαίνουν ότι εργάζεται κανεί περισσότερο. Μπορεί να πάρει τα παιδιά σου στον τόπο εργασία ή να πάρει δουλειά στο σπίτι. Αλλά αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει χρόνος χωριστά για την οικογενειακή ζωή. Και Υπάρχουν όλο και λιγότεροι συνειδιοκτήτε στα δικηγορικά γραφεία, ενώ οι περισσότερες γυναίκες είναι απλώς μισθωτοί στα δικηγορικά γραφεία. Αυτό σημαίνει ότι όσοι εργάζονται σε ένα δικηγορικό γραφείο αφιερώνουν 100% του χρόνου τους στη δουλειά τους. Αυτό είναι τρομερά ε, ανδροκρατική αντίληψη που εξαιρεί τι γυναίκε. Σε ένα άρθρο που διάβασα, αυτή η γυάλινη οροφή στην οποία αναφερθήκατε, οδήγησε τι γυναίκε σε αδιέξοδο. Λέτε επίση ότι κάποιοι θα μπορούν να είναι μέντορες, να δίνουν συμβουλές στους νέους εργαζόμενους. Ναι, είναι σημαντικό για να ε, εξοικειωθεί κανείς με τον τόπο εργασίας και να δημιουργήσει δίκτυα και να έχει κάποιον να συζητήσει τις ε, προοπτικές ανέλυξης. Αλλά όποιο δικηγόρο θέλει να προωθηθεί, δεν χρειάζεται απλώ συμβουλέ. Χρειάζεται πραγματικά έναν σύμμαχο, κάποιον που να του αναλαμβάνει. Τι σημαίνει αυτό. Η διαδικασία ένταξη σε ένα δικηγορικό γραφείο είναι συνήθως διαφανής. κανεί αίτηση, συνεντεύξει ε, από κάποιους νέου δικηγόρους, από κάποιου από το τμήμα προσωπικού, από κάποιους από τους ετέρους και μετά σε παίρνουν ή όχι. Αλλά ξεκινάει αυτή η διαδικασία παροχής συμβουλών. Αλλά αν περάσει μερικά χρόνια σε ένα δικηγορικό γραφείο, πρέπει να σε βοηθήσει κάποιο από του ιδιοκτήτε, κάποιο από του εταίρου, του partners στα αγγλοσαξονικά. Πρέπει δηλαδή να σε στηρίζουν απόλυτα. Και εδώ δεν κάνει αίτηση. Για να γίνει συνειδιοκτήτη, ε, πρέπει να σε προτείνουν ορισμένοι από του ίδιου συνειδιοκτήτε. Και ε, κατόπιν, αφού σε ορίσουν, σε βοηθούν να φτάσει σε αυτό το επίπεδο και για να φτάσει, παρακολουθεί από ορισμένου από του κύριου ε, δικηγόρου. Και έτσι μόνο γίνεσαι συνειδιοκτήτη. Και ένα ιδιοκτήτης φυσικά μετά θα διαλέξει κάποιον που να του μοιάζει. Και αυτό δεν αφορά μόνο τι γυναίκες. Άρα και για άτομα από, άλλες, από άλλη εθνική προέλευση και άλλες τέτοιε μειονότητε. Αυτό είναι κάτι το κοινό και πρέπει να αλλάξει. Γιατί αυτή η διαδικασία δεν είναι επίσημη και σίγουρα δεν είναι διαφανής. Είναι ιδιαίτερα αδιαφανής. Επίσης υπάρχει πάρα πολύ σεξουαλική παρενόχληση στα δικορικά γραφεία εξακολουθεί να υπονομεύει οποιαδήποτε πρόοδο επετεύχθη για την προώθηση των γυναικών. Και επίσης και η παρενόχληση γενικότερα, η εργασιακή παρενόχληση. Περίπου 50% και των ανδρών και των γυναικών ε, στα ερωτηματολόγια μας ε, μας είπαν ότι πιέζονται και παρενοχλούνται. Και επίσης, από ό,τι φαίνεται αυτά δεν ισχύουν μόνο για τους δικηγόρους. Όλες οι γυναίκες που εργάζονται σε επενδυτικά γραφεία, για παράδειγμα, έχουν παρόμοιες εμπειρίες. Εξετάσαμε σταδιακά μέσω ερωτηματολογίων και αυτούς τους τομείς για να δούμε τι κάνουν για να υπερβούν κάποιες από τις ανισότητες που βρίσκουμε στα δικαιωρικά γραφεία και διαπιστώσαμε ότι η κατάσταση είναι ίδια. Άρα δεν είναι μόνη η δικηγορία ε, που αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα αυτή ε, παρουσίαση που μας κάνετε, κυρία Έλλης. Αυτό που μας περιγράψετε είναι η πραγματική ζωή. Με εντυπωσίασε μάλιστα ο αριθμός των εργάσιμων ωρών που αναμένεται κανείς να δουλέψει σε ένα χρόνο. Προσπάθησα να το μετατρέψω σε ημερήσιες ώρες εργασίας και δεν το κατάφερα. Αλλά η διπλανή μου είπε πάνω από 12 ώρες την ημέρα πάνω από 12 ώρες την ημέρα πρέπει να δουλεύει κανείς για να χρεώσει αυτά. Έχουμε τρελαθεί τελείως μου φαίνεται. Τώρα ακούσαμε τις δύο παρουσιάσεις λοιπόν και όποιος θέλει μπορεί να θέσει ερωτήσεις. Εγώ έχω μία άμεσα, αν μου επιτρέπετε. Προς την κυρία Νάτερ, στη μελέτη σας αναφέρατε συχνά τις ε, χώρες του αγγλοσαξονικού δικαίου και τις υπόλοιπες. Και στις ε, χώρες ε, του common law είδαμε σε κάποιες περιπτώσεις ότι οι άνδρες υπερ-αντιπροσωπεύονται στις υψηλότερες βαθμίδες. Έχετε κάποια εξήγηση γι' αυτό. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά ανάλογα με τον τύπο δικαίου. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Μάλιστα, ο λόγος είναι ότι στις ε, χώρες common law ε, το κύρος είναι πολύ διαφορετικό. Η διαδικασία του να φτάσει κανείς σε τέτοιες ε, θέσεις είναι διαφορετική. στην υπηρετική Ευρώπη ε, είναι πιο σαφείς οι διαδικασίες, πιο ξεκάθαρες οι διαδικασίες για το να φτάσει κανείς σε θέσεις στο δικαστικό σώμα και στα δικαστήρια. Να μιλήσω γερμανικά καλύτερα. Ε, ναι, βεβαίως, ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να πω ότι η διαδικασία για να εργαστεί κανείς στα δικαστήρια στις χώρες αστικού δικαίου είναι πιο διαφανής. Υπάρχει σαφής διαδικασία, ενώ στις χώρες του common law όλα αυτά γίνονται μέσω δικτύων και συστάσεων. Ιδιαίτερα οι προαγωγές. Και ακριβώς αυτά τα δίκτυα, στα οποία αναφέρθηκαν και οι προηγούμενες ε, ομιλήτριες, αυτά τα δίκτυα δημιουργούνται από νωρί όταν μπαίνει κανείς στο επάγγελμα και οι άνδρες αλληλοϊποστηρίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά δεν είναι μόνο θέμα φίλου. Είναι θέμα και ε, εθνοτικής προέλευσης και το αποτέλεσμα είναι ότι ο καθένας προωθεί τους ομοίους του. Και τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι πρέπει να γίνει μια ατομή εδώ. Να γίνει πιο διαφανής η διαδικασία, ούτως ώστε να υπάρχουν δυνατότητες για όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ιδιότητα. Εγώ δεν έχω ερώτηση, απλά θέλω να πω ότι πιστεύω πως τα απορίσματα σας είναι πάρα πολύ σημαντικά για την Επιτροπή μας και οι δύο μελέτες μας τις εξηγήσατε πολύ καλά και έχουμε και κάποιες συστάσεις για το τι θα μπορούσε να γίνει και πιστεύω ότι εμείς ως Επιτροπή θα πρέπει να ακολουθήσουμε και να δώσουμε μια συνέχεια σε όλα αυτά. Θα σύστηνα λοιπόν στους συναδέλφους να δουλέψουμε πάνω σε αυτό στο μέσο του προγράμματος δράσης για το gender mainstreaming θα προσπαθήσω να δω τι μπορούμε να κάνουμε και να δουλέψουμε περισσότερο σε σχέση με τα όσα έχουμε ήδη ε, εγκρίνει. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τις συμβολές σας. Για μένα ως εισηγήτρια για το gender mainstreaming ήταν πάρα πολύ σημαντικά αυτά που άκουσα και έχω και συναδέλφους εδώ που θα βοηθήσουν να διαδοθούν αυτά τα πορίσματα αλλά και σε όσους λείπουν θα προσπαθήσουμε να τους ενημερώσουμε. Ευχαριστώ. Τέλεια το συμπέρασμά σου. Να ευχαριστήσω και εγώ τις ομιλήτριές μας. Η Κομισιόν έχει κάτι να μας πει. Σε συγγνώμη που δεν σας έδωσα το λόγο. Ναι, βεβαίως ε, μπορείτε να πάρετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Όντως πρόκειται για πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες που ε, ακολουθούν τις ίδιες γραμμές ε, με αυτά που εμείς κάνουμε στην DG Justice ε, στο τμήμα για το ειρήντα των φύλων. Προσπαθούμε να εστιάσουμε σε αυτά τα θέματα, ιδιαίτερα αυτό που τονίσατε εδώ. Δεν αφορά μόνο την τομεακή διακρίση και διαχωρισμό, αλλά θα πρέπει να πάμε πιο βαθιά στους διάφορους κλάδους, να καταλάβουμε ποιες είναι οι διαφορές και πώς λειτουργεί αυτό το η γυάλινη οροφή ή άλλη φραγμή το Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων που αναφέρθηκε πριν έχει κάνει παρόμοιο προβληματισμό και μελέτη, αλλά κυρίως ε, σε άλλους τομείς όπου πάλι οι γυναίκες ε, και οι άνδρες δεν έχουν την ίδια πορεία. Και σήμερα το πρωί είχαμε το συνέδριο για τα θεμελιώδη δικαιώματα που κυρίως εστιάσαμε στις γυναίκες σε ταραχώδες καιρούς και Μιλήσαμε για τη γενική αχειραφέτηση καθώς και το, τη διαφορά μισθών ανάλογα με το φύλλο. Πιστεύω ότι και στις δύο σας μελέτες τονίζετε αυτές τις συζητήσεις, ε, απηχούνται τα θέματα που εσείς ε, αναφέρατε και εκεί υπάρχουν ένα σωρό διαφορετικοί φραγμοί, όπως για παράδειγμα δεν έχει να κάνει αυτό μόνο με το, τη σταδιοδρομία, αλλά και για πραγματικά εμπόδια, όπως αναφέρθηκε ότι χρειάζεται κανείς να έχει έναν υποστηρικτή και μπορεί να είσαι άτυχος ή όχι. Και αυτό που μου αρέσει πολύ επίσης στη μελέτη σας είναι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και ιδιωτική ζωής και πώς μπορείς να κάνεις κάτι για να μπορέσει να έχει και ιδιωτική ζωή, ιδιαίτερα με αυτό το μακρά ωραίο εργασία και τις ευέλικτες μορφές εργασία Μπορεί κανείς να πάει και λίγο σπίτι του, αλλά όσοι έχουν φροντίδα άλλων, που πράγμα που σημαίνει γυναίκες κυρίως ακόμα, ε, δυσκολεύονται. Καλό θα ήταν λοιπόν να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία για να προβληματιστούμε για την ισότητα των φύλων στην κοινωνία μας και σε αυτή την περίπτωση ε, στα νομικά επαγγέλματα. Καλωσορίζουμε λοιπόν τη μελέτη σας και θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε και θα ρίνουμε και το Ευρωκοινοβούλιο να ακολουθήσει, να, να συνεχίσει τη μελέτη αυτή. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, λέει η Πρόεδρος. Πρέπει να ενώσουμε τις προσπάθειές μας, πιστεύω όλοι οι άνθρωποι καλή βούληση, καλή θέληση να συνεργαστούμε. Ναι, ξέχασα να σα πω ότι χθες ξεκίνησε ένα πρόγραμμα δράση για τη διαφορά μισθών με βάση το φύλλο. Ορισμένα στοιχεία από αυτά που αναφέρθηκαν σε αυτέ τι μελέτε, αναφέρονται και εκεί. Προσπαθούμε να έχουμε δηλαδή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράση για να αντιμετωπίσουμε κάποια από αυτά τα θέματα που σχετίζονται με την ανισότητα των φύλων στην αγορά εργασία. Σα ευχαριστώ πολύ και είμαι βεβαία ότι και εμείς θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτό το πρόγραμμα δράσης να προχωρήσει για να προοδεύσουμε σε αυτό το θέμα. Γρήγορα, η Σίλβια. Ευχαριστώ. Τώρα δεν θέλω να μακρηγορήσω, αλλά συζητάμε για το ότι οι υποψήφοι, για παράδειγμα, από τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα για το δικαστήριο. Έτσι μπορούμε να προωθήσουμε τη θέση των γυναικών. Αλλά ο χρόνος που μας παίρνει για να γίνει αυτό είναι πάρα πολύ και είναι καλό που έχουμε μελέτες για να επιταχύνουμε τα πράγματα. Πρόεδρος. Μα ναι, καταλήγουμε πάντα στο ίδιο συμπέρασμα. Το θέμα είναι όμως να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις. Θα συνεχίσουμε να ασχολούμεθα με το θέμα αυτό και είμαι σίγουρο ότι η Γιούτα θα κάνει ό,τι μπορεί για να προωθήσει την ισότητα των φίλων. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας και κλείνουμε αυτό το θέμα της μερίσιας διάταξης και περνάμε στο σημείο 30 της ημερήσιας διάταξης. Το οποίο είναι μια συνεδρία εργασία workshop, για το εάν η διαμεθοριακή, το διαμεθοριακό καθεστώ κληρονομικής διαδοχής είναι πρόκληση ή όχι. Σίγουρα είναι πρόκληση. Θα μπούμε λοιπόν στις λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας εργασίας. Λοιπόν, είναι ιδιαίτερα δυσχερές το θέμα αυτό. Η Νομική Επιτροπή ε, έχει ασχοληθεί σχετικά πρόσφατα. Ο κανονισμός για την κληρονομική διαδοχή άρχισε να ισχύει πριν από δύο χρόνια. Ήταν ο λόγος που μας απασχόλησε αυτό το θέμα. Μέσω αυτής της συνεδρίας εργασίας θέλουμε να δούμε πώς έχει πάει σε μια πρώτη φάση η εφαρμογή του κανονισμού αυτού με στόχο να κανονίσουμε αν λειτουργεί σωστά εάν παρέχει νομική βεβαιότητα, απλούστευση και προβληψιμότητα. Για τους πολίτες. Έχουμε εδώ διάφορους ε, ειδικού που θα μας μιλήσουν για το κατά πόσον ε, λειτουργεί σωστά αυτός ο κανονισμός. Και πρώτα απ' όλα να δούμε αν λειτουργεί και η τεχνολογία. Γιατί σας παρακαλούμε να δούμε τώρα μία σύντομη παρουσίαση από τον δόκτορα Τζόναθαν Φίτσον του Πανεπιστήμιου του Αμπετζίν για τα κύρια πορίσματα της μελέτης για την αποδεικτική ισχύ των δημοσίων εγγράφων ε, ε, στις χώρες της Ένωσης στα πλαίσια της κληρονομικής διαγωγής. Κάτι το οποίο παρήγγειλε το Τμήμα Πολιτικής ε, για τα θέματα πολιτών και θεσμικών θεμάτων. Η μελέτη αυτή είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τα θέματα των διαμεθοριακών κληρονομικών διαδοχών. Για να δούμε λοιπόν τώρα το βίντεο. Χαίρετε. Είναι μια έκθεση εδώ για την ε, μελέτη για την κληρονομική διαδοχή που έγινε το 2015-2016 από τον καθηγητή Πολ Μπέμοντ, τον δόκτωρα Φίτσον και την κυρία που είναι του κέντρου του Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου του Πανεπιστήμιου του Αμπερντίν. Υπάρχει ένας ε, σύνδεσμος για να το δείτε. Εγώ θα παρουσιάσω την έκθεση, το όνομά μου είναι ε, Dr. Jonathan Fitcher. Ποιο είναι το πλαίσιο για τη μελέτη. Ο κανονισμό για την οικονομική διαχωγή τη Ένωση, ο 650 κάθε 2012, έχει στόχο να εναρμονίσει το ιδιωτικό διεθνέ και του κανόνε για τη σύγκρουση δικαίου για τα 25 κράτη-μέλη που συμμετέχουν για θέματα που έχουν να κάνουν με τι οικονομικέ διαδοχέ. 22 από τα κράτη-μέλη Μία τέτοια ε, διαδοχή μπορεί να βασιστεί σε ένα ή άνω του ενός δημόσια έγγραφα. Άρα χρειαζόμαστε αυτό τον κανονισμό, ούτω ώστε να έχουν τα ίδια αποτελέσματα, ίδια νομικά αποτελέσματα τα έγγραφα αυτά. Ο κανονισμός αυτός έχει δύο διατάξεις, τα άρθρα 59 και 60, που επιτρέπουν διαφορετικά νομικά αποτελέσματα των ε, δημοσίων εγγράφων αυτών, που τους επιτρέπουν να πάνε από το κράτος μέλος όπου ε, δημιουργήθηκαν για να περάσουν στα 24 άλλα κράτη-μέλη. Εάν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι είναι ε, δημόσιο έγγραφο και εάν επίσης ε, ε, πληρεί τον κανονισμό και τότε μπορεί να ενταχθεί στο άρθρο 59. Το άρθρο 59 που είναι το υποκείμενο της μελέτης απαιτεί τα άλλα κράτη-μέλη με βάση μια στενή εξαίρεση δημοσίου συμφέροντος να αποδέχονται αυτό το έγγραφο και να του δίνουν τα ίδια αποδεικτικά αποτελέσματα και ισχύ που θα είχε εάν είχε γραφτεί στο δικό του κράτος μέλος. Αυτή η αποδοχή είναι μια νέα νομική έννοια για το ενωσιακό δίκαιο και μια νέα ε, νομική έννοια για τα εσωτερικά δίκαια. Οι λόγοι για τη μελέτη. Για να ισχύει το άρθρο 59 όπως ε, το προβλέπει ο κανονισμός, οι αρχές των άλλων κρατών μελών πρέπει πρώτον να ε, διαπιστώσουν ότι έχει εκδοθεί ένα από ένα δημόσιο έγγραφο και να δουν τι αποδεικτική ισχύ έχει στο κράτος μέλος προέλευσης και κατόπιν να αποφασίσουν με μία εξαίρεση για λόγους δημοσίου συμφέροντος να δουν πώς ακριβώς θα ε, αναπαραχθεί στο δικό τους νομικό καθεστώς. Το άρθρο 59 του κανονισμού μας δίνει ένα πλαίσιο κανόνων, αλλά δεν δίνει την αναγκαία προφόρηση για τις αρχές των άλλων κρατών μελών για να κάνουν τα βήματα α έως c που ανέφερα. Ο εφαρμοστικός κανονισμός 1329 του 2014 δίδει, στο παράδειγμα 2, μια εθελούσια, ε, ένα εθελούσιο έντυπο το οποίο θα μπορούσε να συνοδεύσει ένα τέτοιο έγγραφο από το ένα στο άλλο νομικό σύστημα. Αυτή η μελέτη ε, επιχειρεί να βοηθήσει τα βήματα α έως ε, σ δίδοντας προφορίες για το είδος των δημοσίων εγγράφων που παράγονται σε κάθε κράτος μέλους και τα διάφορα ε, αποδεικτικά αποτελέσματα που έχουν και οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη πολιτική στα διάφορα κράτη-μέλη. Αυτή η βοήθεια είναι σημαντική για τη Σουηδία, τη Φιλανδία και την Κύπρο, όπου δεν υπάρχουν εθνικά δημόσια έγγραφα διαδοχής. Άρα δεν υπάρχει καμία εμπειρία από το πώς θα αντιμετωπίζονται τα ξένα παρόμοια έγγραφα. Η μεθοδολογία τώρα. Εμείς απευθυνθήκαμε σε εθνικούς εμπειρογνώμονες για όλα τα 25 κράτη-μέλη που συμμετέχουν σε αυτόν τον κανονισμό. Τους ζητήσαμε να μας ε, στείλουν ένα ε, συμπληρωμένο αναλυτικό ερωτηματολόγιο, να μας πούν ποια είναι η δημόσια χρήση αυτών των, ε, η, η εσωτερική χρήση αυτών των δημοσίων εγγράφων. Και επίσης ψάξαμε για στοιχεία για την οποιαδήποτε χρήση αυτής της εξαίρεσης δημοσίου συμφέροντος, το λεγόμενο Lord du Public, που θα ήταν λόγος για να αρνηθούν αναγνώριση αυτών των ε, εισερχομένων εγγράφων. Και πήραμε και επιπλέον εκθέσεις από συμβολιογράφους σε διάφορα κράτη-μέλη, που μετά από ένα αίτημα του Συμβουλίου Συμβολιογράφων συμφώνησαν να μας στείλουν δωρεάν συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Αυτή η πληροφόρηση από τους συμβολιογράφους μας ε, ανέφερε διάφορες δυσχέρειες. Τώρα η έκθεση. Από τα στοιχεία αυτά των εθνικών ε, εκθέσεων και από τις εκθέσεις των συμβολιογράφων ε, υποβάλαμε εκθέσεις αναχώρα για τα εξής θέματα. Πρώτον, τι είδος δημοσίων εγγράφων χρησιμοποιούνται εσωτερικά στο κράτος μέλος. Δεύτερον, τη φύση της αποδεκτικής ισχύω αυτών των δημοσίων εγγράφων στα 22 κράτη-μέλη που έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και τρίτον, οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τη δημόσια χρήση Τη εξαίρεση για λόγους δημοσίου συμφέροντος όταν εισέρχονται δημόσια έγγραφα πριν εισαχθεί αυτός ο κανονισμός στο δικό του νομικό σύστημα. Η έκθεσή μας ε, παρουσίασε τα αποτελέσματα μέσω ενός παραδείγματος, συγγνώμη, ενός παραρτήματος, όπως ακριβώς προβλέπει ο κανονισμός 1329 του 2014. Και κάναμε και συστάσεις για να βελτιωθούν ε, τα έγγραφα αυτά ε, όταν χρειαστεί να περάσουν σύνορα. Ποιε είναι οι συστάσει μας λοιπόν. Πρώτον, προτείνουμε το άρθρο 59 να μην ε, συγχαίεται με προηγούμενα εθνικά νομοθετήματα για δικαστικές αποφάσεις ή δημόσια έγγραφα. Τι σημαίνει αποδοχή. Η αποδοχή σημαίνει διαμεθοριακή μεταφορά ενός τέτοιου εγγράφου και τα αποτελέσματα μπορεί να αμφισβητηθούν εάν ε, ήταν δυνατόν να αμφισβητηθούν στο κράτος προέλευσης και στο κράτος ε, εισόδου. Δεύτερον, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί σωστή συμπλήρωση αυτού του εντύπου που υπάρχει στο παράρτημα 2. Διότι το έντυπο αυτό βοηθάει το κράτος μέλος υποδοχής για να ε, καταλάβουν περί τίνος πρόκειται. Τρίτον, οι συμβολιογράφοι θα πρέπει να ε, έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν, να, δηλαδή να συμπληρώσουν ένα τέτοιο έντυπο όπως έκαναν και προηγουμένως. Τέταρτο. Αυτό το έντυπο θα πρέπει να δίνει αρκετές λεπτομέρειες για την ε, αποδεικτική ισχύ για να μπορεί το κράτος μέλος ε, που το δέχεται να το δεχθεί. Και όπως είπαμε μπορεί να τυποποιηθούν ε, τα δεδομένα που χρειάζονται. Πέμπτον, η κατάργηση των εθνικών ε, προτέρων διαδικασιών του άρθρου 72 θα πρέπει να γίνει ευρύτερα γνωστή. Επίσης προτείνουμε ότι όταν αναθεωρηθεί ο κανονισμός αυτός θα ήταν σκόπιμο να εξετάσουμε δυνατότητα να δώσουμε τη δυνατότητα στις αρχές των άλλων κρατών μελών που λαμβάνουν ένα τέτοιο έγγραφο του άρθρου 59 να κάνουν μία από τις εξής πράξεις. Πρώτον, να απαιτήσουν να υπάρχει το έντυπο του παραρτήματος 2 εάν δεν έχει ε, Δεύτερον, να απαιτήσουν τις μεταφράσεις του δημοσίου εγγράφου και της, ε, του εντύπου αυτού. Και τρίτον, να ζητήσουν και να απαιτήσουν τη βοήθεια από σύμβολογράφους του κράτους προέλευσης. Μέχρι στιγμής καμία από τις δυνατότητες αυτή δεν υπάρχει εάν γίνει ένα αίτημα με βάση το άρθρο 59. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν μας ακούει ο κύριος καθηγητής, αλλά τον ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίαση και τώρα με χαρά θα καλωσορίσω τον κύριο Φρανσουά Τρεμόζα που είναι συμβολιογράφος στην Τουλούζη. Έχετε το λόγο παρακαλώ για 10 λεπτά κι εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μεγάλη μου χαρά που παίρνω το λόγο σήμερα ενώπιόν σας και θέλω να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος των 200.000 ε, ανθρώπων που εργάζονται ε, στα συμβολογράφη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο συμβολογράφος που εργάζεται στην Γαλλία είχα ήδη την ευκαιρία με από την έναρξη ισχύω του κανονισμού περί κληρονομικής διαδοχής να λάβω και να εφαρμόσω δημόσια έγγραφα που προέρχονται από τη Γερμανία, από το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Γερμανία χωρίς καμία δυσκολία δυσκολία και έχω εκδώσει και εγώ έγγραφα ε, με κατέθεση την Ισπανία και την, ε, το Βέλγιο που επίσης κυκλοφόρησαν χωρίς καμία δυσκολία. Τα έγγραφα λοιπόν σας διαβεβαιώ πως κυκλοφορούν πολύ ωραία μέσα στο πλαίσιο του κανονισμού περί κληρονομικής διαδοχής. Ο κανονισμός ε, αυτός θα πρέπει να πω και πρέπει να το πούμε εξ αρχή ότι αποτελεί μεγάλη πρόοδο που διευκολύνει τη ρύθμιση των διεθνών κληρονομικών διαδοχών. Είναι καλό παράδειγμα της πολιτικής των μικρών βημάτων που ήταν τόσο αγαπητή στους ιδρυτές πατέρες το... της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γιατί αυτό, διότι εν τέλει απλοποιεί την ε, ζωή των πολιτών μέσω του γεγονότος ότι το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού είναι εξαιρετικά ευρύ από την ε, έναρξη της διαδικασίας μέχρι την εκαθάριση, την ε, διαδοχή, όλη την τα θέματα δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και δημιουργεί ένα νέο μέσο που επιτρέπει να δίνεται και το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο αντικαθιστά 25 διαφορετικά συστήματα από ένα μόνο που ορίζει πλέον ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο, δηλαδή το κράτος της τελευταίας ε, ε, διαμονής, συνήθως διαμονής του θανόντος. Όλα αυτά πραγματικά λοιπόν απλοποιούν σε πολύ μεγάλο βαθμό την εργασία μας την καθημερινή Φυσικά είμαστε νομικοί, είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τα σημεία που μπορούμε να βελτιώσουμε, κάποιες δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν. Προφανώς εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες, αλλά και πάλι ήθελα να τονίσω αρχίζοντας το θετικό χαρακτήρα αυτού του κανονισμού. Οι δυσκολίες τώρα ποιε είναι. Η πρώτη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε στην πράξη είναι όταν καλούμεθα να εφαρμόσουμε το, το δίκαιο ενός άλλου κράτους από αυτό στο οποίο ε, εργαζόμαστε. Όταν είναι ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα καταφέρνουμε. Όταν όμως πρέπει να εφαρμόσουμε το δίκαιο του Μπουτάν ή του Καζακστάν, η πρόσβαση στην ενημέρωση και στις πληροφορίες είναι πολύ πιο δύσκολη και κάποιες φορές και αδύνατη. Και ωστόσο συμβαίνουν τέτοιες ε, υποθέσεις, ευτυχώς σπανίως. Σε σχέση με το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού, το πρώτο άρθρο ε, απαριθμεί ένα ολόκληρο κατάλογο εξαιρέσεων από το πεδίο εφαρμογή για συγκεκριμένα θέματα. Το πρώτο αποκλεί τα φορολογικά ζητήματα. Και το θυμίζω αυτό γιατί καθημερινά έχουμε πελάτες που έρχονται να μας δουν λέγοντας τέλεια χάρη στο κανονισμό αυτό μπορώ να ρυθμίσω, το, να αποφασίσω εγώ για το δίκαιο και άρα θα πληρώσω τα τους φόρους κληρονομιάς σε αυτή τη χώρα που θέλω εγώ. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Και σας διαβεβαιώ ότι αυτή, η ερώτηση ε, τίθεται πάρα πολύ συχνά και πολύ συχνά επανειλημμένα μέσα στο ίδιο ραντεβού. Οι άνθρωποι αυτό δεν το εμπεδώνουν. Δεν ξέρω γιατί. Μια εξαίρεση όπου εσείς άλλοι είναι το, τα, τα γαμήλια ε, καθεστώτα. Το πρώτο που καλούμεθα να κάνουμε πριν να προχωρήσουμε στην, στην εκαθάριση είναι το να εκαθαρίσουμε το χαμικό καθεστώς. Γιατί διαφορετικά μπορεί να, ε, ε, ε, να ε, γιατί μάλλον πάντοτε υπάρχει συνδυασμός των κανόνων ανάμεσα στα, στους νόμους που διέπουν την κληρονομική διαδοχή και αυτούς που διέπουν το γαμικά καθεστώτα. Δεν έχουν εναρμονιστεί πλήρως ε, οι νομοθεσίες, θα εναρμονιστούν ε, σε 15 μήνες και όλα θα γίνουν ωραία και καλά. Ναι, για διάφορα ζεύγη από την 1η Πρώτου 19, αλλά σήμερα μιλάμε για ε, περιπτώσεις διαδοχή ανθρώπων που έχουν παντρευτεί εδώ και κάποια χρόνια. Έχουμε ακόμα δηλαδή πολύ δρόμο μπροστά μας ε, που θα χρειαστεί να υποστούμε τις συνέπειες της έλλειψης εναρμόνισης είναι για ιστορικούς λόγους όσον αφορά τα γαμικά καθεστώτα. Έδωσα στη μελέτη μου ε, δύο παραδείγματα. Ένα παράδειγμα για την ε, ε, Γαλλία και την Καταλωνία, την Ισπανική Καταλωνία βεβαίως, και ε, όπου καλούμεθα να ρυθμίσουμε εδώ ένα θέμα διαδοχής ε, με ε, χωρισμό περιουσιακών στοιχείων ή με κοινοκτημοσύνη. Όμως δεν είναι το ίδιο, δεν ισχύει το ίδιο, γιατί αν ο Ισπανός συμβολογράφος ε, χειριστεί την υπόθεση θα πει ότι, ο, ότι τα αγαθα, περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στη Γαλλία ε, διέπονται από το καθεστώς διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων ενώ ο Γάλλος θα πει το αντίθετο, όχι ε, και τούμπαλιν. διότι θα θεωρήσει ότι το σύνολο των παρουσιακών στοιχείων εξαρτώνται από την ε, διαδοχή, από την κληρονομική διαδοχή. Ε, δεν υπάρχει λύση για το συγκεκριμένο πρόβλημα, ε, βράχει πρόθεσμα. Τώρα σε ορισμένα χρόνια όταν θα έχουμε εναρμονισμένα γαμικά καθεστώτα, αν αυτό θα λυθεί, δεν ξέρω πώς. Υπάρχει όμως πρόβλημα εδώ, ανάλογα δηλαδή με το ποιο συμβολογράφο σε ποια χώρα αναλαμβάνει την καθάριση. Το δεύτερο σημείο που θέλω να αναφέρω είναι το κριτήριο εγκύτητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό το κριτήριο δεν ε, δημιουργεί πρόβλημα. Όλοι ξέρουν που κατοικούσε ο Θανόν γιατί είχε εγκατασταθεί στις περισσότερες περιπτώσεις ε, για πολλά χρόνια ε, στο ίδιο σημείο στη συγκεκριμένη χώρα. Όμω, μιλάμε για παθολογικέ υποθέσει για ανθρώπου που ζουν ανάμεσα σε δύο χώρε. Πρόκειται συνήθω για ανθρώπου που ε, φτάνοντα ε, στη σύνταξη περνούν 8 μήνε στη Νότια Ευρώπη και 4 μήνε στη Βόρεια Ευρώπη, στη χώρα προέλευσή του. Ποια είναι η συνήθι κατοικία στη Νότια Ευρώπη, όπου περνάτε μεγάλο κομμάτι του χρόνου ή οι χώρε τη Βόρειας Ευρώπη όπου έχουν ε, τη πηγή του εισοδήματό του που κάνουν τη φορολογική του δήλωση ή όπου πηγαίνουν για να παρακολουθούνται από τον ε, γιατρό τους, όπου γιορτάζουν τις οικογενειακές γιορτές. Επίσης τίθεται η περίπτωση ανθρώπων που στη σύνταξη μεταβαίνουν σε άλλη χώρα για θέματα, για λόγους μάλλον οικονομικούς ή πρακτικούς. Κυρίως όταν ε, αυτός ο άνθρωπος έχει τοποθετηθεί σε κάποιο ηροκομείο άνευ της θέλησής του. Πρόκειται για κάποιον ευάλωτο άνθρωπο, ας πούμε ή κάποια άλλη, Αλτσχάιμερ ή κάποια άλλη, όποια και αν η παθολογία. Ακόμα και αν αυτός ο άνθρωπος ζει σε κάποιο χειροκομείο, σε μια χώρα άλλη, αυτός από μόνος του έχει επιλέξει την αλλαγή του κράτους διαμονής του. Αυτές οι δυσκολίες υπάρχουν. Αν απερίπτωση τα αντιμετωπίζουμε, δεν μπορεί να δοθεί μια οικουμενική απάντηση η νομολογία του δικαστηρίου μας βοηθά Ένα άλλο θέμα που τίθεται επίσης είναι να ξέρουμε αν η έννοια της συνήθους ε, κατοικίας προκύπτει με κοινό και αυτόνομο τρόπο από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Ορισμένες ε, καθεστώτα, μάλλον ε, ορισμένες νομοθεσίες ε, παίρνουν την συνήθη διαμονή ως κριτήριο εγκύτητας. Όμως αυτή ορίζεται διαφορετικά ανάλογα με το δίκαιο που χρησιμοποιείται. Ας πούμε, αν πάρουμε το παράδειγμα ενός στενόντος που ήταν παντρεμένος, μπορεί ας πούμε η συνήθις κατοικία να είναι στη χώρα Α, ενώ η κατοικία του ζεύγους να είναι στη χώρα Β. Υπάρχουν τέτοιες ε, περιπτώσεις. Αυτό που είναι βέβαιο ότι η έννοια αυτή θα πρέπει να εναρμοστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι τοπικές αρχές να μην έχουν υπερβολικά εθνικιστική ε, εικόνα του τι σημαίνει συνήθις κατοικία. Να συνειδητοποιήσουν ότι εφαρμόζουν ένα ευρωπαϊκό κείμενο και μία έννοια αυτόνομη ευρωπαϊκού δικαίου και να αφήσουν ε, τα μέρος τα όσα έμαθαν ως φοιτητές και σπούδασαν το ε, εσωτερικό εθνικό τους δίκαιο. Όλα αυτά που μας λέτε είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Απλά θέλω να σας πω ότι ήδη μιλήσατε για 10 λεπτά, οπότε θέλετε να κλείσετε την ομιλία σας. Για τα σύμφωνα διαδοχής ε, βλέπουμε πως στα διπανεπιστήμια αυτό το κομμάτι του κανονισμού δεν διδάσκεται επαρκώς. Ε, ε, οι καθηγητές δεν είναι ε, εξοικειωμένοι. Οι κανόνες θα πρέπει λοιπόν να μελετηθούν στη χώρα αποδοχής κάθε φορά. Σας ευχαριστώ και σε αυτό θα σταματήσω γιατί ξεπέρασα το χρόνο που μου είχατε δώσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Βλέπουμε ότι μιλάτε από πείρας και... Θα ακούσουμε τον παρακαθήμενό σας. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Ιζήτορο Αντώνιο Κάλβο Βιδάλ, που είναι συμβολογράφος στην Ισπανία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ε, καλέσατε, που με καλέσατε εδώ. Ο κανονισμός περί κλονικών διαδοχών είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα της οικοδόμησης Ευρώπης των πολιτών. Ε, λαμβάνει την έμπνευσή του στο σύνολό του από την έννοια της ενότητας. Δηλαδή έχουμε έναν διαθέτη, μία διαδοχή, έναν εφαρμοστέο νόμο, μία δικαιοδοσία, αρμόδια δικαιοδοσία, ένα έγγραφο που βεβαιώνει την ιδιότητα του κληρονόμου, του κληροδόχου, του διαχειριστή ή του εκτελεστή της διαθήκης και αυτό είναι το Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο. Ε, αυτή η έννοια της ενότητας σε ορισμένες περιπτώσεις ε, δεν εφαρμόζεται με απόλυτη αυστηρότητα εξαιτία του περίπλοκου των διασυνοριακών ε, κληρονομικών διαδοχών. Γι' αυτό λόγο γίνονται κάποιες εξαιρέσεις, για παράδειγμα σε θέματα αρμοδιότητας, για λόγους πρακτικούς και δικονομικούς. Απ' την άλλη μεριά, με την έννοια της βεβαίωσης της ιδιότητας του ε, κληρονόμου ε, για λόγους ε, ύπαρξης εσωτερικών αντίστοιχων εγγράφων στα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά το εφαρμοστέο νόμο γίνονται εξαιρέσεις για λόγους οικονομικούς, οικογενειακούς ή κοινωνικούς για συγκεκριμένα ίδια στοιχεία, περιουσιακών στοιχείων. Και θα εστιάσω ακριβώς στον εφαρμοστέο νόμο διότι η πρακτική εφαρμογή του κανονισμού ακριβώς σε αυτό το σημείο κατέδειξε πως υπάρχουν κάποιες αδυναμίες που πιστεύω, πιστεύω προσωπικά ότι θα έπρεπε να τις ε, αντιμετωπίσουμε μέσω μιας ε, διαφορετικής ερμηνείας. Ο κανονισμός έχει καθολικό χαρακτήρα. Δηλαδή όπως ακριβώς αναφέρει ο νόμος, ο, ο ίδιος νόμος εφαρμόζεται ε, όταν δεν είναι νόμος του κράτους, ενός κράτους μέλους, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα θα είναι η ίδια η αντιμετώπιση όλων των κρατών ε, μελών. Ε, η πρόταση της Κομισιόν ήταν να εξαιρεθεί η ε, αναπαραπομπή. Όμως τελικά στο άρθρο 34 συμπεριελήφθη κάτι που σημαίνει ότι η αρχική πρόταση Κομισιόν δεν υλοποιήθηκε. Πράγματι, το να λάβει κανείς υπόψη ε, το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο ενός κράτους που δεν είναι μέλος τρίτου κράτους όταν πρόκειται για μοντέλο που κάνει διαχωρισμό μεταξύ κινητών και ακίνητων πραγμάτων μπορεί να δημιουργήσει διαφορετική μεταχείριση ε, των ε, διαφόρων περιουσιακών στοιχείων. Να θυμάστε ότι τέτοιου είδους ε, μοντέλα ε, ε, προβλέπουν διαφορετική μεταχείριση για, τις κινητέ, για τα κινητά και διαφορετική για τα ακίνητα. Το οποίο σημαίνει ότι περιπλέκεται πολύ περισσότερο προβλε... η πρόβλεψη, η προβλεψιμότητα της εκτέλεσης μιας διαθήκης στο Ισπανικό δίκαιο, σε τέτοιες περιπτώσεις το Ανώτατο Δικαστήριο είχε την ε, τάση να ε, θεωρεί ότι ε, θα πρέπει να, εφαρμοστεί, να εφαρμοστούν οι αρχές ενότητας και της καθολικότητας και με αυτόν τον τρόπο απέριψε την επαναπαραπομπή, την αναπαραπομπή, συγγνώμη, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Στο μέτρο που Ζητώ συγγνώμη, αλλά μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα, λέει η Πρόεδρος. Στο μέτρο που ο κανονισμός ε, επιλέγει επίσης την αρχή της ενότητας και της ε, καθολικότητας του εφαρμοστέου νόμου, ε, θα ε, μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπιστεί το ζήτημα σε όλη την Ευρώπη, όπως το αντιμετώπισε η Ισπανία. Ο κανονισμός του άρθρου 13 παραδέχεται ότι σε ορισμένε περιπτώσεις ε, είναι δυνατό να γίνει ε, αναπαραπομπή και αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται μία ανασφάλεια βεβαιότητα σε ό,τι αφορά τους πολίτες που ε, θα είχαν ε, επιλέξει ε, το νόμο της συνήθους διαμονής τους ακόμα και αν αυτό είναι ένα κράτος το οποίο δεν ανοίξει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπ' αυτή την έννοια μια περιορισμένη εφαρμογή, μια περιοριστική εφαρμογή του 34.2 μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις που δεν είναι οι επιθυμητές. Σκεφτείτε την περίπτωση ενός Ισπανού πολίτη, ο οποίος πεθαίνει μετά τις 17 Αυγούστου 2015 χωρίς ε, διαθήκη και έχει συνήθη διαμονή στην Κούβα όπου βρίσκεται η οικογένειά του και το μεγαλύτερο τμήμα της περιουσίας του. Σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 1, ο νόμος της συνήθους διαμονής του τη μέρα ε, του θανάτου του θα πρέπει να εφαρμοστεί ε, για την ε, διαδοχή του. Δηλαδή ο νόμος της Κούβας. Επειδή όμως πρόκειται για τρίτο κρατός, όχι κρατός μέλος, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις διατάξεις του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου που ισχύουν στην Κούβα. Εκείνη την εποχή, σύμφωνα με το άρθρο 15 του αστικού κώδικα της ε, Κούβας, ε, η διαδοχή του, ε, η κληρονομική διαδοχή του διέπεται από το κράτος το οποίο, του οποίου είναι υπήκος ο Θανών. ανεξαρτήτως το, της θέσης των αγαθών τα οποία κληροδοτούνται. Το οποίο σημαίνει δηλαδή θα πρέπει, ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί μέσω της αναπαραπομπής ο ισπανικός, το ισπανικό δίκαιο. Επίσης, ας ε, δεχτούμε τώρα μια, ένα άλλο σενάριο με τις ίδιες ακριβώς ε, παραμέτρους ε, όπου ο, η συνήθις διαμονή του θανόντος δεν είναι η Κούβα διότι έχει μόλις μετακινηθεί εκεί, μόλις μετακομίσει. Σε αυτή, την περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2, Και δεδομένου ότι τη στιγμή του θανάτου του ο Θανόν είχε ένα πολύ πιο στενό δεσμό με ένα άλλο κράτος, όχι την ε, Κούβα, η εφα... το νόμο του εφαρμοστή θα είναι αυτός του άλλου κράτους. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο νόμος της Κούβας. Δεδομένου ότι με την Κούβα είχε τον πιο στενό δεσμό, παρόλο που δεν ήταν η συνήθις κατοικία του. Βλέπετε λοιπόν ότι... Ε, ε, ε, σε αυτή την περίπτωση δεν θα ε, γίνει αναπαραπομπή. Στην πρώτη, στο πρώτο από τα δύο σενάρια, τα δύο παραδείγματα, ε, όλες οι συνθήκες ε, δείχναν το στενοδεσμό με την Κούβα, αλλά δεδομένου ότι μπήκε σε εφαρμογή ο μηχανισμός της αναπαραπομπής, δεν εφαρμόστηκε, δεν θα εφαρμοζόταν το δίκαιο της Κούβας. Ε, αυτό λοιπόν δείχνει ότι δεν γίνεται σωστή ερμηνεία του άρθρου 34 παράθος 2 Κατά την άποψή μου, μια σωστή ερμηνεία του 34.2 θα έπρεπε να περιλαμβάνει το εξή. Όταν το, ο νόμος του κράτους, στο οποίο ο Θανόν είχε την τελευταία συνήθη διαμονή του τη στιγμή του θανάτου του, είναι επίσης ο νόμος του κράτους με το οποίο έχει το πιο στενό δεσμό, τότε δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται ο μηχανισμός της αναπαραπομπής ε, σύμφωνα με την εξαίρεση που προβλέπει το άρθρο 34 παράγραφος 2. Με διαφορετικό τρόπο όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε το, την ε, ρήτρα δημοσίου συμφέροντος του άρθρου 35 ε, δημοσίας τάξης, συγγνώμη, του άρθρου 35. Σε, ορισμένες, ε, σε ορισμένα καθεστώτα αν ο Θανόν έχει παιδιά, ε, ο, το παιδί του παίρνει διπλάσια, ε, διπλά τη της, ε, κληρονομιάς από ότι η κόρη. σε άλλες περιπτώσεις γίνονται διακρίσεις σύμφωνα με, το, με τη θρησκεία ή το δόγμα. Σε δεδομένου ότι υπάρχουν τέτοιου είδους ε, διατάξεις, η προάσπιση των αρχών και των αξιών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, μεταξύ αυτών ε, η αποφυγή οποιασδήποτε διάκρισης για λόγους φίλου ή πιστής, επιβάλλει την, τον αποκλεισμό της εφαρμογής του άρθρου του, το, το, του κανονισμού. Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να μην εφαρμοστούν οι διατάξεις τελευταίας βούλησης αν είναι αποτέλεσμα μιας ε, ε της ε, ε, μεταγραφής τέτοιων νόμων σε μια διαθήκη. πρέπει ιδιαίτερος να λάβουμε υπόψη αυτή την διάταξη σε ό,τι αφορά ε, την έκδοση του Ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου. Αντίθετα με τις αποφάσεις ε, δικαστηρίων ή τα δημόσια έγγραφα, η έκδοση του Ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου έχει, γίνεται για να χρησιμοποιηθεί σε ένα κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό της έκδοσης όπου θα έχει την ισχύ, την πλήρη ισχύ σύμφωνα με το 69.1 χωρίς να υπάρχει ανάγκη για οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη διαδικασία. Αυτό το αναφέρει, ε, όπως για παράδειγμα αυτές του κανονισμού ε, περί δικαστικών αποφάσεων, ε, που σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος α ε, προβλέπονται συγκεκριμένες ε, διαδικασίες και μία εφαρμογή αυτής της απόφασης αν αυτή έρχεται σε καταφανή αντίθεση με το, με το δημόσια τάξη του κράτους αυτού. Η εξωχώρια ιδιότητα, φύση μάλλον του Ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου, αποδεικνύει ότι ε, η αρχή που το εκδίδουσα αρχή θα πρέπει να αξιολογεί πολύ προσεκτικά τι συνέπειε που μπορεί να έχει αυτό όταν εκτελεστεί σε άλλο κράτο ε, μέλος. μέλο. Αν δεν το κάνει αυτό η εκδίδουσα αρχή, κανένα δεν θα μπορέσει να το κάνει κατά την εφαρμογή του άρθρου 69.1 στο κράτο μέλο στον οποίο εκτελείται. Μπορείτε παρακαλώ να κλείσετε την ε, ομιλία σα με τα συμπεράσματά σα, Ζητώ συγγνώμη που πιέζω. Ο στόχος αυτού του μέτρου δεν είναι άλλος παρά να ενισχύσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και να βελτιώσει την ε, νομική ασφάλεια προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση του κρυονομητηρίου. Ιδιαίτερο διότι μέσω αυτού, όπως αναφέρει το άρθρο 69 παράγραφος 5, για να διευκολυνθεί ο ρόλος των πρωταγωνιστών μιας διασυνοριακής ε, διαδοχής τίθεται στη διάθεσή τους μέσω του ε, κληρονομητηρίου, ένας ε, τρόπος για την ε, πρόσβαση στα εσωτερικά συστήματα εγγραφής σε μητρό. Ευχαριστώ. maybe I can... Ευχαριστώ. Μήπως η Επιτροπή Μήπως η κυρία Βιλαμπαντιά θέλει να μας πει τίποτα. Όχι. Α, εσείς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Τρία σύντομα μη τεχνικά θέματα. Πρώτον, να αναφερθώ στον ε, οδηγό για την κλονική διαδρομή για πολίτε πολίτες που ανέφερε ο κ. Τρεμόζα. Τον προετοιμάσαμε μαζί με τα κράτη-μέλη και τους Ευρωπαίους συμβολιογράφου για να εξηγήσουμε στου πολίτες τα ωφέλη από τον νέο κανονισμό όπως ακριβώς τα ανέφεραν και οι προηγούμενοι ομιλητές, τώρα είναι ε, υπομετάφραση και ελπίζουμε να δημοσιευθεί από την υπηρεσία δημοσιεύσεων σύντομα και κατόπιν θα ξεκινήσουμε μέσω των ε, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μια εκστρατεία για να ενημερώσουμε για την ύπαρξη αυτού του οδηγού. Ήδη Κάνουμε μια εκστρατεία για τον κανονισμό όταν τέθηκε σε ισχύ το καλοκαίρι του 2015. Και ήταν πολύ επιτυχημένη αυτή η εκστρατεία. Ελπίζουμε λοιπόν και ο οδηγός αυτός να ε, έχει ευρεία απήχηση στους πολίτες. Επίσης με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο όπου συμμετέχουν επαγγελματίες του τομέα των νομικών επαγγελμάτων ε, για να συζητήσουν για αστικά και εμπορικά θέματα. Δημιουργήσαμε μια ομάδα εργασίας όπου συμμετέχουν και οι συμβολιογράφοι, η Επιτροπή, τα κράτη-μέλη και πάλι λοιπόν οι συμβολιογράφοι για να προκύψουν και κάποια τεχνικά δελτία για να ενημερώσουμε τους πολίτες για το τι έγραφα απαιτούνται για να καταγραφούν σε Μητρώα ε, τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ε, ε γίνει αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής για να ξέρουν ε, πώς ακριβώς θα αντιμετωπιστούν τέτοια θέματα σε κάθε κράτος μέλος. Όλα αυτά για να βοηθήσουμε την καθημερινή εφαρμογή του κανονισμού αυτού από τους επαγγελματίες του κλάδου και από τους πολίτες. Επίσης, η Επιτροπή παρήγγειλε μια μελέτη που ολοκληρώθηκε φέτος και θα δημοσιευθεί στο ίντερνετ στη δικτυακή μας πύλη σύντομα για το τι κάνουν ή προτίθεται να κάνουν τα κράτη-μέλη για την ηλεκτρονική καταγραφή του Ευρωπαϊκού Κληρονομητηρίου το λεγόμενο ECS που είναι ένα σημαντικό στοιχείο του κανονισμού ο στόχος του είναι να επιτρέψει στους κληρονόμους να αποδείξουν σε ένα άλλο κράτος μέλος ότι είναι νόμιμοι κληρονόμοι ενός περιουσιακού στοιχείου που ε, είναι σε άλλο κράτος μέλος. Και θα ήταν χρήσιμο και για τους επαγγελματίες να ξέρουν αν κάποιος σε κάποιο άλλο κράτος μέλος έχει ήδη εκδώσει ένα τέτοιο κληρονομητήριο για να μην υπάρχουν συγκρουόμενα τέτοια ECS Κάναμε μια μελέτη προκατακτική για να δούμε τι κάνουν τα κράτη-μέλη, αν ήδη καταγράφουν τα κληρονομητήρια και περίπου τα μισά κράτη-μέλη καταγράφουν ηλεκτρονικά αυτά τα ECS. Το θέμα είναι εάν θα είχε έννοια η Ένωση να προτείνει υποχρεωτική νομοθεσία για να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να καταγράφουν τα κληρονομητήρια που εκδίδουν και αν θα ήταν χρήσιμο τα κράτη-μέλη να διασυνδέουν τα μητρώα τους ε, κλινομητηρίων. Και βεβαίως όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι αναφανδόν υπέρ αυτής της ιδέας, αλλά πρέπει να δούμε πόσο συχνά προκύπτουν τέτοια συγκρουόμενα ίσιας. E Γιατί φυσικά θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί κανόνες δικαιοδοσίας όταν εκδίδεται ένα ECS. Και τέλος, αν δεν το προσέξατε, τον περασμένο μήνα το δικαστήριο εξέδωσε την πρώτη απόφαση στα πλαίσια εφαρμογής του κανονισμού. Άλλες δύο υποθέσεις ε, είναι σε εξέλιξη. Η ακροματική διαδικασία έγινε για τη μία χτες και για την άλλη θα γίνει σε λίγες μέρες. Θα είναι λοιπόν σημαντικές αυτές οι αποφάσεις. Και η πρώτη ήδη είναι σημαντική γιατί λέει ότι εάν κάποιος ε, κληρονόμος που εφήγει από κάποια διαδικασία σε άλλο κράτος μέλος θα πρέπει να ε, ωφεληθεί από το ότι σε κάθε κράτος μέλος ε, θα πρέπει να γίνεται ε, σεβαστή η διαδικασία που έχει εφαρμοστεί από άλλο. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, είναι πολύ τεχνικές. Ήθελα απλώς όμως να υπογραμμίσω ότι ήδη έχουμε την πρώτη απόφαση του δικαστηρίου για την εφαρμογή του κανονισμού αυτού. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους αν υπάρχουν ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σε αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες ε, παρουσιάσεις. Δεν βλέπω. Ωραία. Εντάξει, έτσι θα τηρήσουμε και το χρονοδιάγραμμα εργασιών μας. Α, η Ζωέλ. Θέλω να συγχαρώ τους ομιλητές μας γιατί ξέρω πόσο τεχνικά είναι τα θέματα αυτά, γιατί και εγώ έχω ασχοληθεί. Γιατί βεβαίως είναι εύκολο να λες ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται ο κανόνας της συνήθους κατοικίας. Αλλά ποιος είναι ο κανόνας που καθορίζει την ε, ε, βούληση. Και ε, εγώ είμαι από τη Βρετάνη όπου ζουν πολύ ηλικιωμένοι Άγγλοι. Στην Αγγλία είναι πολύ σημαντικό τι καθορίζει η Διαθήκη. Ενώ στη Γαλλία υπάρχει πάντα η νόμιμη μοίρα. Ε, των απογόνων. Άρα έχει σημασία ε, σε ποιο νόμο υπάγεται κανείς. Και ε, τελικά ασκείται το δίκαιο του τόπου κατοικίας και έτσι όλοι αυτοί οι Άγγλοι θα θέλανε να δώσουν στην κυρία με την οποία ζουν την περιουσία τους, την παίρνουν τα παιδιά τους. Θα προκύψουν λοιπόν Συγκρούσει που δεν θα μπορεί να επιλύσει ένα δημοσιογράφος, ε, ένας σύμβολιογράφος. Γιατί η κυρία που ζει με έναν Άγγλο στη Γαλλία και νομίζει ότι θα μπορέσει να μείνει στο σπίτι δεν μπορεί γιατί τα παιδιά που ίσω είναι από την Αγγλία θα κληρονομήσουν το σπίτι το οποίο θα πουληθεί κτλ. Ήταν ε, περίπλοκα όσα μα εξήγησε ο, ο από τη Γαλλία αλλά είναι η καθημερινή πραγματικότητα για τους συμβολογράφους. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Μα συμφωνώ απόλυτα. Ξέρω τι δράματα ζουν και την έλλειψη ενημέρωση που έχουν οι πολίτε. Ο Ταντέο Εύκα. Θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, επί του θέματος αυτού. Θεωρώ ότι ένας οδηγός, ένα εγχειρίδιο για τους κληρονόμους είναι απόλυτα αναγκαίος. Αλλά εφιστώ την προσοχή σας επί της ανάγκης κατάρτισης των ε, δικαστών για την ομολογία των δικαστηρίων. Ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους κανόνες, οι αποφάσεις των δικαστηρίων. Μου ετέθη πρόσφατα το εξή ερώτημα από έναν Πολωνό πολίτη που έχει διπλή υπηκότητα. Πολωνική και γαλλική. Όχι, συγγνώμη, γερμανική και ζει στη Γερμανία. Γιατί τέθηκε ένα θέμα κληρονομική διαδοχής για κάποιου απογόνους. Και τη στιγμή που η απόφαση του δικαστηρίου απεστάλλει, έμαθαν ότι χρειαζόταν κάποιο άλλο πιστοποιητικό, που να λέει ότι αυτή η απόφαση είναι σύνομη με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Βεβαίω, το Γερμανικό Δικαστήριο του έστειλε αυτό το πιστοποιητικό, αλλά χρειάστηκε να πληρώσουν και πάλι 280 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, για να λάβουν ε, αυτό το επιπλέον ε, πιστοποιητικό. Όλοι λοιπόν πρέπει να έχουν περισσότερη προφόρηση και οι κληρονόμοι αλλά και οι επαγγελματίες του κλάδου. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Αν δεν υπάρχουν ε, άλλες ερωτήσεις, να ευχαριστήσω και εγώ τους προσκεκλημένους μας για τις ε, εξαίρετες παρουσιάσεις και ολοκληρώνουμε για το θέμα αυτό και να πούμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη πληροφόρηση και θα παρακολουθήσουμε το θέμα, θα δούμε τι αποφάσεις θα προκύψουν από το δικαστήριο και τώρα να δώσω την προεδρία στον πρόεδρό μας ο οποίος ε, μετριοφρόνος κάθε στην τελευταία σειρά. Yes, dear colleagues, Αγαπητοί συνάδελφοι, 31 τώρα. Και βεβαίως η κυρία Ντελβό έχει πολλά να μας πει ακόμη για να εξετάσουμε και το σχέδιο έκθεσης που έχει εκπονήσει για τις τήσεις εκθέσεις 15 και 16 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Κυρία μου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχουμε την ετήσια έκθεση που δεν είναι ετήσια αλλά είναι διετής έκθεση για τη φορά της χρονιά 2015 και 2016 για τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που είναι θεμελιώδεις για τη λειτουργία της Ένωσης αλλά δεν είναι και οι μόνες αρχές που εξυπηρετούν την ε, ορθή λειτουργία της Ένωσης και δεν πρέπει να τις θεωρήσουμε ως εμπόδια στην αποτελεσματικότητά της. Αφού διάβασα τη συνέκθεση της ε, Κομισιόν, τα συμπεράσματα της ΚΟΖΑΚ, ε, τη δουλειά της Επιτροπής των Περιφερειών και τι γνωμοδοτήσει των Εθνικών Κοινοβουλίων, φαίνεται πως όλα τα μέρη καταβάλουν μια αυξανόμενη προσπάθεια ώστε να τηρήσουν τις αρχές, να τηρούν τι τις αρχές της και της αναλογικότητας. Από το 2014 τα Εθνικά Κοινοβούλια έδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή πολιτική μέσω των νέων μέσων εργαλείων που δημιουργήθηκαν μέσω του REFIT και η Κομισιόν συνέχισε να εφαρμόζει το ενισχυμένο σύστημα βελτίωσης της νομοθεσίας και Βλέπουμε πως ε, γίνονται αισθητές οι επιρροές αυτής της δέσμευσης. Ας πούμε είχαμε 65 γνωμοδοτήσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων, μεγάλη αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος και η μη συμμόρφωση των μελετών ε, αντικτύπου της Κομισιόν έχει μειωθεί, πράγμα που ακόμα καλύτερα δηλαδή. Έχουμε μια έκθεση εξέτασης, μια, μια επιτροπή εξέτασης ε, των υποθέσεων που έχουν μειωθεί στο 23% και το υπόλοιπο πάντοτε ξαναδουλεύει τις μελέτες σύμφωνα με τα σχόλια που λαμβάνει από αυτή την Επιτροπή. Ενθαρρύνουμε λοιπόν τους πρωταγωνιστές να συνεχίσουν σε αυτό το δρόμο ακριβώς έτσι ώστε να εξασφαλιστεί και να ενισχυθεί η απόδοση και η αποτελεσματικότητα της Ένωσης. Ενθαρρύνουμε στη χρήση των υφιστάμενων ε, εργαλείων που έχουν δημιουργηθεί από το 2015, δηλαδή πρόσβαση στις μελέτες αντικτύπου και στους οδικούς χάρτες μέσω του, ε, και των, των, της εργαλειοθήκης. Επίσης οργανώνονται μελέτες και ενημερώσεις του, και τακτικές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Κομισιόν. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα site που λέγεται «Βοηθήστε μας να μειώσουμε τις διατυπώσεις, δώστε μας τη γνώμη σας» και το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να γνωμοδοτήσει κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας και αυτά όλα υπάρχουν στη βάση δεδομένων Connect και όλες οι πληροφορίες ε, που προέρχονται από τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα Rectex. Πρέπει να ενθαρρύνουμε λοιπόν τις ανταλλαγές ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια και πιστεύω ότι μπορεί να δημιουργούμε ένα σωρό εργαλεία για να ενισχυθούν οι αρχές της επικουρικότητα και της αναλογικότητας και να αυξάνεται η συμμετοχή, όμω πρέπει αυτά τα εργαλεία να χρησιμοποιούνται κιόλα. Δεν νομίζω λοιπόν πως πρέπει να προσθεθούν κι άλλα μέσα, γιατί αυτό δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να αυξάνει την περίπλοκο χαρακτήρα του συστήματος, ενώ εμεί επιθυμούμε το αντίθετο, την απλοποίηση. Την περασμένη μόλις εβδομάδα ο πρόεδρος της Επιτροπής άρχισε τη, ε, ε, δημιούργησε μάλλον Task Force ε, μας, η οποία ξεκίνησε επισήμω για την επικουρικότητα και την αλλαλογικότητα. Σύμφωνα με τον κανονισμό του Κοινοβουλίου, η δική μας Επιτροπή είναι αρμόδια επί της ουσίας. Πιστεύω πως η Επιτροπή μας λοιπόν θα εκπροσωπηθεί σε αυτή τη Task Force με τρία μέλη. Αυτά και να πω ότι είμαι βεβαίως έτοιμη να συνεργαστώ με τους σκιώδεις ώστε να βελτιώσουμε την έκθεση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό το project γύρω από την πρόταση του κυρίου Γιούγκερ τώρα η μορφή. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο τι ακριβώς θα είναι. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο. Ο κύριος κάρίμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας τη Μαρή για την προετοιμασία του σχεδίου έκθεσής της. Βεβαίως, Στη διάρκεια των ετών είχαμε ευκαιρίες να ανταλλάξουμε απόψεις για αυτά και άλλα θέματα επανελειμμένως. Αλλά θα ήθελα να της προσφέρω τη δική μου υποστήριξη στη δουλειά που κάνει και στον τρόπο που, με τον ίδιο τρόπο που ανέκαθεν με υποστήριζε σε αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα. Όσον αφορά την Επιτροπή, Πρόεδρε, με ενδιαφέρον άκουσα την αποσαφήνιση που εσείς μόλις μας δώσατε, γιατί εγώ είχα την εντύπωση ότι ο πρόεδρος Γιούνκερ είχε δώσει σαφώς όθηση και ότι αυτή θα είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθεί, Αν όχι θα το ξαναδούμε σε εν καιρό, αλλά πιστεύω πως αυτή είναι η κατεύθυνση όντως που προτείνει η Κομισιόν, ίσως κάπως θα μας αποσαφηνίσουν. Όχι η μορφή συμμετοχής του Κοινοβουλίου δεν είναι ακόμα απόλυτα σαφής, λέει ο Πρόεδρος. Μάλιστα, ευχαριστώ. Οπότε, Πρόεδρε, δεν ξέρω αν η Μαρή θέλει να στηρίξει αυτή την ιδέα ή όχι, αλλά ίσως να ήταν καλό να κάνουμε μια σχετική ακρόαση εδώ, σε κάποια φάση, για να εξετάσουμε αυτές τις ιδέες πιο εις βάθος. Το ρίχνω ιδέα. Το σχέδιο έκθεσης Μάντι νομίζω θα μπορούσαμε επίσης να το βελτιώσουμε αναφερόμενοι στην αναλογικότητα που συχνά την ξεχνάμε και όπως τόνισα και σε προηγούμενες μου εκθέσεις στο παρελθόν πιστεύω πως η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσο η νομοθεσία είναι αναλογικά ισορροπημένη σε σχέση με τα κείμενα που παράγει. Και ο έλεγχος της αναλογικότητας θα πρέπει να γίνεται κάθε φορά και να απορρίπτονται οι προτάσεις με δυσανάλογο φόρτο επί της ανταγωνιστικότητας και μικρομεσαίων. Αντίκτυπο και, ε, αντίκτυπος και το κόστος για τις περιφέρειες επίσης θα πρέπει να μετρηθεί. Η αξιολόγηση λοιπόν της αναλογικότητας είναι πολύ σημαντική για να παραμένουν ανταγωνιστικές εταιρείες και η Task Force που ερευνά, μα εξετάζει μάλλον διεθνείς νομοθεσίες και την ανταγωνιστικότητα των εταιριών και θα πρέπει να αποτελεί τμήμα κλειδί όλων αυτών. Σε προηγούμενες εκθέσεις μου είχα ζητήσει παράταση της προθεσμίας των 8 εβδομάδων για τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτό δεν εμφανίζεται εδώ, αλλά ξέρω ότι έχουμε κάνει παλιότερα συζητήσεις επ' αυτό. Υπάρχουν, ας πούμε, περιπτώσεις όπου φυσικές καταστροφές μπορεί να συμβούν που να εμποδίσουν τα Εθνικά Κοινοβούλια από το να, συνε... να... να τηρήσουν αυτή την προθεσμία των 8 εβδομάδων. Θα μιλήσω με τη Μάντη, να δούμε αν υπάρχει χώρος ε, περιθώριο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 Επίσης θα ήθελα να δω πιο λεπτομερείς επεξηγηματικές δηλώσεις από την Κομισιόν εκεί όπου έχουμε ανάλυση με βάση στοιχεία για τις προτάσεις της. Η εμπειρία δείχνει ότι όταν ένας, μια μελέτη που δεν είναι αρκετά προσεκτική και εξονυχιστική και δεν αναλύει ε, κάθε επιλογή ε, εις βάθος θα υπάρξουν προβλήματα για την υιοθέτηση της νομοθεσίας συχνά και μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στην απόσυρση αυτής της νομοθεσίας. Γι' αυτό είναι καλύτερο να κάνουμε μια πολύ καλή ε, διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς όσο γίνεται νωρίτερα, ώστε να αποφύγουμε προβλήματα αργότερα. Ε, επίσης, με χαροποιεί που η Κομισιόν δεσμεύεται στο να κάνει περισσότερες διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους πολίτες, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτό θα γίνει όσο γίνεται νωρίτερα. Κάποιες φορές ε, υπάρχουν μη επιθυμητές και όχι σκόπιμες επιπτώσεις που πρέπει να προσέξει η Κομισιόν ώστε να λάβει αποφάσεις όντας πιο ενήμερη για οποιαδήποτε πολιτική επιλογή. Και ε, ακόμη θα ήθελα να επαναλάβω την πρόταση από την προηγούμενη μου έκθεση που υιοθετήθηκε εδώ στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια και ζητούσε την αξιολόγηση ε, αντικτύπου για, στην επικουρικότητα και στην αναλογικότητα μετά από το τριμερή διάλογο. Να δούμε δηλαδή κατά πόσο μια πρόταση που έχει ουσιαστικά τροποποιηθεί εξακολουθεί να ισχύει σε θέματα επικουρικότητας και αναλογικότητας. Ε, προσβλέπω λοιπόν συνεργασία μου με τη ΜΑΤ και με τη Μαριών για αυτό το τόσο σημαντικό φάκελο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, Καταρχήν να ευχαριστήσω την κυρία Ντελβό για την πολύ καλή αυτή έκθεση που σχολιάζει την ετήσια έκθεση Κομισιόν για την επικορικότητα και την αναλογικότητα για τα, το 2015 και το 2016. Όπως είπα και σε προηγούμενες συζητήσεις, είναι πολύ σημαντικό να διαθέτουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία εκεί που η Ευρώπη μπορεί να σημειώσει πρόοδο και εκεί που μια τέτοια νομοθεσία θα έχει προσθέμενη αξία. Ε, η αλήθεια βέβαια είναι ότι η ε, ακατάλληλη χρήση της επικορικότητας και της αναλογικότητας ε, δίνει τροφή στους ευρωσκεπτικιστές και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέλος Οκτωβρίου δημοσίευσε την πρωτοβουλία καλύτερες λύσεις για καλύτερα αποτελέσματα ε, και σε αυτή την έκθεση η Κομισιόν παρουσιάζει τις προστάσεις της ε, για να βελτιώσει την διαφάνεια, την νομιμοποίηση ε, και την λογοδοσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις διαβουλεύσεις, δημόσιες διαβουλεύσεις και την δυνατότητα των εμπλεκομένων και ενδιαφερμένων μερών να επηρεάσουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Μέχρι την, ε, το 2017 που θα δημιουργηθεί το... Ε, μάλλον όταν το 2017 ενεργοποιηθεί το site στο ίντερνετ που θα επιτρέπει στους ε, ενδιαφερόμενους να παίρνουν μέρος και η καλύτερη χρήση της επικουρικότητας και της αναλογικότητας θα βοηθήσει στην λήψη των πιο κατάλληλων αποφάσεων για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που, αντιμετωπι... που ε, αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Task Force που σύστησε την περασμένη εβδομάδα. Task Force για την επικορικότητα και την αναλογικότητα. Περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, η Task Force θα αρχίσει να λειτουργεί στις αρχές του επόμενου έτους, δηλαδή σε ένα μήνα περίπου. Δεν πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα έχει αρκετό χρόνο για την πρόσληψη προσωπικού και πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτή η Task Force. Thank you very much. Πρόεδρος κ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξεκινώ ευχαριστώντας την κυρία Ντελβό για την έκθεσή της. Όπως πάντα θα εργαστώ πρόθυμα μαζί της. Σε ό,τι φορά την διαδικασία ελέγχου της επικουρικότητας, διαδικασία της κίτρινης κάρτας όπως ονομάζεται πολύ συχνά, δεν έχω πιστεί, επουδενή, επουδενή λέω, ότι τα εθνικά κοινοβούλια παίρνουν σοβαρά, στα σοβαρά αυτή τη διαδικασία. Μου έχει δημιουργηθεί εντύπωση ότι ορισμένα εθνικά κοινοβούλια δεν θεωρούν ότι αξίζει η δουλειά που πρέπει να κάνουν για να συμμετάσχουν αξίζει την προσπάθεια. Γιατί έχουμε δώσει στα εθνικά κοινοβούλια αρκετά κίνητρα έτσι ώστε να συμμετάσχουν ή όχι. Αν θέλουμε τα εθνικά κοινοβούλια να πάρουν στα σοβαρά αυτή τη διαδικασία, πρέπει και εμείς οι ίδιοι να παίρνουμε στα σοβαρά τη συνεισφορά τους. Και δεδομένου ότι το κατόφλι το οποίο προβλέπει η συνθήκη είναι πολύ ψηλό, δεν εκπλήσει που ορισμένα κοινοβούλια δεν έχουν ως προτεραιότητα την ε, υλοποίηση της ε, διαδικασίας ελέγχου της επικουρικότητας. Αυτό πρέπει να το εξετάσουμε. Προφανώς δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη συνθήκη εδώ και τώρα. Θα ήταν άλλωστε μια πολύ κακή ιδέα να ξεκινήσει μια τέτοιου είδους διαδικασία να αναθεώρηση συνθήκη. Αλλά να εξετάσουμε πώς μπορούμε να κινητοποιήσουμε τα εθνικά κοινοβούλια έτσι ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία της Κίτρινης Κάρτας για να βελτιωθεί η νομοθεσία και να αποφύγουμε περίπλοκες και ε, έντονες ε, συζητήσεις πώς βελτιώντας τις ίδιες νομοθετικές προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λέει ο πρόεδρος Κομισιόν. Θα ήθελα να λάβει το λόγο. Αλλά επειδή έχουμε καθυστερήσει παρακαλώ πολύ με λίγα λόγια. Η Επιτροπή. Μια σύντομη απάντηση για το θέμα της Task Force. Η Κομισιόν ελπίζει ότι τα όργανα τα οποία, από τα οποία ζητήθηκε να ορίσουν μέλη θα το κάνουν πριν το τέλος του χρόνου. Η ίδια η Task Force κατά τα άλλα θα καθορίσει τους διαδικαστικούς κανόνες με βάση τους οποίους θα λειτουργεί. Αυτά μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ε, δεν ξέρω αν ικανοποιήθηκε απόλυτα ο κύριος Ράνιεφ, αλλά εντάξει. Λοιπόν, προθεσμία για τροπολογίες 8 Δεκεμβρίου. 5 ώρα το απόγευμα. Η κυρία Ντελβό δεν θέλει να μας πει τίποτα. Επόμενο θέμα. 32. εξέταση ενός σχεδίου εκθέσεως για την προσαρμογή μιας σειράς απονομικών ε, ενεργειών στον τομέα της δικαιοσύνης. Ο εισηγητής μας είναι ο κύριος Σάγερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο θέματα μας απασχολούν, αλλά μπορούμε να τα συζητήσουμε από κοινού γιατί συνδέονται. Από ό,τι κατάλαβα πρέπει να είμαι πολύ σύντομος γιατί έχουμε καθυστερήσει. Επειδή είναι πολύ περίπλοκο το θέμα αυτό, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, που εργάζονται, γιατί δεν είναι και τόσο συναρπαστικό, αλλά θέλει πολύ και σκληρή δουλειά. Εγώ εργάζομαι για το θέμα της επιτροπολογίας εδώ και 10 χρόνια και το Κοινοβούλιο ασχολείται με αυτό τουλάχιστον 20 και έχω ασχοληθεί με τα σημαντικότερα θέματα γι' αυτό πριν από 10 χρόνια, αν ρωτούσα αρκετούς συναδέλφους για το τι είναι οι εφαρμοστικές και, τα, και κατεξοδότηση πράξεις, πολλοί μπορεί να μην ήξεραν. Αλλά τώρα, συζητώντας διάφορες επιτροπές που συνέβαλαν σε αυτή την έκθεση, μπορώ να σας πω με μεγάλη περηφάνεια ότι τώρα τα ξέρουν πολύ καλά. Και ο λόγος είναι ότι το Κοινοβούλιο δεν είχε τέτοιες δυνατότητες ε, παλιότερα αλλά στις περισσότερες εθνικές νομοθεσίες ακόμη και αν δεν υπάρχει μία ε, δυνατότητα ελέγχου των κατεξοδότησης ενεργειών οι κυβερνήσεις εξαρτώνται από τα κοινοβούλια που μπορούν φυσικά να τις αμφισβητήσουν ανα πάσα στιγμή. Αλλά εδώ ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχουμε αυτού του είδους ε, την ισχύ αλλά επειδή έχουμε αντιμετωπίσει ήδη ε, πολλά θέματα ε, με πολλές λεπτομέρειες που δεν τα συζητούν συνήθως τα Εθνικά Κοινοβούλια και επειδή θέλουμε να έχουμε το πάνω χέρι στην εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας και τώρα μετά τη Λισαβόνα έχουμε να το κάνουμε γι' αυτό λοιπόν τώρα πλέον έχουν γίνει από το 2013 τρεις προτάσεις omnibus για να εναρμονιστεί η υπάρχουσα νομοθεσία με το νέο νομοθετικό ε, κανονιστικό πλαίσιο και με τη συνθήκη της Λισαβόνας και οι τρεις προτάσεις αυτές απέτυχαν λόγω της αντίστασης του Συμβουλίου και τώρα έχουμε άλλα δύο νομοθετήματα. Ένα για τον τομέα της δικαιοσύνη και έναν για διάφορους τομείς με τον ίδιο στόχο δεν είναι το πιο δύσκολο τμήμα της προσπάθειας αυτής. Το πιο δύσκολο θα είναι τώρα δηλαδή, δεν είναι η πιο δύσκολη φάση της διαδικασίας. Η πιο δύσκολη θα είναι όταν ε, περάσουμε στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ την Επιτροπή για αυτή την πρόταση. Θεωρώ ότι τώρα που έχουμε τη Διοργανική Συμφωνία για την καλύτερη νομοθέτηση έχουμε περισσότερες δυνατότητες να περάσει. Οπότε να ευχαριστήσω και τις διάφορες επιτροπές. Η μέθοδος εργασίας μου ήταν να συλλέξω τα στοιχεία και τις απόψεις όχι μόνο μέσω γνωμοδοτήσεων όσο συνήθως γίνεται των Επιτροπών αλλά και με άλλες διαδικασίες και επειδή θεωρώ ότι ως ε, Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων πρέπει να έχουμε οριζόντια και άρα υπερασπίσιμη αντιμετώπιση και επειδή και άλλες επιτροπές συμφωνούσαν δεν προτείνω πολλές αλλαγές γιατί έλαβα υπόψη τις γνώμες των διαφόρων επιτροπών. Έχουμε κάποιες διαδικαστικές δυσχέρειες, αλλά η έκθεσή μου βασίζεται στις γνωμοδοτήσεις των επιτροπών το Κοινοβούλιο είχε πάντα ένα σταθερό στοιχείο στην αντιμετώπιση του. Είναι η πενταετής ισχύς ε, της λεγόμενης ρήτρα δύση για επανεξέταση των θεμάτων. Συμφωνούν όλες οι επιτροπές. Καταλαβαίνω ότι στην Επιτροπή δημιουργεί ε, γραφειοκρατικό άχθος, αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε περαιτέρω, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να τους βοηθήσουμε αλλά το Κοινοβούλιο θέλει να έχει το πάνω χέρι επί του κανονιστικού πλαισίου και όχι μόνο επί των επιμέρους αποφάσεων. Υπάρχουν λοιπόν δύο σχέδια εκθέσεων που σας προτείνω που περιέχουν την άποψη του Κοινοβουλίου για τα τρία βασικά νομοθετήματα συν 368 και αναμένω τις απόψεις σας και ξεκινάει και η διαδικασία τροπολόγησης για να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμά μας. Θα ήθελα πριν από την 20η επέτειο της απόφασης για την επιτροπολογία να έχουμε καταλήξει. Και αρκετά νωρίτερα αν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θέλει κανείς τον λόγο η κυρία Κάουφμαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ τον Σνάλφο Σάιρ για την εργασία του. Αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα του χρόνου που παίζει ρόλο φυσικά. Όπως ξέρετε, τα τρία θεσμικά όργανα αποφασίσαμε ότι το θέμα αυτό είναι επίγον. Πρέπει όλες οι βασικές νομοθετικές πράξεις να προσαρμοστούν στη νέα ε, κατάσταση. Νομίζω ότι κάναμε τα μαθήματά μας εντός αγωγικών εμείς εδώ εντός του Κοινοβουλίου και όλες οι επιτροπές έχουν την ίδια άποψη και αυτό έχει την αξία του. Θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο για αυτές τις νομοθετικές πράξεις. Και τονίζω το θέμα αυτό της πενταετούς διάρκειας. Υπάρχει ψήφισμα επ' αυτού το 14 νομίζω, όπου τονίσαμε ότι θεωρούμε ότι πενταετής περίοδος για την περιορισμένη μεταφορά είναι κάτι ε, που θέλουμε να προωθήσουμε και συμφωνεί και η ομάδα μου επ' αυτού. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή θέλει να προσθέσει τίποτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και είμαι εντυπωσιασμένος από την εργασία του εισηγητή σας και από τις γνωμοδοτήσεις. Η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση αυτή πριν το τέλος του 2016 σεβόμενη τη δέσμευσή της για καλύτερη νομοθέτηση. Είναι μια δεύτερη προσπάθεια για να υπάρξει αυτή η ευθυγράμμιση των νομοθετημάτων με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που εισήγαγε η Συμφωνία της Λισαβόνας. Όπως τα είδατε, η Κομισιόν έχει αλλάξει προσέγγιση σε σχέση με την πρώτη της προσπάθεια. Ε, γίνεται αναδιάταξη ε, προσπάθεια τροποποίησης. Δεν είναι αυτή η αυτόματη προσπάθεια προσαρμογής που απέτυχε. Και κάτι που μπορεί να έχει σημασία για τον επικείμενο τριμερή διάλογο, η Κομισιόν έχει μια εντελώς μη πολιτική, μια ε, ουδέτερη. Προσπαθούμε να προσαρμόσουμε το παλιό πλαίσιο στις ε, ή εφαρμοστικές πράξεις. Επειδή Οι περισσότερες νέες πράξεις τροποποιούν τα βασικά νομοθετήματα και αυτό γίνεται μέσω κατοεξοδότηση πράξης. Κάναμε όμως ε, αξιολόγηση αναπερίπτωση και ορισμένες λοιπόν θα γίνουν μέσω εφαρμοστικών πράξεων. Γιατί θεωρούμε ότι ήταν περιπτώσεις ε, καθαρά πραγματικά εφαρμοστικής φύσης. Κάποιες επιτροπές από ό,τι είδαμε και το αναφέρει και η εκθεσή σας, το Κοινοβούλιο επιθυμεί να γίνει προσαρμογή μέσω κατεξοδότηση πράξεων. Θα φαντάζεστε βέβαια ότι στο Συμβούλιο η τάση είναι αντίστροφη. Πολλές προτάσεις της Επιτροπής θέλουν να εφαρμόζονται μέσω εφαρμοστικών πράξεων. Άρα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Και κάτι ακόμη. σε κάποια επιτροπή και περιλαμβάνεται και στην έκθεση τη δική σας τώρα σε κάποια επιτροπή προτάθηκε λοιπόν να γίνει κάποια απάλληψη. Αυτό σημαίνει ότι αν θέλετε να αλλάξετε κάτι γιατί έχει υπάρξει τεχνική πρόοδος για παράδειγμα θα έπρεπε να γίνει νέα νομοθέτηση θα πρέπει να συζητήσουμε πολύ πιο αναλυτικά αυτές τις καταστάσεις στον επερχόμενο λοιπόν τριμερή διάλογο και παραλαμβάνω αυτό που είπα η Κομισιόν συστηματικά προτιμάει μία διοική προσέγγιση. Δεν θέλουμε να έχουμε πολιτική ε, χορήγηση εξουσιών ο εισηγητής έδειξε το θέμα της πενταετούς διάρκειας Νομίζω ότι έχουμε όλοι, νομίζω ότι υπάρχουν όλες τις δυνατότητες για να ανακληθεί μια χορήγηση εξουσιών, αλλά αυτή είναι η κυρίαρχη άποψη στο Συμβούλιο, άρα πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Ευχαριστώ. Προθεσμία για τροπολογίες 12 Δεκεμβρίου. 12 το μεσημέρι. Οπότε κλείνουμε τα 32 και 33. Πριν από την ακρόαση θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα 35-38 αξιολόγηση των ε, ε, εφαρμοστικών πράξεων ή άλλα μέτρα ελέγχου. Εν, συντομία, θα ελέγξουμε τις, της εκτελεστικής πράξεις Κομισιόν, τέσσερα έγγραφα. Τα τρία πρώτα αφορούν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τα οποία πρέπει να προσαρμοστούμε. Και το τέταρτο αφορά μια απόφαση χρηματοδότησης για την χρηματοδότηση του προγράμματος δικαιοσύνη 2018. Έλεξα τα έγγραφα όλα. Δεν βλέπω κάτι που να υπερβαίνει τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κανένα μέλος της Επιτροπής αυτής ε, δεν υπέβαλε κάποια αντίρρηση. Συνεπώς ε, προτείνω να δώσουμε ε, την απαλλαγή. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, λέει ο Πρόεδρος, από τα μέλη κλείνουμε και αυτά τα σημεία και περνάμε στο σημείο 39 που είναι η ακρόαση περί κοινωνικ... Ε, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Είμαστε υπεύθυνοι για αυτό το θέμα μια και εμπίπτει στο ε, εταιρικό δίκαιο. Θέλουμε να εξετάσουμε τις τελευταίες εξέλιξεις ε, στον τομέα αυτό και επίσης να μάθουμε τι μπορούμε να περιμένουμε στο μέλλον και ιδιαίτερος πώς το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν υπόψη τις ε, κοινωνικές ανησυχίες που υφίστανται κατά τις δραστηριότητε τους. Οπότε καλωσορίζω τους ε, ομιλητές μας ε, που με την εμπειρία τους θα μας ε, διαφωτίσουν Θα δώσω το λόγο στον πρώτο μιλητή και τον του ζητώ να περιοριστεί σε 10 λεπτά, αν είναι δυνατόν. Για να μπορέσουν και τα μέλη να υποβάλουν ενδεχομένω ερωτήσεις. Στο τέλος των ομιλιών. Ο λόγος λοιπόν στον κύριο Ρόελ Νιόβενκαμπ, ε, πρόεδρος της ομάδας εργασίας του ΟΣΑ για τις ε, υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές. Θα μας παρουσιάσει τις κατευθύνσεις γραμμές του ΟΣΑ για τις πολυεθνικές εταιρείες στην πράξη και το ρόλο των εθνικών σημείων επαφής ε, στην υπεύθυνες, επιχειρηματικέ επιχειρηματικές

Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, Πρόεδρε, σήμερα για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Τις τελευταίες εβδομάδες ακούμε για τη Συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα, αλλά πολλοί δεν ξέρουν ότι υπάρχει και μια Συμφωνία των Παρισίων για την, ευθύνη, την εταιρική ευθύνη, δηλαδή για την υπεύθυνη επιχειρηματική ε, συμπεριφορά. Και είναι μοναδική αυτή η συμφωνία στον τομέα της ε, εταιρική ευθύνη για δύο λόγους. Καταρχάς, είναι δεσμευτική για τις κυβερνήσεις δηλαδή έχει την ίδια νομική ισχύ όπως και μια συνθήκη και βασικά αυτό που είπαν οι κυβερνήσεις ε, του ΩΣΑ και άλλες που έχουν συνυπογράψει αυτό, αυτή τη συμφωνία ε, ήταν να κάνουν ένα εθνικό σημείο επαφής, φρικτό όνομα για μια, ένα μηχανισμό παραπώνων ένα δεύτερο στοιχείο που συμβάλλει στη μοναδικότητα αυτής της συνθήκης υπάρχει ένας μηχανισμός όντω παραπώνων παγκόσμιος που προσπαθεί να λύσει προβλήματα που έχουν επισημανθεί στα εθνικά σημεία επαφής από συνδικάτα, μικιό, τοπικές κοινότητες ή αυτόχθονες λαούς και ε, ο μηχανισμός αυτός ε, από το 2011 έχει σχηματιστεί και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει μάλλον επεκταθεί. Επειδή όλα αυτά ακούγονται αρκετά αφηρημένα θα σας δώσω ένα δύο παραδείγματα για το τι κάνει αυτός ο μηχανισμός εδώ έχουμε ένα παράδειγμα, όλοι ξέρετε ότι Heineken είναι μια διάσημη μπύρα, πιείτε κι άλλοι, πιείτε κι άλλοι. Υπήρξε όμως ένα, μια καταγγελία που κατετέθη στο Εθνικό Σημείο επαφή της Ολλανδίας πριν από δύο χρόνια και σχετιζόταν με ένα θέμα που είχε, γίνει, είχε λάβει χώρα πριν από 15 χρόνια σε μια από τις θηγατρικές της Heineken στο Κονγκό. Τότε δηλαδή ε, ε, αγνοούνταν 68 ε, άνθρωποι ψέματα, ε, ε, απολύθηκαν 68 ε, άνθρωποι και αυτά όλα στην μέση του εμφυλίου πολέμου. Άρχισαν διαπραγματεύσει λοιπόν τα σημεία επαφή με την Χάινεκεν και τα δύο μέρη ενήργησαν πολύ υπεύθυνα και βρέθηκε μία ενδιάμεση συμφωνία ώστε όλος αυτός ο κόσμος αποζημιώθηκε για τις απώλειες της εκείνες τις εποχές Πολύ καλό παράδειγμα για το πώς ε, περίπλοκα ζητήματα εταιρικής ευθύνης μπορούν να λυθούν με αυτό το μηχανισμό. Ας πούμε, βλέπετε εδώ τώρα πάνω αριστερά τα, ό,τι απέμεινε από το Ράνα Πλάζα το εργαστάσιο στο Μπαγκλαντές που κατέρευσε με πάνω από 1.100 νεκρούς, κυρίως ε, γυναίκες. Έχουμε υποθέσεις με ε, για το Ραναπλάζα, Πλάζα, κάποιες ε, λύθηκαν και από το Δανέζικο ε, σημείο επαφής έχουμε ακόμα μια υπόθεση και στη Γερμανία επίσης καταγγελία κατά του ελεγκτή. του εργοτού ελεγκτού του Ραναπλάζα, γιατί δεν το πιστέψετε, αλλά είχε γίνει έλεγχο στο Ραναπλάζα. Δεξιά βλέπετε μια υπόθεση που μας απασχολεί από το ελβετικό σημείο επαφής. Ε, έγινε παράπονο από ένα συνδικάτο ε, κατά της FIFA που διοργανώνει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στο Κατάρ τα καλά νέα είναι ότι η FIFA και οι εργαζόμενοι βρήκαν μια συμφωνία μεταξύ τους με την αιγίδα του Εθνικού Σημείου Επαφής και με βάση τις κατευθύνσεις γραμμές του ΟΣΑ. Καταρχάς η FIFA τώρα θα ασκήσει τη δέουσα επιμέλεια στα έργα που θα κάνει στο μέλλον, αλλά και θα γίνονται και επιθεωρήσεις στους χώρους εργασίας στα εργοτάξια του Κατάρ. Αυτό δεν αφορά μόνο αναπτυσσόμενε χώρε. Βέβαια. Αυτό δε, Πολλοί πιστεύουν ότι η εταιρική ευθύνη αφορά μόνο αναπτυσσόμενε χώρε, Όχι, δεν είναι καθόλου αλήθεια αυτό. Γιατί κάτω δεξιά βλέπετε το τάρανδο των, του λαού των Σάμι που είναι αυτόχθον λαός στα βόρεια της Νορβηγίας που είναι κτηνοτρόφοι ε, ταράνδων νομα, ε, νομάδες και κάποιοι θέλησαν εκεί να φτιάξουν ένα πάρκο ε, σε βοσκοτόπια ταράνδων. Ήρθαν λοιπόν οι Σάμι στο σημείο παραπώνων της Νορβηγίας και πάλι υπήρξε μια συμφωνία διαμεσολάβηση όπου οι Σάμι αποζημιώθηκαν για το πρόβλημά τους. Recent examples that have been solved. Αυτά είναι πρόσφατα παραδείγματα και δείχνουν την προστιθέμενη αξία αυτών των σημείων επαφής στον τομέα τη εταιρική Ευθύνη. Ακούσατε ότι δεν ποτέ δεν λέω CSR, δηλαδή εταιρική κοινωνική ευθύνη, γιατί δυστυχώ αυτό έχει πολύ κακό όνομα. Σε πολλά μέρη εκτός της Ένωσης πραγματικά συνδέεται με την φιλανθρωπία. Δεν έχω τίποτα κατά τη φιλανθρωπία, αλλά υπεύθυνη, εταιρική, μάλλον εταιρική ευθύνη, όπως λένε ε, λέει ο είναι πολύ πιο εμπεδομένο στη δομή κάθε εταιρεία. Δεν είναι θέμα δημοσίων σχέσεων, δεν είναι θέμα για ωραία λόγια ή ωραία σχέδια, αλλά σημαίνει την ε, ένταξη ε, της εταιρική ευθύνης μέσα στις βασικές λειτουργίες της κάθε εταιρεία. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι δεν είναι δεσμευτικό για τις εταιρείε αυτό δεν πρόκειται για δικαστήριο, αλλά για έναν μηχανισμό επίλυσης διαφορών και προβλημάτων. Είναι υπέρ των εταιριών. Δεν είναι κατά των εταιριών. Είναι μια εξυπηρέτηση των εταιριών που τις βοηθά να ξεφύγουν από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Γι' αυτό και είναι μοναδικός μηχανισμός αυτός. Δεν είναι νομικό δεσμευτικό για τι εταιρείε, αν και υπάρχουν μεγάλε προσδοκίε από τι κυβερνήσει. Σε 48 κυβερνήσει του ΩΣΑ που αναμένουν αυτό το είδος τη συμπεριφορά από τις μεγάλους ομίλους. Υπάρχουν επίσης μαρτυρίες ότι δεν είναι μόνο το σωστό που πρέπει να κάνει κανείς, αλλά και από εταιρική προοπτική είναι το έξυπνο πράγμα που πρέπει να κάνει κανείς, γιατί πολλές έρευνες αποδεικνύουν ότι πολλές εταιρείες που λειτουργούν έτσι υπεύθυνα έχουν και καλύτερες επιδόσεις ε, οικονομικά, οικονομικές. Εδώ να σας δείξω το σύστημα εθνικών ε, σημείων επαφής. Πρόκειται για έναν οικουμενικό μηχανισμό γιατί καλύπτει ε, μια οικουμενική αλυσίδα αξίας. Το δανέζικο σημείο μπορεί να λύσει ζητήματα στον Μπαγκλαντές που δεν είναι μέλος του ΩΣΑ. Η κινέζικη εξαγωγική ε, βιομηχανία προς τη ΣΥΠΑ επίσης καλύπτεται από τις κατευθυντήριες γραμμές του ΩΣΑ. Μπορούμε να λύσουμε θέματα διαφθοράς στο Μαλί ή το Καμερούν. Είναι λοιπόν οικουμενικός αυτός ο μηχανισμός, βασικά προσπαθεί να λύσει βασικά προβλήματα. Θα δείτε ότι πολλά ζητήματα που έρχονται στα σημεία επαφής μας αφορούν πολύ καλές εταιρείες, αλλά οι προκλήσεις είναι τεράστιες. Για παράδειγμα, η Coca-Cola μόνο έχει γύρω στις 10, 10 εκατομμύρια αγρότες που δουλεύουν ε, στα ζαχαρότευσλα. Η Nestlé, οι Unilever έχουν 100.000 προμηθευτές, πάνω από 100.000 προμηθευτές. Δεν θα μπω σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά είναι σημαντικό να τονίσουμε, νομίζω, τον αντίκτυπο του συστήματος. Πολλής λόγος γίνεται γι' αυτό και ξέρετε, ΜΚΟ δεν είναι τόσο ενθουσιώδης γιατί προτιμούν ένα δικαστήριο για την εταιρική ευθύνη, για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, CSR, έχουν ε, λοιπόν ένα σωρό βρεθεί και πολλά ωφέλη, ας πούμε, ε, βελτιωμένη υγεία και ασφάλεια, ε, βελτιωμένος διάλογος εργοδότη-εργαζομένων, ας πούμε η πάυση της εκμετάλλευσης ε, των ε, προστατευόμενων δρυμών όπου ζουν οι γορίλες στο Κονγκό, ένα σωρό ωφέλη. Soft law Αυτή η ήπια νομοθεσία τίνει να γίνει σκληρότερη. Ας πούμε, οι διάφορες, τα διάφορα γραφεία ε, εξαγωγικά θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ε, δηλώσεις που αφορούν την κάθε εταιρεία από το Εθνικό Σημείο Επαφής γιατί αν μια εταιρεία δεν λειτουργεί καλή την πίστη δεν θέλει να δεχτεί τη διαβούλευση θα χάσει την υποστήριξη της οικονομικής διπλωματίας του Καναδά ας πούμε η συγκεκριμένη αλλά ε, περισσότεροι ισχύ, ε, ε, περισσότερο εξετάζουν και οι σε την εταιρική ευθύνη, πώς λειτουργεί η κάθε εταιρεία και πιέζουν το κάθε εταιρεία για να λύσουν αυτά τα θέματα. Αυτή είναι η τάση λοιπόν. Μια άλλη τάση έχει να κάνει με τη δέουσα επιμέλεια, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες, αλλά βασικά η ευθύνη της αλυσίδας προμηθειών έχει ενταχθεί στον εγχειρίδιο του ΟΗΕ και του ΟΣΑ αλλά και στην δήλωση την τελευταία του Διεθνούς ε, Γραφείου Εργασίας δέουσα επιμέλεια είναι αυτή που πρέπει να διέπει την αλυσίδα προμηθειών. Περισσότερες εταιρείες ε, δεν καθιστούν αυτή τη δέουσα επιμέλεια υποχρεωτική. Ε, κυβερνήσεις με συγχωρείτε, και το κοινοβούλιο, τα κοινοβούλια ακολουθούν αυτή τη τάση γιατί για τα ορυκτά των ε, συγκρούσεων ε, έχουν καταστήσει υποχρεωτική εκεί την εφαρμογή της εταιρικής ευθύνης. Υπάρχουν και για τις αλυσίδες της υφαντουργίας. Στη Γαλλία γίνεται λόγος για νομοθετήματα περί δουλείας πάλι στο πλαίσιο της εταιρική ευθύνης. Υπάρχουν λοιπόν εγχειρίδια για τη δέωση επιμέλεια ανατομέα, ανακλάδο. Αυτή είναι η δουλειά που έχουμε κάνει ανάλογα με τον κάθε τομέα. Και τέλος θέλω να πω για όλα αυτά, όλες αυτές τις νομικές εξελίξεις θα πρέπει να είμαι ε, ουδέτερος γιατί η Γαλλία είναι μέλος της δικής μου επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Ένωση, Δεν είμαι ούτε υπέρ ούτε κατά όσον αφορά τον υποχρεωτικό χαρακτήρα. Αυτό όμως που δεν μπορώ να είμαι ουδέτερος είναι ότι πρόκειται για πολιτικές που δεν βασίζονται σε μαρτυρίες. Δεν ξέρουμε τι κάνουν οι εταιρείε. Και οι ΜΚΟ λένε ότι οι εταιρείε δεν κάνουν τίποτα. Ε, οι εταιρείε λένε ότι κάνουν ό,τι πρέπει. Αλλά στην πράξη η πολιτική ασκείται στα τυφλά. Μόνο στη Γερμανία, και αυτό θέλω να το τονίσω, στη Γερμανία υπάρχει μία συμβιβαστική στο Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης για την ε, εταιρική ευθύνη που λέει ας αρχίσουμε πρώτα να μετράμε τι κάνουν οι εταιρείε και μόνο εφόσον οι γερμανικές εταιρείε αποδειχθεί ότι κάτω από το 50% εξ αυτών έχουν στεναρό σύστημα δέουσας επιμέλειας με το 2020 τότε θα εξετάσουμε τις ε, υποχρεωτικές ε, επιλογές. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα συμβιβασμό ανάμεσα σε αυτού που πιστεύουν και σε αυτού που δεν πιστεύουν, αλλά εν πάση περιπτώσει το καλό είναι ότι θα προκύψει και κάποια νομοθεσία με πολιτική με βάση τι ε, μαρτυρίε και, και τα, τα στοιχεία. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω πως η μέτρηση της καλής θετική δουλειά των εταιριών είναι απαραίτητη. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα θα ακούσουμε την κυρία Γκρανζόν που είναι μέλος της Γαλλικής ε, Εθνοσυνέλευσης. Εσείς προωθείτε μια πράσινη κάρτα για την κοινωνική εταιρική ευθύνη που έχει υποστηριχθεί από ε, νέα εθνικές συνελεύσεις και από την γαλλική νομοθεσία, την πρόσφατη γαλλική νομοθεσία για τη δεωση επιμέλεια για τις μητρικές εταιρείες και τις θηγατρικές εταιρείες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ σήμερα να σας μιλήσω για την ε, ε, εταιρική κοινωνική ευθύνη. Ε, πολλοί εδώ και χρόνια κρούν τον κοντάνα του κινδύνου σε ό,τι αφορά τις ε, πολυεθνικές εταιρείες και τις θυγατρικές τους, καθώς επίσης και των προμηθευτών τους και των εταιρεών στις οποίες κάνουν υπεργολαβία. Η έλλειψη αυτής της κοινωνικής ευθύνης ενθαρρύνει πρακτικές ε, των οποίων οι συνέπειες μπορεί να είναι δραματικές, όπως για παράδειγμα στη βιομηχανία του κοβαλτίου. Ε, είμαι πεπισμένη ότι οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να περιορίζονται στο να αυξήσουν τα κέρδη του, έχουν και μια κοινωνική ευθύνη και δεν θα πρέπει να κρύβονται πίσω από την ευθύνη ε, των θηγατρικών τους ή των υπεργολάβων τους ή των προμηθευτών του είναι ευθύνη δική μας, ε, αν οι νόμοι δεν το επιβάλλουν αυτό, να το καταστήσουμε δυνατό. Θα ήθελα να σας αναφέρω τις ε, πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, που έχουν αναλυθεί τα τελευταία χρόνια ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2010 έχει οθετήσει αρκετούς κανονισμούς, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά και τα υπερβαλλοντικά δικαιώματα, για, το διαμα, για τη ε, βιομηχανία του διαμαντίου του 2002, του ξύλου του 2010 και των ορυκτών ε, το 2017. Επιπλέον έχουμε το μη οικονομικό reporting, την υποβολή εκθέσεων του 2014 μέσω της εφαρμογής ενός ε, συστήματος ε, επιμέλειας, δεύουσας επιμέλειας για το, την προέλευση ε, των πρώτων υλών για διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα για το ξύλο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε το αυτή την εθελοντικής ε, συμμετοχής, ε, ε, το συμμετοχή σύστημα να γίνει υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα ορυκτά. Η, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση δημιούργησε το σύστημα της πράσινης κάρτας Κάτι που οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια φιλόδοξη νομοθετική πρόταση για το ίδιο θέμα. Θα εφαρμοζόταν σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το σύστημα, ανεξαρτήτως της δραστηριότητά τους, με ένα, ενδεχομένως ένα κατόφλι, έτσι ώστε οι, οι πιο μικρές επιχειρήσεις να μην συμπεριληφθούν ε, θα περιέλαμβανε συγκεκριμένες υποχρεώσεις ό,τι αφορά την, ε, τον έλεγχο και την φροντίδα ε, των θυγατρικών τους εταιριών, των υπεργολάβων τους και των προμηθευτών τους για να για ένα σύνολο θεμάτων όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά δικαιώματα και άλλα. Τέλος, θα προέβλεπαν αυτοί οι κανόνες συγκεκριμένες κυρώσεις αποτελεσματικές, αναλογικές ε, και αποτρεπτικές ε, ενδεχομένως αναλογικές των, της ζημιάς που έχει προκληθεί. Αυτή η πράσινη κάρτα δεν αναπτυχθήκε, δεν υλοποιήθηκε στην Γαλλία, αλλά η συζήτηση δεν έχει κλείσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, δεδομένων και των τελευταίων ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για παράδειγμα το ψήφισμα της 25 η Οκτωβρίου 2016 για την ευθύνη των επιχειρήσεων σε θέματα σημαντικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτε χώρε. Στο άρθρο στο παράγραφο 28 αναφέρει ε, ότι σε, ε, ε, τις προθέσεις ε, της, ε, των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τον ιδιωτικό τομέα και για τις αλυσίδες προμήθειας που θα είναι πιο αποτελεσματικές, πιο επέφθυνες. Όλες αυτές οι, εθνικές, οι εθνικές πρωτοβουλίες τις οποίες αξιολογεί η Κομισιόν όπως και της Γαλλίας συνυπάρχουν με τις, με τις δραστηριότητες της Κομισιόν. Ε, το 2013 μετά το δράμα του Ράνα Πλάζα η πρόταση της, ε, η πρόταση, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγινε νόμος το 2017 ο νόμος αυτός τι λέει στη Γαλλία, λέει, δημιουργεί την ε, υποχρέωση για τις εταιρείε που απασχολούν ε, οι ίδιες ή θηγατρικές τους τουλάχιστον 5.000 εργαζόμενους στη Γαλλία ή τουλάχιστον 10.000 σε όλο τον κόσμο να διαθέτουν ένα πρόγραμμα ε, ε παρακολούθησης και να το εφαρμόζουν. Αυτό το πρόγραμμα θα έχει ε, λογικά μέτρα για να αποφευχθούν ε, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τη, επίσης εναντίον της υγείας και της ασφάλειας, καθώς επίσης και του περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει τις ίδιες εταιρείε, τις θηγατρικές τους, έμεσες και άμεσες, ε, τους υπεργολάβους τους και τους προμήθευτές τους με τους οποίους έχουν ε, εμπορικές ε, σχέσεις σχετικές με τη δραστηριότητά τους. Περιλαμβάνει ιδιαίτερα τα εξή μέτρα. Ένα, μια χαρτογράφηση των κινδύνων, μια τακτική αξιολόγηση της κατάστασης των θηγατρικών υπεργολάβων και προμηθευτών, δράσεις για τη μείωση των κινδύνων, την πρόληψή τους, ένα μηχανισμό εκτακτής ανάγκης, και ένα μηχανισμό για την αξιολόγηση των μέτρων που λαμβάνονται. Αυτή η υποχρέωση ε, για την κατάρτιση ενός ε, σχεδίου παρακολούθησης ε, δεν θα αρκούσε αν δεν υφίσταντο και κυρώσεις. Και υπάρχουν δύο ειδών κυρώσεων. Πρώτον, ο νόμος προβλέπει ότι αν μια εταιρεία δεν δημιουργήσει, ε, δεν συστήσει τέτοιου είδου ε, σχέδιο, έχει τρει μήνες για να το κάνει. Μετά από αυτό, οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος ή εμπλεκόμενος, μπορεί να είναι συνδικαλιστές, μια οργάνωση, μια, κυβερνητική οργάνωση κλπ, ε, οι ίδιοι εργαζόμενοι μια μιας μπορεί να προσφύγουν στα δικαστήρια για να εξαναγκαστεί η επιχείρηση να συστήσει συντάξει αυτά του είδου τα σχέδια. Δεύτερη κύρωση η αστική ευθύνη η οποία μπορεί να δημιουργηθεί ε, με δυνατότητα να ζητηθεί αποζημίωση μετά από απόφαση της δικαιοσύνη. Τέλος, στον νόμο αυτό προβλέπεται η δυνατότητα ένας δικαστής ε, να επιβάλλει πρόστιμο ε, σε μια, τέτοια, σε μια εταιρεία, ενδεχομένως και αποζημίωση έως 30.000 ευρώ. Ε, αυτή η απόφαση, αυτή η δυνατότητα όμως έχει προσληφθεί στο συνταγματικό δικαστήριο. Ε, η, τα σχέδια παρακολούθησης ε, δεν θα είναι μια τυπική υποχρέωση. Ε, με, βάση, με αυτές τις κυρώσεις που έχουν προβλεφθεί θα γίνουν μια πραγματικότητα ο έλεγχος των ε, θηγατρικών εταιριών και των ε, εμπορικών εταίρων θα, είναι, θα γίνει υποχρεωτικά ε, ακόμα και όταν ε, οι θηγατρικές δεν ελέγχονται πλήρως οι, οι προμηθευτές. οι δικαστές θα αξιολογούν τα προληπτικά μέτρα τα οποία προλαμβάνουν τα σχέδια παρακολούθησης και θα ε, προβλέπουν και θα μπορούν να επιβάλλουν και συγκεκριμένες ε, ε, κυρώσεις όπως η υποχρέωση διακοπής εμπορικών σχέσεων με συγκεκριμένους προμηθευτές κλπ. Για όλους τους Ευρωπαίους αυτή η διαδικασία θα πρέπει να αποτελέσει σύμβολο της ευαισθησίας μας η πράσινη κάρτα που θα μπορούσαν να λαμβάνουν με βάση τέτοιους νόμους οι επιχειρήσεις θα αποτελεί μια πρόσθετη, θα τους δίνει μια πρόσθετη αξία ε, και θα βελτιώνει ε, την, το κύριο του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα ο τρίτος μας ομιλητής. Ο κύριος Νταν Ρις που είναι διευθυντής του προγράμματος για καλύτερη εργασία του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Το πρόγραμμα Καλύτερη Εργασία είναι ένα εργαλείο για την βελτίωση των συνδικών εργασίας και της ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια βιομηχανία ενδυμάτων και υποδημάτων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας για την δυνατότητα που μου δίνετε για να εκπροσωπήσω το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας για την προσπάθεια που κάνει για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας μέσω του προγράμματος μας αυτού και ιδιαίτερα στην ένδυση και υπόδηση. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα, καλύτερη εργασία. Είμαστε εταιρική σχέση μεταξύ του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και της, ε, ε, του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης που είναι παράρτημα της Παγκόσμιας Τράπεζας. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε και τη λειτουργία των επιχειρήσεων και την ανταγωνιστικότητα. Εργαζόμαστε σε 8 χώρες με πολλές εταιρείες στην αλυσίδα προμηθειών, με εθνικούς εμπλεκομένους τους ε, εργαζόμενους, τους εργοδότες και τις κυβερνήσεις. Συνεργαζόμεθα με πάνω από 100 παγκόσμιους παραγωγούς και λιανοπολιτές ε, ενδυμάτων και δίνουμε υπηρεσίες σε πάνω από 1.500 ε, επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 4 εκατομμύρια εργαζομένων. Στόχος μας είναι να κάνουμε μια εξολόγηση των συνθήκων εργασία, να δώσουμε στους βιομηχανου ένα πρόγραμμα δράσης για βελτίωση της κατάστασης και το πρόγραμμα δράση και εκθέσεις προόδου είναι ε, διαθέσιμα σε όλου του πελάτε του, στην αλυσίδα ε, προμηθειών εφοδιασμού για να ξέρουν και εκείνοι τι να κάνουν. Τα περισσότερα κάνουμε, που κάνουμε τα κάνουμε μέσω οικοδόμησης των δυνατοτήτων των εργαζομένων και των ε, managers για να υπάρξουν ε, βιώσιμες βελτιώσεις συνθήκες εργασίας ούτως ώστε να σέβονται τον εθνικό νόμο και τα διεθνή πρότυπα εργασίας και να μπορούν να το κάνουν αυτό σε, με βιώσιμο τρόπο. Η εταιρική αυτή σχέση μεταξύ αυτών των δύο οργανισμών μας έγινε με βάση συλλογή στοιχείων. Είχαμε μια ανεξάρτητη μελέτη αντικτύπου πενταετή που έκαναν ανεξάρτητη πανεπιστημιακή, έγινε σε πέντε χώρες. Είναι η μεγαλύτερη τέτοιου τύπου μελέτη που έχει γίνει ποτέ. Περιλάμβανε στοιχεία και ερωτηματολόγια από πάνω από 15.000 εργαζομένους και χιλιάδες ε, στελεχών επιχειρήσεων. Θέλαμε λοιπόν να βελτιωθεί η κατάσταση στα εργοστάσια και αν βελτιωθεί η κατάσταση σε τι βασίζεται και τι αντίκτυπο έχει στους εργαζομένους, στις οικογένειές τους, ε, για τις επιχειρήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού και για την περαιτέρω πρόοδο των επιχειρήσεων. Είναι μια μοναδική προσπάθεια. Είναι μοναδική αυτή η έκθεση. Ποια είναι τα πορίσματα αυτής της έκθεσης λοιπόν. Πρώτον, το πρόγραμμα αυτό είχε μεγάλη επιτυχία στη βελτίωση των συνθηκών εργασία σε όλε τι χώρε όπου εργαζόμεθα. Μείωση των διακρίσεων και τη ε, καταναγκαστικής εργασία, αύξηση των ε, εβδομαδιαίων αποδοχών από, με πάνω σε πάνω από 15 λίρες τη βδομάδα στο Βιετνάμ, μείωση των ωρών εργασίας σε πολλά ε, εργοστάσια, στη χορήγηση μονίμων συμβολέων αντί για προσωρινών συμβολέων σε πολλούς εργάτες και ναι μεν δεν επιτύχαμε σε όλα αλλά επιτύχαμε σε πολλά για να, να εφαρμόζεται και η εθνική εργασιακή νομοθεσία και οι διεθνείς προδιαγραφές. Ποια είναι η βάση της αλλαγής. Είναι η συμμετοχή όλων και των οργανώσεών τους. Αλλά όταν εξετάσαμε τι ακριβώς ήταν η βάση της αλλαγής, ο, κινητήρας, ο κινητήρας της αλλαγής, ταυτοποίησαν δύο στόχους. Πρώτον, η σημασία του κοινωνικού διαλόγου. Τα εργοστάσια που είχαν μηχανισμούς ποιότητας και δυνατότητες ε, διαλόγου των εργαζομένων με τους ε, ε, διοικούντες, τα πάνε καλύτερα. Και το δεύτερον, η ενθάρρυνση της πλήρους συμμετοχής των, των γυναικών στην ε, οικονομική δραστηριότητα. Έτσι μειώνεται και το χάσμα στις αποδοχές και το χάσμα στις ώρες εργασίας στην Αιτή, στο Βιετνάμ, την Ικαράγουα και μειώθηκαν οι ανησυχίες των γυναικών για σεξουαλική παρενόχληση και δόθηκε περισσότερη πρόσβαση στην ε, ε, φροντίδα κατά την εγκυμοσύνη. Και κάτι άλλο που εντόπισαν οι ερευνητές μας. Εκεί που συνεργαστήκαμε και με τους εργαζόμενους και με τους εργοδότες επιτύχαμε να προωθήσουμε και τη θέση των γυναικών και για να τα πάνε καλύτερα και οι επιχειρήσεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Κάναμε μία έρευνα μεταξύ των εργοστασίων όπου δώσαμε κατάρτιση ε, στους, ε, στα στελέχη για να είναι και ε, στελέχη που ασχολούνται και με τη διαχείριση του προσωπικού. Και διαπιστώσαμε ότι στα εργοστάσια αυτά, σε σύγκριση με εργοστάσια που δεν έχει δοθεί αυτή η κατάρτιση, οι επιχειρήσει θα πήγαν 22% καλύτερα. Και πολλέ φορέ όταν οι επιστάτε των εργαζομένων ήταν γυναίκε, τα πράγματα ήταν ακόμη καλύτερα. Κάτι άλλο. Η επένδυση στη βελτίωση των συνδικών εργασία είναι επένδυση, όχι κόστος. Έχουμε πολλά παραδείγματα αυτού σε όλες τις χώρες όπου εργαστήκαμε. Και εδώ ένα παράδειγμα από το Βιετνάμ. Εντοπίσαμε ότι στα εργοστάσια όπου οι εργαζόμενοι είπαν αισθανόμαστε ασφαλείς, ότι δεν υφιστάμεθα διακρίσεις, όπου ξέρουν σε ποιον να διαμαρτυρηθούν και όπου τους πλήρωναν με βάση το συμβόλαιό τους, στα εργοστάσια αυτά διαπιστώσαμε 8% περισσότερη κερδοφορία σε σχέση με τα εργοστάσια όπου οι εργαζόμενοι είπαν ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και στο Βιετνάμ, ε, αν ήταν παρόμοιες άλλες συνθήκες, η έρευνα κατέληξε ότι σε πενταετή βάση βελτιώνεται κατά 25% η κερδοφορία του εργοστασίου. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα εργοστάσια κατασκευής ε, ε, ε, ρούχων πολλές φορές έχουν τη φήμη ότι έχουν σκληρές συνθήκες. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Και όταν εξετάσαμε τι συμβαίνει και στα σπίτια των εργαζομένων και στις γειτονιές όπου μένουν, όταν είδαμε ότι οι εργαζόμενοι είχαν περισσότερο χρόνο και περισσότερο εισόδημα για να ασχοληθούν με την οικογένειά τους, για να αφιερώσουν και χρήμα και χρόνο στην οικογένειά τους και για να μειώσουν τα χρέη τους και για να στείλουν και ε, εμβάσματα πίσω στη χώρα, για παράδειγμα, ή την περιοχή προέλευσή τους, τότε βελτιώνεται και η ανάπτυξη των κοινοτήτων προέλευσης και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα του προγράμματος. Και τελικό πόρισμα. Οι επιχειρήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού έχουν σημαντικό ρόλο επιλέγοντας από πού να εφοδιαστούν. Σημαντικό ρόλο για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. 80% των ε, διευθυντικών στελεχών εξέφρασαν ανησυχία για την αρνητική επίπτωση πρακτικών όπως τελευταία, τελευταία στιγμή αλλαγή στις παραγγελίες. Θεωρούν ότι τέτοιες πρακτικές δημιουργούν ανάγκη για αύξηση των ορών εργασίας, περισσότερα ατυχήματα και περισσότερη πίεση και ε, κατά, ε, πίεση των εργαζομένων. Καταλήγοντας. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα η μελέτη αυτή. Μοναδική όπως είπα, έχουμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία από πολλές επιχειρήσεις. Εξετάσαμε το, το αντίκτυπο λοιπόν της ε, βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, την ε, απόδοση των επιχειρήσεων και στη βελτίωση της αλυσίδας εφοδιασμού. Ακόμη λοιπόν και σε ένα κλάδο εντατικό εργασίας και υψηλής ε, έντασης το να δώσεις φωνή στους εργαζόμενους, το να τους δώσεις δυνατότητες να επικοινωνήσουν, να μπορούν ε, να ε, υποβάλουν παράπονα που να ληφθούν υπόψη, όλα αυτά προωθούν αλλαγές στα εργοστάσια και οι επιχειρήσεις που το κάνουν αυτό είναι πιο επικερδείς. Ιδιαίτερα μεταξύ των επιχειρήσεων τις οποίες εξετάσαμε. Και αν δούμε τι θα γίνει στο μέλλον και ανεξάρτητα από την εισαγωγή περαιτέρω τεχνολογίας στον κλάδο αυτό και άλλες έντας εργασίας, είναι σίγουρο ότι ο κλάδος αυτός θα παράσχει εκατομμύρια θέσεων εργασίας σε περιοχές που χρειάζεται εργασία. Αν αυτές οι δουλειές είναι αξιοπρεπείς, τότε ο κλάδος μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα για ένταξη χωρίς αποκλεισμού των κοινωνιών γιατί οι θέσεις αυτές θα πάνε στο 40% χαμηλότερων αμοιβών σε εργαζόμενους που για πρώτη φορά εργάζονται, δηλαδή γυναίκες και νέους. Και όταν ε, τα άτομα αυτά μπορέσουν να ξεφύγουν από τη φτώχεια μέσω αυτών των αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, τότε θα ξεφύγουν και οι οικογένειες και οι κοινότητές τους. Ευχαριστώ πολύ. συγγνώμη πρέπει να ζητήσω καταρχάς ε, από τον απόμενο μιλητή, ο κύριος Βιντάν Κέτφλικ, πρόεδρος της ομάδας εργασίας για την υπεύθυνη συμπεριφορά των επιχειρήσεων στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Η προοπτική των επιχειρήσεων για τις ε, γραμμές του ΟΣΑ για τις πολυεθνικέ επιχειρήσεις. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ονομάζομαι Κράτη Φλίχα και αυτό το όνομα είναι ειδικά φτιαχμένο για διεθνείς σχέσεις. Ε, να σας δώσω την ε, άποψη της ΠΙΑΚ όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές ε, του ΟΣΑ. Είναι η Συμβουλευτική Επιτροπή των Ομίλων και των Εταιριών προς τον ΟΣΑ και συστήθηκε όταν ξεκίνησε και ο ΟΣΑ ώστε να ε, μπορεί να συμμετέχει στην διαδικασία του ΟΣΑ. Το να είναι κανείς ε, υπεύθυνος ε, ε, ε, είναι προς το συμφέρον του διεθνούς επιχειρηματικού κλίματος. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία από τη μια πλευρά μέσα στο άνοιγμα προς τις διεθνείς επενδύσεις και από την άλλη πλευρά την ευθύνη. Τα δύο βασικά μου μηνύματα για σήμερα είναι πρώτον ότι πιστεύουμε πως ο ΣΑ και οποιασδήποτε κατευθύνες γραμμές, ε, μάλλον και οι, αυτές οι κατευθύνες γραμμές είναι πολύτιμο ε, μέσο και θα πρέπει να μείνουν ε, στην καρδιά της ανάπτυξης της υπεύθυνη εταιρικής συμπεριφοράς και έπειτα υπάρχει ιδιαίτερη πρόκληση στο να υλοποιήσουμε αυτό το δυναμικό των κατευθύνων γραμμών και των εθνικών σημείων επαφής. Κατευθύνει γραμμέ είναι η πιο ολοκληρωμένη μορφή προώθησης της υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά, και όπως ήδη εξηγήθηκε από τον κύριο Νίερ Κάμπα παρέχουν ε, ε, εθελοντική ε, εταιρική ηθική και αναπτύχθηκαν σε πολύ στενή συνεργασία με τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις εταιρείε και τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ουσία είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο μέσα για την ανάπτυξη της υπεύθυνη εταιρική συμπεριφοράς ε, στις ε, ε, διεθνώς. Οι <clears throat> κατευθυντήριε γραμμέ αυτέ έχουν μάλλον δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι ευέλικτε. Είναι κατευθυντήριε γραμμέ που λένε σαφώ ότι η φύση και ο βαθμός της δέουσας επιμέλεια εξαρτάται από τις συγκεκριμένες περιστάσεις και ιδιαίτερα από το μέγεθος της κάθε εταιρεία είτε πρόκειται για μεγάλη είτε για μικρομεσαία. Δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι οι θελημένα δεν μπορούν νομικώς να επιβληθούν. Στόχο έχουν να προωθήσουν, να παροτρύνουν σε μια υπεύθυνη συμπεριφορά και όχι να ρυθμίσουν νομικές ε, ε, ε, διαμάχες ή διαφορές. Γίνονται αντιληπτές ως μια διαδικασία μάθησης εγώ, όπω είπε ο κύριο Νιουρκάμπ, ε, δεν είμαι ουδέτερο. Πιστεύω πω είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο, διότι έτσι δημιουργείται μια τελείω διαφορετική κουλτούρα, νοοτροπία στην αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Η εθελοντική, η κούση βάση στην ουσία δημιουργεί μια, ε, μια δραστήρια προσέγγιση και όχι μια αμυντική προσέγγιση. Ωστόσο, ε, δεν είναι και απόλυτα ελεύθεροι πώς θα αντιμετωπίσουν αυτές τι κατευθύνσεις γραμμές οι εταιρείε. Πρέπει να τις στηρίσουν και πρέπει να φτιάξουν μια πολιτική η οποία να είναι συμβατή με αυτές τις συστάσεις. Εμείς ως ΒΙΑΚ e Προωθούμε τις κατευθυντήριες γραμμές ανάμεσα στα μέλη μας. Έχουμε αναπτύξει, έχουμε μάλλον φτιάξει ένα φυλάδιο και ευχαρίστω σας, το στείλω στη γραμματεία σας. Οι κατευθύνε γραμμέ δεν είναι μόνο μια απέτηση από πλευρά προ τι εταιρείε. Προωθούν ένα ισότιμο πεδίο που είναι συμφέρον για τι εταιρείε και προστατεύουν τι εταιρείε από μη ρεαλιστικέ προσδοκίε από άλλε πλευρέ, από άλλου θεσμού. Είναι γεγονός ότι ένα κεντρικά αναγνωρισμένο παγκοσμίω μέσο για την υπεύθυνη συμπεριφορά των εταιριών είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ίδιες τις εταιρείες, γιατί υπάρχει σημείο αναφοράς στην υπόθεση αυτή. Και έτσι ανησυχούμε για την ε, το πιθανό πολλαπλασιασμό τέτοιων μέσων από διάφορες διεθνείς πηγές που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν ε, τα ίδια, ε, τις ίδιες και αντιφατικές προσδοκίες και για μας είναι σημαντικό να μείνει αυτό το κεντρικό σημείο. Ο τρόπος να προχωρήσουμε είναι η πρακτική συνεργασία και τα συγκεκριμένα βήματα μπροστά επί τη βάση των κατευθυντήριων γραμμών και αρχών. Και αυτή είναι και η βάση των βιώσιμων στόχων του ΟΗΕ. Πώς θα κινητοποιηθεί ενέργεια ώστε να λυθούν παγκόσμια ζητήματα, όχι να απαγορεύσουμε, αλλά να προωθήσουμε. Να αναφέρω μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία στον τομέα της εταιρική κοινωνικής ευθύνης που είναι η η υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση που αναπτύσσεται από το Ολλανδικό Οικονομικό Συμβούλιο και αυτό βασίζεται στην ιδέα ότι πολλά προβλήματα στον τομέα της υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά σε τρίτες χώρες προκαλείται από πολλαπλά προβλήματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι εταιρείε που κάνουν λάθη, αλλά είναι ο συνδυασμός περιστάσεων, περιβάλλοντος, τοπικών αρχών, και άλλων ε, συνιστοσών. Όταν θέλουμε λοιπόν να λύσουμε το πρόβλημα, η λύση δεν είναι να τα ρίξουμε στην εταιρεία και να πούμε εσείς πρέπει να αλλάξετε, αλλά να φέρουμε κοντά όλους τους εταίρους, τη τοπική κυβέρνηση, την κυβέρνηση της χώρας ε, που εδράζει η εταιρεία, της ΜΚΟ και τα λοιπά. Να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα για να δούμε σφαιρικά πώς θα το λύσουμε. Είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα αυτή. και πιστεύω πως θα ήταν χρήσιμο για το Κοινοβούλιο να οργανώσουμε ε, ε, ε, μια κρόαση για το, το, θέμα αυτό. That is the, national contact point. μηχανισμός εθνικών σημείων επαφής. Τα εθνικά σημεία επαφή είναι ένας μοναδικός μηχανισμός εφαρμογής. Τα σημεία επαφή έχουν δύο λειτουργίες. μία είναι να προωθούν τις κατευθύνσεις και η δεύτερη είναι να, μην, να παρέχουν έναν μηχανισμό παραπώνων εξοδικαστικό. Βασικά βασίζεται στη διαμεσολάβηση και στην συμφιλίωση, διαλλαγή, Δηλαδή, θεμελιώδη διαφορά ανάμεσα σε αυτό το μέσο της ε, υπεύθυνη τη εταιρεία και του νομικού μέσου. Και υπάρχει και μια ιστορία του νορβηγικού σημείου επαφή που δείχνει αυτή τη διαφορά προσέγγιση. Είχαν μια υπόθεση όπου μετά από κάποιε ε, συνεδρίε ε, ε, ήταν σαφέ πω η εταιρεία δεν είχε κάνει λάθο και κάνανε μια συνδιαλλαγή όπου ήταν εκεί ο Γενικό Διευθυντή και ο νομικό του σύμβουλο. Και κάποια στιγμή το σημείο επαφή είπε: Δεν είναι δυνατόν εσεί ω διευθυντή τη εταιρεία απλά να εκφράσετε την ε, θλίψη σας και να ζητήσετε συγγνώμη. Ναι, είμαι πρόθυμος να το κάνω αυτό, είπε ο διευθυντής και ο νομικός σύμβουλος ε, τρομοκρατήθηκε από τις πιθανές νομικές επιπτώσεις. Με δύο λόγια, αυτή είναι η ουσία, η διαφορά ανάμεσα σε μια διαδικασία ε, ε, Διευθέτηση αυτού του τύπου εξοδικαστική και της νομικής διαδικασίας που θέλει να ε, πηρύψει ευθύνες για το παρελθόν. Είμαστε πεπισμένοι για τη δυναμική και τη θετική επιρροή αυτής της προσέγγισης. Επίσης, τα σημεία επαφής ήταν ε, ε, από αντικείμενο μια κοινή δήλωση τη ΜΠΕΚ και τη αρμόδια επιτροπή του ΩΣΑ. Ήταν η μόνη φορά στην ιστορία του ΩΣΑ όπου οι τρει κοινωνικοί εταίροι έφτασαν σε κοινή θέση, σε κοινή δήλωση όπου εξέφρασαν δηλαδή την υποστήριξή του για το σύστημα των Εθνικών Σημείων Επαφής και ζήτησαν από τις κυβερνήσεις να ενισχύσουν περαιτέρω την απόδοση των Εθνικών Σημείων Επαφής και όλος ιδιαίτερος και όπου Αυτά τα σημεία επαφής έπρεπε να επιταχύνουν. Το σύστημα αυτό λοιπόν ε, λειτουργεί όχι μόνο μέσω των διαδικασιών, αλλά λόγω των συζητήσεων που ε, πυροδοτούν αυτές οι, ε, οι συνδιαλλαγές. Δεν είναι εύκολο για μια εταιρεία που δεν είναι, συνηθισμένη σε ένα τέτοιο μέσο να το χρησιμοποιήσει. Όταν όμως το κάνει, συνήθως μένει ευχαριστημένη και βλέπει ότι τα εκτήματα. Επίσης, αυτή τη διαδικασία ξεδιπλώνει τη συζήτηση και ευρύτερα στην κοινωνία. As in the guidelines, και πάλι εδώ με τις κατευθυντήριες γραμμές είμαστε πεπισμένοι ότι η ουσία αυτής της διαδικασίας ώστε να λειτουργήσει ως διαμεσολάβηση είναι πολύ σημαντική. Είχαμε μια συνάντηση με 30 πολυεθνικές εταιρείες συν την ηγεσία του ΩΣΑ το περασμένο Ιούνιο για να συζητήσουμε πώς θα κινηθούμε περαιτέρω στον τομέα αυτό. Και εδώ πιστεύουμε ότι μια τέτοια συζήτηση μπορεί να είναι καθοριστική για σας αν ενδιαφέρεστε λοιπόν, είμαστε πρόθυμοι να ε, οργανώσουμε μια παρόμοια ε, συνάντηση και πιστεύουμε ότι η προώθηση αυτού του συστήματος των εθνικών σημείων επαφής θα ήταν πολύ θετικό στοιχείο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κ. Ζεγόμ Σαπλιέ, εργάζεται στον Ευρωπαϊκό Συνασπισμό για την Εταιρική Δικαιοσύνη. Το θέμα του σήμερα θα είναι πώς τα κράτη-μέλη ε, δρούν για να, προβλα... να προλάβουν την κατάχρηση και τις παραβέσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια επαγγελματική οικονομία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που θέλετε να ακούσετε τις, τη γνώμη τη κοινωνία των πολιτών για το πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη μπορούν να καταστήσουν σε επιχειρήσει πιο κοινωνικά υπεύθυνε. Και σε αυτό θα εστιάσω. Σε ό,τι αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η προστασία αυτή είναι βασικό στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη σημασία τα τελευταία χρόνια. Οι συνθήκε τη Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστούν σαφέ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την υποχρέωση να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τη όταν υιοθετεί και εφαρμόζει νομοθεσία, καθώ επίση και στι σχέσει τη με τον ε, υπόλοιπο κόσμο. Το 2011 η ο Οργανισμό των Εθνών υιοθέτησε ε, κατευθυντήρε γραμμέ για τι επιχειρήσει και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα κράτη-μέλη έχουν πλέον τη δυνατότητα να εφαρμο... Ε, την υποχρέωση να εφαρμόσουν αυτές τις κατευθυντήρε γραμμέ ε, μέσω κανονισμού και εθελοντική συμμετοχή πρωτοβουλειών. Το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σε ανακοίνωθέν της είχε αναφέρει ότι μέχρι το 2012 θα είχε δημοσιεύσει ένα πρόγραμμα δράσης τη Ευρωπαϊκή Ένωση για, τα, για τις επιχειρήσεις και ενθάρρυνε και τα κράτη-μέλη να κάνει το ίδιο. Πέντε χρόνια μετά ακόμα δεν έχει δημοσιευθεί αυτό το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα δράση. Ε, πιο θετικά όμως 13 ε, κράτη-μέλη δημοσίευσαν εθνικά προγράμματα δράση. 19 συνολικά σε όλο τον κόσμο. Ε, τρία, τρεις αδυναμίες βρίσκουμε σε αυτά. Πρώτον, παρόλο ότι βλέπουμε κάποια βελτίωση στα τελευταία ε, εθνικά πρόγραμματα δράση, Τις περισσότερες ε, φορές αυτά απλώς περιγράφουν την ισχύουσα κατάσταση, δεν δίνουν ε, πληροφορίε για τα μελλοντικά βήματα που θα αναλυφθούν. Δεύτερη αδυναμία, τα προγράμματα αυτά εστιάζουν κυρίως σε θελοντική συμμετοχή των επιχειρήσεων, σε δράσεις όπως κατάρτιση, έρευνα, ευαισθητοποίηση, πρόθεση βέλτιστων πρακτικών, ενημερωτικά εργαλεία κλπ. Γίνεται πολύ ε, ε, μικρή, επορισμένη σε ισχύω αναγνώριση ότι, ε, θα, ότι πρόκειται για υποχρεώσεις των εταιριών. θα, τρίτη αδυναμία, αυτά τα σχέδια αγνοούν την δυνατότητα προσφυγής ε, υπάρχουν ε, ε, σημαντικότατα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζουν τα θύματα προκειμένου να αποσφύγουν στη δικαιοσύνη. Είναι πρακτικά, διαδικαστικά, δικονομικά, οικονομικά και νομικά αυτά τα εμπόδια. Πολλά από αυτά τα εθνικά σχέδια δεν αναγνωρίζουν καν τη σοβαρότητα του προβλήματος και κανένα δεν δίνει ε, λύση στο θέμα της ε, δικαστικής προσφυγής. Αν λοιπόν αυτά τα εθνικά ε, προγράμματα δράσης δίνουν την εικόνα του πώς είναι η κατάσταση ευρωπαϊκή στα κράτη, αυτή η εικόνα είναι πραγματικά απογοητευτική, ανεπαρκής με ελάχιστες εξαιρέσεις δεν υπάρχει κανένα αντίστοιχη, καμία αντίστοιχη πρωτοβουλία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό αποδεικνύει την ε, έλλειψη εσωτερική πολιτικής ε, ε, ε, αποφασιστικότητας και δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλα λέει εντός και άλλα λέει εκτός των σύνορων της. Ορισμένες χώρες έχουν παρέμβει έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει. Εγώ τώρα εκπροσωπώ 21 ε, μέλη από 15 χώρες και θα ήθελα να σας κάνω μερικές προτάσεις για να βελτιωθεί το νομικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το θέμα. Ε, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων έχει αρμοδιότητα για αυτό το ζήτημα ε, και πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δείξει συνοχή και να αναλάβει τα ενία μιας παγκόσμιας προσπάθειας έτσι ώστε ο άνθρωπος να γίνει το κέντρο των προσπαθειών μας. Ε, η πρώτη μας ε, πρόταση ε, αφορά την υποχρέωση δέουσας επιμέλειας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε ό,τι αφορά αυτό, οι εταιρείε αυτές τις στιγμές έχουν δομή πολύ περίπλοκη, πολλές εταιρείε. Και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να, ελέγχεται, να ελέγχονται οι φθηγατρικές τους, οι προμηθευτές τους κλπ. Ο πρόεδρος παρακαλεί τον ομιλητή να μιλάει λίγο πιο αργά. Αυτή η νομοθεσία περί δέουσας επιμέλειας ε, είναι, αναγνωρίζεται ότι ε, δίνει ε, ένα πλαίσιο και κάποια κίνητρα σε για να εξασφαλίζουν την, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις δραστηριότητε τους. Και ε, η εταιρική ευθύνη μετατρέπεται σε μια νομική υποχρέωση με αυτόν τον τρόπο ε, έτσι ώστε να, οι εταιρείε να δείχνουν μια δέουσα προσοχή ε, όταν δρούν οικονομικά και συνεργάζονται με άλλες επιχειρήσεις. Αυτή η νομοθεσία διευρύνει το πεδίο εφαρμογή της δέους επιμέλειας στις θηγατρικές και στους επιχειρηματικούς συνεργάτες των εταιριών. Εξετάσαμε τις αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το θέμα και από ό,τι φαίνεται ε, είναι λογικό, δείχνει να είναι λογικό και δυνατό από νομικής πλευράς η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση σε αυτό το τομέα. Ο συνδυασμός του άρθρου 50 με το άρθρο 114 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εναρμονίζει την νομοθεσία προκειμένου να διασφαλίζει ότι θα λειτουργεί σωστά η εσωτερική αγορά. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν επανειλημμένω ερμηνεύσει τι συνθήκε έτσι ώστε να δίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια ευρία αρμοδιότητα να εναρμονίζει τι οικονομικέ και τι νομικέ υποχρεώσει ε, των επιχειρήσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα παράδειγμα. Οπότε ε, το σημαντικό είναι να εξασφαλίζουμε τα, τις ίδιες, τα ίδια πρότυπα ευθύνης για την, ε, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις εταιρείες των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες της γαλλικής νομοθεσίας που είναι η πρώτη η οποία μετέφερε σε, ε, στον αστικό της ε, κώδικα ε, την, το, την υποχρέωση δέουσα επιμέλεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι πραγματικά πρωτοπορή η Γαλλία. Αυτός ο νόμος καθορίζει την ε, αστική ευθύνη για βλάβες που θα προκληθούν από μια εταιρεία η οποία δεν έχει δείξει την δέουσα επιμέλεια. Μια, ένας κατάλογος ε, μεταρρυθμίσεων ε, στη Γερμανία, τη Βρετανία και λοιπά έχουν, έχει ήδη δημοσιευθεί, όλο και περισσότερες χώρες αναλαμβάνουν δράση και στις κάτω χώρες θα υιοθετεί πολύ σύντομα ένα παρόμοιο νόμο δέουσας επιμέλειας. Πιστεύουμε ότι είναι υποχρέωσή μα να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτές τις εξέλιξεις και να μειώσουμε ε, τον κίνδυνο δραματικών γεγονότων στα οποία θα εμπλέκονται ευρωπαϊκέ εταιρείε. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν μπορεί να δράσει και πρέπει να δράσει έτσι ώστε να μειωθούν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ευρωπαϊκές εταιρείες. Καλό λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, κάνει ξανακάνει έκκληση να αναλυφθεί δράση, να ενθαρρύνει την Κομισιόν και να γίνει το ίδιο ε, ο χώρος για ένα πραγματικά υγιή διάλογο. Τώρα, δεύτερη πρόταση που κάνουμε είναι οι συλλογικέ προσφυγές. Ξέρουμε ότι οι ε, προσφυγές ε, είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει σε μια ομάδα ατόμων που έχουν βλαθεί από τις ίδιες παράνομε πρακτικές να ζητήσουν ε, την ε, πάυση τους και αποζημίωση. Αυτό θα αντιμετώπιζε το πρόβλημα του υψηλού κόστους που θα είχε το κάθε άτομο χωριστά να προσφύγει στην δικαιοσύνη. Ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρώπης, συγγνώμη, το ε, Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν, έχουν υποδείξει ότι μια τέτοιου, ένα τέτοιο σύστημα συλλογικής προσφυγής θα ήταν χρήσιμο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013 σύστησε και ενθάρρυνε τα κράτη-μέλη να προβλέψουν τέτοιου είδους συλλογικές προσβάσεις σε όλες τις περιοχές όπου ε, γίνονται παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή και η Επίτροπος Γιουροβά τον Οκτώβριο του 2017 ανακοίνωσε ότι η τέτοιου είδου δυνατότητα για τους πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητηθεί στο πλαίσιο ενός προγράμματος New Deal για τους καταναλωτές που θα δημοσιευθεί το Μάρτιο 2018. Το πρόβλημα όμως της, ε, του περιορισμού ε, αυτών των συλλογικών προσφυγών σε θέματα καταναλωτών ε, είναι ότι υπάρχουν και άλλες περιοχές τις οποίες οι κακοί κακές πρακτικές από πλευράς των επιχειρήσεων μπορούν να αποδειχθούν ως επιβλαβείς σε τομείς όπως το επιχειρηματικό δίκαιο, το περιβαλλοντικό δίκαιο και τα θεμελιώδη δικαιώματα όταν για παράδειγμα γίνεται παράνομη μόλυνση, συστηματική διάκριση ε, ή κατάχρηση των εργασιακών δικαιωμάτων, ε, παραβιάσεις ε, του, της ιδιωτικότητας στον κυβερνοχώρο κλπ. Όλες αυτές είναι προκλήσεις που όταν κάποιος θέλει να προσφύγει στη δικαιοσύνη έχει ψηλό κόστος και μόνο οι συλλογικές προσφυγές θα μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα. Είμαστε πεπισμένοι λοιπόν ότι χρειάζεται και αναλυθεί ε, δράση για να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει οι κανόνες να εναρμονιστούν και οι ε, νομοθετικές ε, υποθέσεις, πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε κατακαιρματισμό της νομοθεσίας. Ενθαρρύνουμε λοιπόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καλέσει την Γενική Διεύθυνση Justice ε, το, στο μέλλον η, η νομοθεσία περί συλλογικών προσφυγών να κατοχυρώνει ε, τα, τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην, για την παραβίαση οποιοδήποτε θεμελιωδών ή ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα τελειώντας να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει πολλές ε, δεσμεύσεις τα τελευταία χρόνια σε διεθνές επίπεδο ε, και έχει ενθαρρύνει και τον υπόλοιπο κόσμο ε, να αναλάβει δράση. Πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει τα λόγια της πράξη και να θέσουμε το, στο επίκεντρο την ε, ε, αποφυγή ε, επεισοδίων όπως του Ράνα Πλάζα, του ατυχήματος του Ράνα Πλάζα που είχε πάνω από χίλια θύματα. Επίσης εταιρείε στην Ινδία, την Ιγυρία ή και τη Ρουμανία που με τις πρακτικές τους καταστρέφουν ολόκληρες κοινωνίες ή οικοσυστήματα όπως επίσης ακόμα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την παρόν χρήση εργατικού δυναμικού στη Γεωργία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο τελευταίο ομιλητής μα είναι ο κ. Αλέν Ντέκερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι τμήματάρχη στη Γενική Διεύθυνση ΦΙΣΜΑ ε, λογιστικά και οικονομικέ εκθέσει. Θα μα πει τι μπορούμε να, να αναμένουμε από τι καθεντήριε γραμμέ για την υποβολή μη οικονομικών εκθέσεων. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και την Επιτροπή σα για την ε, πρόσκληση στην Κομισιόν να συμμετάσχουμε. Η ομιλία μου αφορά τις κατευθύνσεις γραμμές της Κομισιόν για τις μη οικονομικέ εκθέσει. αλλά θα το διευρύνω λιγάκι για να θέσω αυτές τις ε, κατευθύνσεις γραμμές σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Την εφαρμογή της οδηγίας για τι μη οικονομικέ πληροφορίε και την ευρύτερη συζήτηση που γίνεται για το θέμα της ε, μη οικονομικής ε, αποστολής στοιχείων. Η οδηγία αυτή είναι κυρίως ένα μέσο διαφάνειας δεν ε, επιβάλλει υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις, απλώς ζητάει να παρουσιάσουν και να κάνουν εκθέσεις ή επιχειρήσεις για τις πολιτικές τους και τις πρακτικές τους. Και φυσικά συμφωνώ με τους προηγούμενους ομιλητές ότι η διαφάνεια είναι βασικό στοιχείο της εταιρική ε, κοινωνικής ευθύνης. Η οδηγία αυτή ενεκρίθη το 2014 και μεταφέρθηκε στο Εθνικό Δίκαιο έπρεπε να μεταφερθεί μέχρι το τέλος του 16. Οι μη δεσμευτικέ καθεντήρε γραμμέ υιοθετήθηκαν τον Ιούνιο και οι πρώτε εκθέσει που θα πρέπει να μα στείλουν οι εταιρείε θα δημοσιευθούν το 2018. Δηλαδή, η οδηγία νομίζω ότι είναι όντως σημείο τομής για την ενίσχυση της ε, διαφάνειας ε, της λειτουργίας των εταιρεών, αλλά ακόμη είναι νωρί για να δούμε τι επίπτωση θα έχει η εφαρμογή τη οδηγία στο μέλλον. Τώρα, το πεδίο εφαρμογή. Τι καλύπτει η οδηγία και ποιου καλύπτει. Η οδηγία απαιτεί οι εταιρείε να δημοσιοποιούν πληροφορίε για μια σειρά θεμάτων μεταξύ των οποίων περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, ανθρώπινα δικαιώματα, μέτρα κατά καταπολέμησης διαφθοράς και των δολοκιών και ε, η πολυμορφία του προσωπικού του σε σχέση με την ηλικία, το φύλλο, την, ε, το έθνος και πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας τους, για τις πολιτικές τους, δέωση επιμέλεια, τι επιπτώσεις έχουν αυτές οι πολιτικές, οι κύριοι κίνδυνοι που σχετίζονται με τα θέματα αυτά και επίσης μερικοί βασικοί δείκτες μη οικονομικοί για τα θέματα αυτά. Όχι μόνο απαιτείται να δημοσιοποιούν πληροφορίες για τις πολιτικές τους, αλλά η οδηγία απαιτεί οι επιχειρήσεις να μας πούν και αν δεν έχουν πολιτικές για κάποια από τα θέματα που καλύπτει. Αν κάποιες εταιρείε, για παράδειγμα, δεν ασχολούνται με τα θέματα αυτά, δεν μπορούν να μην μας πούν τίποτα. Το θέμα αυτό πρέπει να αναφερθεί και να αναφερθεί ότι δεν κάνουν τίποτα. Ποιες επιχειρήσεις καλύπτει καλύπτει τις κοινοφελείς ε, επιχειρήσεις, τις εισηγμένες, ε, τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές άνω των 500 εργαζομένων ως μέσο, κατά μέσο όρο κατά διάρκεια του έτους. Τα κράτη-μέλη μπορούν να προσθέσουν και άλλες κατηγορίες εταιριών που μπορεί να θεωρηθεί ότι ε, η λειτουργία τους έχει σημασία για το κοινό συμφέρον. Δηλαδή, οι εταιρείε αυτές είναι περίπου 6, είναι μεταξύ 6 και 10.000. Θα, θα εξαρτηθεί και από το ποιε εταιρείε και επιχειρήσεις θα προσθέσουν τα κράτη-μέλη στον ορισμό. Και επειδή υπάρχει μία χώρα που δεν έχει ακόμη μεταφέρει το νομοθέτημα και δεν έχει υιοθετήσει και εθνικά μέτρα εφαρμογή, υπάρχει κάποια αβεβαιότητα. Αυτή τη στιγμή μελετάμε τα μέτρα εθνικής εφαρμογής αναλυτικά. Αύριο, για παράδειγμα, συμμετέχω σε μια εκδήλωση που οργανώνουν ε, ορισμένοι οργανισμοί, όπου θα υποβάλουν μια έκθεση που έκαναν για την εφαρμογή της οδηγίας ακριβώς. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον λοιπόν για την οδηγία μεταξύ διαφόρων σημαντικών συμμετεχόντων στην ευρωπαϊκή οικονομία. Τι προσπαθούμε να επιτύχουμε με αυτές τις ε, μελέτες. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να καταλάβουμε εάν τα κράτη-μέλη έχουν σωστά νομικά μεταφέρει τις απαιτήσει οδηγία, Αλλά θέλουμε επίση να καταλάβουμε καλύτερα πώς έχουν μεταφέρει τις προϋποθέσεις και απαιτήσει. Για παράδειγμα, υπερέβησαν τα όρια τη οδηγία. Πώς ε, χρησιμοποίησαν τη δυνατότητα να επιτρέπεται στι εταιρείε να δημοσιεύουν χωριστά αυτές τις πληροφορίες ή αν θα πρέπει να είναι μέσα στον απολογισμό της εταιρείας. Πώς αντιμετωπίζουν θέματα όπως ε, τον ελεγκτικό έλεγχο και την μακροπροληπτική ευθύνη. Έτσι θα δούμε τι επίπτωση μπορεί να έχει οδηγία. Υπάρχει τώρα έντονη συζήτηση γύρω από τα θέματα αυτά σε διάφορα πλαίσια. Ένα από τα θέματα που συζητιέται πολύ είναι το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Όπως ξέρετε, η ειδική ομάδα με επικεφαλής τον Μάικλ Μπλούμπεργκ δημοσίευσε συστάσεις για ε, τις οικονομικές πληροφορίες ε, που αφορούν την κλιματική αλλαγή τον Ιούνιο και προσπαθούμε να περάσουμε κάτι παρόμοιο και στη δική μας ε, οδηγία. Επίσης, υπάρχει η υψηλή επίπεδο ομάδα εμπειρογνωμόνων για το θέμα της βιώσιμης ε, χρηματοδότησης και περιμένουμε την έκθεση της ομάδας αυτής μέχρι το τέλος του 2018 και υπάρχει και μια ευρύτερη συζήτηση μεταξύ διαφορών φορέων και επιχειρήσεων για το ρόλο των διαφόρων πλαισίων για υποβολή εκθέσεων που έχουμε μέχρι στιγμής. Η οδηγία βασίζεται ηθελημένα σε αρχές. Δεν θέλει να επιβάλλει συγκεκριμένο τρόπο υποβολής εκθέσεων, και η συζήτηση συνεχίζεται για το αν χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνηση ή σύγκληση των πλαισίων υποβολής εκθέσεων. Τι περαιτέρω θα μπορούσε να γίνει για συγκεκριμένους δείκτες ή τι παραμέτρους ε, ποσοτικές μπορούμε να καθορίσουμε. Μία δυσχέρεια είναι ότι επειδή καλύπτει πολύ ευρύ φάσμα η οδηγία, ε, θα μπορούσε από τομέα σε τομέα να είναι πολύ διαφορετικές ε, οι παράμετροι ή οι δείκτες. Για παράδειγμα, μια πετρελαϊκή εταιρεία θα έχει πολύ διαφορετικές ε, παραμέτρους από μια εταιρεία στον τομέα της ένδυσης. Χρειάζεται λοιπόν πολύ τεχνική δουλειά για τον τομέα αυτό, για το θέμα αυτό. Η οδηγία επίσης προβλέπει αναθεώρηση. Η νομικά δεσμευτική προθεσμία είναι η 6η Δεκεμβρίου 18. Το μεγάλο θέμα όμως είναι εάν θα έχουμε επαρκή στοιχεία μέχρι τότε για να έχει έννοια μια αξιολόγηση της εφαρμογής της οδηγίας. Όπως σας είπα, οι πρώτες εκθέσεις δεν θα δημοσιευθούν από τις επιχειρήσεις μέχρι του χρόνου. Και αν οι επιχειρήσεις αποφασίσουν να υποβάλουν χωριστές εκθέσεις για τα στοιχεία αυτά, κάτι που επιτρέπει η οδηγία, οι πληροφορίες αυτές υπάρχει δυνατότητα να ε, δημοσιευθούν ακόμη και έξι μήνες μετά την υποβολή του ισολογισμού. Δηλαδή μερικές τέτοιες εκθέσεις μπορεί να δημοσιευθούν το τρίτο τέταρτο του 18. Αν γίνει αυτό, θα έχουμε μόνο ένα χρόνο ε, εκθέσεων και πολύ λίγο χρόνο για να τις αξιολογήσουμε. Υπάρχουν και άλλα θέματα που θα πρέπει να τα δούμε πολύ προσεκτικά το υπάρχουν πλαίσιο για υποβολή εκθέσεων. Για παράδειγμα, η Παγκόσμια Πρωτοβουλία για υποβολή εκθέσεων. Πώς θα συνδυαστούν με την εφαρμογή αυτής της οδηγίας, λοιπόν, τα διάφορα αυτά πλαίσια. Και η εφαρμογή των συστάσεων Bloomberg, τι επίδραση θα έχει στην εφαρμογή της οδηγίας. Πολλά πρέπει να κάνουμε, λοιπόν, για να εξολογήσουμε την εφαρμογή και τον αντίκτυπο της οδηγίας. Και άλλα θέματα αιωρώνται. Ορισμένοι λένε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ενοποιημένο πρότυπο υποβολής εκθέσεων που να περιέχει και τις οικονομικές και τις μη οικονομικές πληροφορίες. Η Νότια Αφρική, για παράδειγμα, είναι πρωτοπόρα σε αυτό το τομέα. Υπάρχουν λοιπόν μερικά παραδείγματα, αλλά αυτό θέτει περίπλοκα θέματα. Για παράδειγμα, ο ρόλος του ελέγχου της ποιότητας ε, αυτών των εκθέσεων, ο ρόλος των λογιστών δηλαδή. Και πολλά θέματα έχουν να κάνουν με την ψηφιοποίηση και άλλες τεχνολογίες που θα μας επέτρεπαν να υποβάλλονται αυτές οι εκθέσεις και για τα οικονομικά και τα μη οικονομικά με καινοτόμους νέους τρόπους για να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια των εταιριών και προς τους επενδυτές και προς άλλους. Πολλά λοιπόν πρέπει να γίνουν ακόμη όπως είπα, αυτή τη στιγμή ασχολούμεθα με την αξιολόγηση της εφαρμογής. Θα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά την εφαρμογή της οδηγίας και εν ευθέτω χρόνο είμαι σίγουρος ότι η Επιτροπή θα κάνει δημόσιες δηλώσεις για το τι περαιτέρω προτίθεται να κάνει από αυτού. Με συγκεκριμένα ποια μορφή όμως θα ήταν πρόωρο να σας πω σε αυτή τη φάση. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. τώρα είναι η σειρά των βουλευτών να θέσουν ερωτήσει αν έχουν. Thank you. I, um... Η κυρία Χάουταλα, ευχαριστώ. Έχω κάποιες ερωτήσεις, αλλά πριν από αυτό, αν μου επιτρέπετε, ως ε, ιδέα που προέκυψε από όλες τις συζητήσεις που ακούσαμε, πιστεύω πως η Επιτροπή μας είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σταυροδρόμι και θα πρέπει να, να λάβουμε την πρωτοβουλία να εξετάσουμε τη δυνατότητα νομοθέτησης ώστε να ενισχύσουμε την εσωτερική αγορά για τη δέουσα επιμέλεια των εταιριών και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Εάν το κάνουμε, αν δεν το κάνουμε αυτό, πιστεύω η Επιτροπή δεν ε, φαίνεται να είναι αρκετά εμπνευσμένη. Αυτή είναι λοιπόν η ταπεινή μου πρόταση, ώστε να τη συζητήσουμε πιο μετά. Έχω όμως ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πολύ για τις ε, πολύ εμπνευσμένες σας εισηγήσεις. Όσον αφορά αυτό το BIAC, το η ομάδα εργασίας ε, το, που εσείς αντιπροσωπεύετε, εσείς των εργοδοτών. Έχω κάποια εμπειρία από τα εθνικά σημεία επαφή. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν κάποια πρότυπα για το πώ ε, στείνονται αυτά τα εθνικά σημεία, γιατί συχνά δεν έχετε ανεξάρτητου ανθρώπου, ανεξάρτητα άτομα που δεν εμπλέκονται με τη μία ή την άλλη πλευρά. Μπορείτε αυτό να το σχολιάσετε. Πιστεύω ότι η Νορβηγία έχει ε, πολύ καλό μοντέλο που θα μπορούσαμε να μεθούμε ώστε να λειτουργεί το σύστημα παραπώνων ή καταγγελιών. Δεύτερον, θα ήθελα να ρωτήσω τη συλλογική αποζημίωση. Αυτό απευθύνεται στον Ζεράρ Σαπλιέ. Όταν η Επίτροπος Γιούροβα ε, Ξεχωρίζει με αυτή την πρόταση που σχετίζεται με την προστασία του καταναλωτή και λέει ότι υπάρχει δυνατότητα διεύρυνσης ώστε να ε, ε, δώσουμε έναν πρακτικό τρόπο πρόσβασης της δικαιοσύνης για τα θύματα των πολυεθνικών ομίλων. Έχετε μια ιδέα για το πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Is that all, Mrs. Αυτά μόνο, κυρία Χάουταλα. Πολύ ωραία. Μπορώ να πω κι άλλα, αλλά εντάξει. Η κυρία Ρέγνερ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ε, παρουσιάσεις που μας κάνατε. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα ε, να σας ακούμε, ώστε να έχουμε μια ευρεία εικόνα. Ο καθένας από εσά εστιάζει σε κάτι άλλο και έτσι έχουμε πραγματικά μια πολύ ε, γενική ενημέρωση και εικόνα για το θέμα ερώτησή μου προς την κυρία Γκρανζόν σε σχέση με αυτό που παρουσίασε ο κύριος Τέκα Ντέκερς δηλαδή διαφάνεια και υποχρεώσεις ε, για αναφορές για τα μη οικονομικά θέματα όλα αυτά ε, όλες αυτές οι αναφορές και τα μεταθέματά τους και οι κατευθύνες γραμμές, σε ποιο βαθμό αυτά χρησιμεύουν για τα όσα έχει κάνει η Γαλλία. Με ενδιαφέρει πολύ σε ποιο βαθμό αυτές όλες οι αναφορές χρησιμεύουν. Βοηθούν στην επίτευξη του στόχου, ώστε όντως να ε, αναλαμβάνουν περισσότερε ευθύνε οι εταιρείε. Δεύτερη μου ερώτηση, εγώ τη συσχετίζω με αυτά που εσείς παρουσιάσατε προς τον κύριο Γκβάτφλιχ. Σας άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά και θα ήθελα να γνωρίζω πώς εσείς κρίνετε και βλέπετε αυτό που κάνει η Γαλλία, το γαλλικό τρόπο δηλαδή, να ζητήσουμε από τις εταιρείε να αναλάβουν αυτή την υποχρέωση. Τι σημαίνει αυτό για σας, εσείς θεωρείτε πως βοηθάει, θεωρείτε ότι είναι φόρτος, βάρος, ώστε να έχουμε κάπως πιο πλήρη εικόνα και να συνδυάσουμε λίγο τις παρουσιάσεις σας. Ο κύριος Κοφεράτη. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους ε, φιλοξενούμενους μας για τα όσα μας είπαν, για το γενικό, τη γενική εικόνα που σχεγράφησαν. Πιστεύω και όχι μόλις τώρα πως η διαφάνεια, η διαφάνεια και η ευθύνη των εταιριών είναι αυτές που προσφέρουν ε, αγαθά Ακόμα και αυτές που ασχολούνται μόνο με χρηματοπιστωτικά θέματα απλά. Και το απλά, εντάξει, δεν είναι και τόσο απλά. Ε, εν πάση περιπτώσει, το σημαντικό είναι η προστασία των Ευρωπαίων πολιτών, τόσο όταν είναι καταναλωτές, όσο και όταν είναι παραγωγή. Τα επιχειρήματα τα οποία περιλαμβάνονται στη διαδικασία εταιρικής ευθύνη, κοινωνικής εταιρικής είναι λοιπόν πολύτιμα. Το πρόβλημα ωστόσο δεν λύνεται ούτε και με τις συζητήσεις που κάναμε τα τελευταία χρόνια στο εσωτερικό εδώ του Κοινοβουλίου και πιστεύω ήταν να θεσμοθετήσουμε την λογοδοσία την κοινωνική. Αυτή θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική για τις εταιρείε ή θα πρέπει να παραμείνει επί της εθελοντικής βάσης που έχει σήμερα τα βήματα που έχουν γίνει σε αυτή την υπόθεση είναι λίγα. Είναι μικρά. Το θέμα της εταιρικής ευθύνης ε, ήδη άρχισε να συζητιέται από το απόμακρο 1993 και σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου γίνονται πολλές προσπάθειες αλλά αποτελέσματα ισχνά. Όσοι έχουν τώρα οι κανόνε. οι, εταιρείε οι εταιρείες διακινδυνεύουν μόνο τη φήμη του. Τυπώνουν ένα ωραιότατο τόμο όπου συνοψίζουν την εταιρική του ευθύνη. Τώρα αν όλα αυτά είναι βάσιμα ή όχι, κανείς δεν ξέρει. Αν παραβιαστούν, ε, θα χάσει λίγη αξιοπιστία η εταιρεία, αλλά τίποτα περισσότερο. Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων λοιπόν από το 1993 μέχρι σήμερα, εταιρείε που είχαν επενδύσει πολύ στην κοινωνική ευθύνη, έπειτα έγιναν υπεύθυνε για καταστροφικές επιπτώσεις των ενεργειών τους, ας πούμε, όπως οι πετρελαϊκές εταιρείε, οι οποίες ε, μόλι ρήπαναν τη Βόρεια Θάλασσα, γιατί ε, ε εξορίγνιαν πετρέλαιο στη Βόρεια Θάλασσα και μετά βούλιαξαν καράβια, βούλιαξαν πετρελοφόρα ενώ διατυμπάνιζαν την υποστηθέμενη κοινωνική τους ευθύνη δεν έκαναν τίποτα στη συνέχεια. κατά τη γνώμη σας λοιπόν θα έπρεπε να καταστεί υποχρεωτική η λογοδοσία κοινωνική ή όχι. Ε, αυτό το καταλαβαίνω, ε, αλλά δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι θα πρέπει να γίνει τελικά. Και έπειτα πιστεύω ότι θα ήταν καλό να επιβληθούν και κάποιες κυρώσεις. Δεν θα, έστω και το να δημοσιευθεί η απομάκρυση από τα όσα έχει δηλώσει η εταιρεία και τα όσα έκανε δηλαδή στην πράξη. Γιατί το να συντάσσουμε ορότατες εκθέσεις κοινωνικής ευθύνης, αυτό μπορεί να ε, γίνει μέσω αθέμητου ανταγωνισμού που σε αυτή την ε, περίοδο στην οικονομία μας ε, προτάσσονται. Λένε τι ωραία που σέβονται το περιβάλλον, λένε πόσο σέβονται τα δικαιώματα των ανθρώπων και μετά στην πράξη κάνουν άλλα Άρα λοιπόν όποιος παραβιάζει τους όρους του παιχνιδιού θα πρέπει να τιμωρείται. Ίσως λοιπόν σε κάποιο πιο απόμακρο ε, μέλλον θα πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχει μια υποχρέωση και υπάρχει και η τιμωρία ή η κύρωση. Και άλλωστε οι κυρώσεις μπορεί να παίξουν αποτρεπτικό ρόλο, πολύ σημαντικό όπως γνωρίζουμε. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ποια είναι η, θέση, η γνώμη σας σε σχέση με αυτή την υπόθεση που λίγο απέχει από την πραγματικότητα, αλλά που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα ο κύριος Λεμπρετό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω όλους ε, όσοι ήρθαν εδώ να μας ε, διαφωτίσουν. Το θέμα αυτό είναι, έχει σχέση με τις πολυεθνικές. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί κανείς ε, ε, αναρωτιέται αν δημιουργείται ένα σύστημα δύο ταχυτήτων. Αφενό, οι επιχειρήσεις επιχειρήσει, οι μεμονωμένοι ε, επιχειρηματίε, ε, ε, οι οποίοι διέπονται από ένα σκληρό νομοθετικό πλαίσιο, και από την άλλη μεριά οι, ε, ε, οι πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες δεν υπακούν κατά βάση κανένα νόμο. Μιλούμε για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και τελικά τι είναι. Πρόκειται για έναν τρόπο να ε, βελτιστοποιήσουμε κοινωνικά τον ε, υπέρμετρο φιλελευθερισμό. Καλό είναι να καταλάβουμε λοιπόν τι συμβαίνει και να δράσουμε. Είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να βρούμε λύσεις soft ε, νομοθεσίας, ε, ε, ήπιας νομοθεσίας. Ε, εμείς προτιμάμε τη σκληρή νομοθέτηση, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας. Νομίζω ότι πολύ σωστά αναζητούμε την διαφάνεια και μίλησαν όλοι οι παρεμένοντες, όλοι οι ομιλητές γι' αυτό. Διαφάνεια στις πολυεθνικές εταιρείε. Ε, γιατί θα μας δώσει την ευκαιρία να τις αναγκάσουμε να προχωρήσουν. Πέραν όμως αυτών των πρακτικών ενθάρρυνσης και ήπιας νομοθεσίας, ε, πέραν από το γεγονός ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε πιο σκληρή νομοθεσία, ε, εσείς ε, Πότε πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε μια τέτοια κατάσταση. Ε, δεύτερον, σε ό,τι αφορά την ήπια νομοθεσία, θα μπορούσατε να μου πείτε για αυτά τα εθνικά σημεία επαφή, ποια είναι τα πιο αποτελεσματικά. Εγώ είμαι Γάλλο. για παράδειγμα, το γαλλικό σημείο επαφή είναι αποτελεσματικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Ντυρό. Ένα Γάλλο μετά από ένα άλλο Γάλλο. Κάτι του σπανίως συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να πω στον κύριο Λεμπρετό ότι θα ήθελα να επιχειρηματολογήσει το γιατί μόνο οι πολυεθνικές εταιρείε είναι υπεύθυνε για την σημερινή κατάσταση σε όλο τον πλανήτη. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν νομίζω ότι φταίνε μόνο οι πολυεθνικές εταιρείε. Και ορισμένε εθνικέ ε, εταιρείε που έχουν τη δυνατότητα να ε, δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο και έχω και παραδείγματα χαλικών εταιριών που έχουμε δει στη Βερμανία και αλλού έχουν δυνατότητα να δρουν ε, με τρόπο που αντιβαίνουν στους ε, ε κανόνες οι οποίοι επιβάλλονται στη Γαλλία. Για μένα η περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη πέραν του αν θα είναι υποχρεωτική ή όχι είναι ηθικό ζήτημα που, θα πρέπει να το έχουμε ήδη ξεπεράσει στις ισχυρές χώρες. Το ερώτημα είναι, η αξία του ανθρώπου είναι η ίδια παντού σε όλο τον πλανήτη. Αυτή είναι η πραγματική ερώτηση. Όταν η Total ή κάποιε άλλες γαλλικές επιχειρήσεις ε, δραστηριοποιούνται στη Βερμανία ή αλλού, ε, τα κοινωνικά υπερβαλλοντικά πρότυπα ε, είναι ίδια με αυτά της Γαλλίας. Η, η, μια ε, συμπεριφορά ή κάποιες πρακτικές οι οποίες θα ήταν απαράδεκτες στη δική τους χώρα μπορούν να είναι δεκτές κάπου αλλού. Αυτή είναι η πραγματική ερώτηση. Δεν είναι δυνατόν η ερώτηση να είναι μόνο νομική, γιατί από νομικής ε, ε, πλευράς μπορούμε να τους πούμε φροντίστε οι, οι υπεργολάβοι σας να σέβονται την εθνική νομοθεσία του κράτους το οποίο δραστηριοποιείται. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Η πραγματική ερώτηση είναι ποια είναι η αξία που δίνουμε στην ανθρώπινη ύπαρξη και δεύτερον θα μπορούσαμε να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στην δέουσα επιμέλεια και στην ευθύνη. Για μένα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το συνταγματικό δικαστήριο στη Γαλλία κατέριψε το πρόστιμο, την πρόβλεψη του προστίμου, αλλά για μένα η δέουσα επιμέλεια είναι μια υποχρέωση κάποιο ε, να παρακολουθεί μια κατάσταση. Ενώ η κοινωνική ευθύνη είναι μια ευθύνη να πράξει κάποιο, να πάρει μέτρα. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αν μπορούμε να προχωρήσουμε, να σημειώσουμε πρόοδο και στο θέμα της υποχρέωσης. Όχι μόνο της δέουσας επιμέλειας. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις, λέει ο Πρόεδρος. Ίσως να ξεκινήσουμε από αριστερά, όπως κοιτάω εγώ την αίθουσα, με τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το νομικό χαρακτήρα της οδηγίας των εκθέσεων που θα υποβληθούν. Ε, δεν θα αναφερθώ σε άλλες πτυχές του δικαίου, που, εργασιακού δικαίου, δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δεν αποτελούν αρμοδιότητά μου. Να πω ότι αυτές οι εκθέσεις θα είναι υποχρεωτικές, ε, η οδηγία είναι δεσμευτική η οδηγία υποχρεώνει τις επιχειρήσεις ε, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή τη να δημοσιεύουν εκθέσεις. Και όχι μόνο τις υποχρεώνει, η οδηγία προβλέπει επίσης ότι τα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων έχουν νομική ευθύνη για την δημοσίευση. Αν δηλαδή ε, σε αυτές τις εκθέσεις υπάρχουν πληροφορίες ψευδείς ε, ή ανακριβείς, τότε είναι υπεύθυνο το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης. Και όλες οι κυρώσεις που προβλέπει η ανακριβης τοτε ειναι υπευθυνο το διοικητικο συμβουλιο της επιχειρησης και ολες οι κυρωσεις που προβλεπει η οδηγια για τα λογιστικά πρότυπα μπορούν να εφαρμοστούν, να επιβληθούν. Οπότε υφίσταται ένα σαφές και δεσμευτικό νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση στις, ε, στην υποβολή μη οικονομικών εκθέσεων. Ευχαριστώ. Κύριο Σαπλίε, για το θέμα της ε, πρότασης για τις συλλογικέ προσφυγές και για πώς αν μπορεί να διαβρυνθεί το παιδί Το θετικό είναι ότι ε, η βάση του, της σύστασης του 2013 αφήνει το περιθώριο στα κράτη-μέλη να, να υπερβεί ε, τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ε, μπορεί να, τα κράτη-μέλη να περιλάβουν και τα ανθρώπινα δικαιώματα και μάλιστα ενθαρρύνονται να το κάνουν. Δεν πρόκειται λοιπόν για θέμα νομικού εμποδίου αλλά πολιτικής βούλησης. Το ερώτημα είναι, ένας καταναλωτής που αγόρασε ένα αυτοκίνητο από τη Volkswagen θα πρέπει να έχει περισσότερες δυνατότητε συλλογική προσφυγής από ότι οι Ούγγροι και οι Ρουμάνοι ε, που έχουν μολυνθεί από Κιάνιο στο Δούναβι. Αυτό είναι το ερώτημα και η Γενική Διεύθυνση Justice έχει κάνει πολύ λίγα πράγματα ε, για αυτό το ζήτημα. Ε, για τον τρίτο πυλώνα, δηλαδή των κατευθυντήρων γραμμών του ΟΗΕ. Ίσως η Γενική Διεύθυνση Justice θα έπρεπε πράγματι να αλλάξει προσέγγιση. Ελπίζω δεν είναι αργά. Για το θέμα της ε, υπέρβασης του, της ε, ήπιας νομοθεσίας ε, που ρώτησε ο κ. Λεμπρετών, νομίζω ότι η, ε, όλη μου η παρουσίαση ακριβώς αυτό ζητούσε προφαρός προφανώς χρειαζόμαστε ε, ευφυείς, ήπιες νομοθεσίες, αλλά αυτή τη στιγμή με όλα όσα συμβαίνουν τελευταία δεκαετία υπάρχει μια τάση να μετακινηθούμε προς μια πιο αυστηρή νομοθεσία. Τώρα, κύριος Ντυρό, αν μπορούμε να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στη δέουσα επιμέλεια και την ευθύνη. Μπορούν, υπάρχουν πολλές, πολλοί τρόποι ε, να νομοθετήσουμε για την ε, δεούσα επιμέλεια. Ε, οι διαγωνισμοί, η νομοθεσία περιδεύουσας επιμέλεια κλπ. Νομίζω ότι η πιο καλή λύση είναι αυτή που ακολουθήθηκε στη Γαλλία. Είναι ένα μοντέλο αστικού, συνομοθεσίας νομοθεσία αστικού δικαίου που επιτρέπει στους ε, ε, βλαφθέντες να προσφύγουν στο δικαστήριο. Ευχαριστώ. Κύριος Γουάντφλικ. ευχαριστώ Πρόεδρε. Μερικά από τα ερωτήματα θα έχριζαν ε, μακροσκελούς αντιμετώπισης, αλλά θα είμαι σύντομος. Θα έπρεπε να υπάρχει μια τυποποιημένη προσέγγιση βεβαίως από πλευράς των επιχειρήσεων. Ο καλύτερος τρόπος, αν υπάρχει περισσότερη υποποίηση, θα ήταν καλό. Αλλά πώς θα προκύψει αυτό. Υπάρχει μια διαδικασία στον ΩΣΑ εδώ και χρόνια με την αποτίμηση μεταξύ ομοτήμων για την ε, ε, καλύτερη εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να τα επιβάλλουμε είναι καλύτερα να τα επιβάλλουμε ή καλύτερα να επιτρέψουμε να γίνει με φυσιολογικό ας πούμε αυτόματο τρόπο η ανάπτυξή του. Το γαλλικό σύστημα λειτουργεί καλύτερα από τα άλλα. Ποια είναι η γνώμη μας για το γαλλικό νόμο επ' αυτού. Θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά όπως εξήγησα στην παρουσίασή μου, τα προβλήματά μας είναι ότι είναι υποχρεωτική η γαλλική προσέγγιση και υπάρχει κίνδυνος διάδοσης. Ε, υπάρχει ο γαλλικός νόμος, αλλά τώρα υπάρχει και ο ολλανδικός που θα εγκριθεί σε λίγο και ο ελβετικός, άρα εάν υπάρχουν πολύ διαφορετικά εθνικά πρότυπα, θα είναι πολύ δύσκολο στις εταιρείε να συμμορφωθούν. Η φιλοσοφία του γαλλικού νόμου βασίζεται στις κατευθύνες γραμμές και τις αρχές. Η πιο δύσκολη ερώτηση. Θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική αυτή η υπεύθυνη συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Μα ακριβώς ε, πρόκειται ε, για το ότι είναι θελούσια. Υπάρχουν πολλοί νόμοι στον κόσμο. Οι επιχειρήσεις που έχουν καλή θέληση το, εφαρμο, το εφαρμόζουν. Υπάρχει ποινικό δίκαιο, οικονομικό δίκαιο, πολλά στοιχεία εφαρμογής αυτών των νόμων αποτελούν υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά και είναι υποχρεωτική. Ο λόγος για τον οποίο αυτό που τώρα αποκαλούμε υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά δεν είναι υποχρεωτικός είναι επειδή τίθενται θεμελιώδη θέματα. Για παράδειγμα για την ε, εξοεδαφικότητα. Ένα δημοκρατικό σύστημα πάντα μπορεί να πει ότι θέλουμε για τα α, β, γ θέματα υποχρεωτική νομοθεσία. Αλλά τότε δεν είναι υπεύθυνη η εταιρική συμπεριφορά, είναι απλώς η μόρφωση με τον νόμο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι θεμελιώδες στοιχείο της ε, υπεύθυνης συμπεριφοράς το να είναι θελούσια και είναι παντού ρωτηθήκαμε η ίδια η ανθρώπινη συμπεριφορά. Ναι, σε αυτό βασιζόμαστε. Ναι, ότι κάθε ανθρώπινο όν έχει την ίδια αξία. Και οι επιχειρήσεις συμφωνούν με αυτό. και μπορούμε να διακρίνουμε την δέουσα επιμέλεια από την υπεύθυνη συμπεριφορά, πρέπει να τονιστεί ότι οι καθητήριες γραμμέ περιέχουν δύο βασικά στοιχεία. Πρώτον, ο συγκεκριμένο ορισμό της Ευθύνη. που είναι ότι πρέπει να αποφεύγονται ε, οι βλάβες και το άλλο είναι διαδικαστικό, που είναι η δέωση επιμέλεια. Η δέωση επιμέλεια υπάρχει μόνο αν υπάρχει ένας πιο συγκεκριμένος ορισμός, μια πιο συγκεκριμένη σύσταση, που επίσης υπάρχει χαρακτηριστήρες γραμμές. Ο κύριος Ρης, να με συγχωρείτε θα είμαι πολύ σύντομος γιατί πρέπει να φύγω, για τη διαφάνεια που αναφέρθηκε επανειλημμένα. Ναι. Αν έχεις ένα αξιόπιστο δημόσιο σύστημα, τότε οι άνθρωποι ανταποκρίνονται και υπάρχει συμπληρωματικό κίνητρο στις επιχειρήσεις για να συμμορφωθούν. Πολλοί αναφέρθηκαν στη σημασία της διαφάνειας. Βεβαίως, πρέπει να είναι και απόλυτα διαφανές, αλλά και ρωμαλαίο και να έχει ε, την αναγκαία σημασία για να προκαλέσει τη σωστή συμπεριφορά. Τώρα άλλοι ξέρουν καλύτερα από μένα το θέμα για το αν υπάρχει ανάγκη για να περάσουμε από ήπια, ήπια σε πιο δεσμευτική νομοθεσία. Σε πολλά δεν υπάρχει συνένεση από αυτού του θέματος, αλλά θα μπορούσα να πω ότι συζητούμε τα θέματα της υπεύθυνης εταιρική ε, συμπεριφορά, γιατί πολλοί εργαζόμενοι ζουν σε δικαιοδοσίες όπου δεν υπάρχει πολλή πρόσβαση στη δικαιοσύνη και δεν μπορούν εύκολα να ασκηθούν τα δικαιώματά τους. Άρα πρέπει να κοιτάξουμε τι άλλα μέσα υπάρχουν για να στηρίξουμε, να δώσουμε τη δυνατότητα προσφυγής και να στηρίξουμε το, τη διαδικασία ε, προσφυγής στη δικαιοσύνη ε, στις χώρες αυτές. Ευχαριστώ κυρία Καούζον. Ευχαριστώ. Πολλέ ερωτήσει για του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονε. Πιστεύω πω όντω είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σημείο επαφή όπω έχει φτιαχτεί στη Γαλλία και επιτρέπει τη χορήγηση συμβουλών, το συντονισμό. Είναι σημαντικό για να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτό το σχέδιο επαγρύπνησης και να συζητήσουμε και δείκτες. Διαφάνεια, ναι, είναι απαραίτητη ορατότητα, για την πραγματικότητα, για τα διακυβεύματα, για την καθετερία, διευκρίνηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλυφθεί και των μέσων που έχουν τεθεί στη διάθεση της επίτευξης των στόχων και έπειτα επικοινωνία για τα αποτελέσματα. Ε, γιατί διαφορετικά είναι δύσκολο να μετρηθούν και αυτά. Και έπειτα εξέλιξη των δεσμεύσεων, γιατί μπορεί να ακούσουμε ότι οι εταιρείε ε, ε, παίρνουν χρόνο σε σχέση με τις δεσμεύσεις ε, μήνες, ίσως και χρόνια να φτιάξουν ε, δράσεις. Μπορούμε να περιμένουμε, μόνο που πρέπει η εξέλιξη αυτή να αναπτύει με συγκεκριμένα μέσα, μετρήσιμα. Έπειτα, δυνατότητα προσφυγής. Και εδώ η ευθύνη για τις συνέπειες και αυτό είναι σημαντικό να το τονίσουμε γιατί οι συνέπειες. Μπορεί να προσπαθήσουμε να τις αποφύγουμε, αλλά να αποφύγουμε τις αρνητικές επιπτώσεις, όμως οι συνέπειες απαραίτητο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τις ίδιες τις εταιρείες. Φυσικά, κάποιες φορές θα ήταν ε, το ελάχιστο απαραίτητο αν υπάρχουν συνέπειες για, για έναν άνθρωπο ή αν είναι οι συνέπειες στο περιβάλλον, έπειτα για την ηθικότητα, την νομιμότητα. Είναι περίπλοκο για τον νομοθέτη να δουλέψει για την ηθικότητα. Η εφαρμογή της νομιμότητας επιτρέπει να έχουμε στοιχεία αναφοράς για να μπορούμε να προβούμε και σε ε, διαβήματα που να είναι κοινωνικά υπεύθυνα. Όσον αφορά την ευθύνη, θα ήθελα να επιμείνω στο στόχο των μέσων και μέσα από αυτό να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε ε, επιπτώσεις αρνητικές. Οι δεσμεύσει θα πρέπει επίση να είναι προσωπικέ, ε, πραγματικέ, νομικές, να έχουν συνέπειε. Η υποχρέωση λοιπόν είναι δεσμευτική και συνοδεύεται και επιτρέπει να ξεκινήσει κανείς σε προσφυγή. Και με βάση αυτές τις διάφορα, διάφορα στάδια ακολουθείται η ευθύνη από το δικό μας project. Ευχαριστώ. Κύριε Νέορκαμπ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάποιες παρατηρήσεις. Είμαι και Πρόεδρε του Εθνικού Σημείου Επαφής στην Ολλανδία, οπότε εξορισμού δουλειά μου και ως πρόεδρο της ομάδας εργασίας για να σχολιάσω τις καλές ή τις κακές πρακτικές των εθνικών σημείων επαφής είναι πάντοτε δύσκολο. Πάντως το γαλλικό σημείο είναι πολύ, λειτουργεί πολύ καλά, είναι τριμερές, δηλαδή οι εταιρείε και τα συνδικάτα είναι μέλη και γι' αυτό είναι επιτυχέ. Το νορβηγικό, δανέζικο και ολλανδικό μοντέλο είναι επίση πολύ καλά εγκαθιδρυμένα γιατί έχουν ανεξάρτητα μέλη το αβερετανικό μοντέλο επίσης είναι πολύ καλό που υπάρχουν ουδέτερα μέλη στο εποπτικό όργανο. Υπάρχει και ένα ανεξάρτητο εποπτικό σύστημα. Αυτά είναι τα τρία κύρια μοντέλα που έχουν δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα. Όταν αφορά αυτό το άλμα από το ήπιο στο ε, πιο ισχυρό δίκαιο, το θέμα εδώ είναι τι λειτουργεί Εάν περάσουμε από το ήπιο λοιπόν στο σκληρό δίκαιο, αυτό σημαίνει ότι το ήπιο δίκαιο δεν λειτουργήσε. Και γι' αυτό τόνισα ότι δεν ξέρουμε αν λειτουργεί ή όχι. Πρώτα θα πρέπει να αρχίσουμε να αξιολογούμε κατά πόσο το ήπιο δίκαιο λειτουργεί ή όχι. Αυτό θα κάνουν οι Γερμανοί τώρα πριν να κάνουν το άλμα, να περάσουν στο δίκαιο αυτό καθ' αυτό. Γιατί όπως σας είπα η πολιτική μέχρι στιγμής λειτουργεί χωρίς στοιχεία. Και αυτή η συζήτηση περί υποχρεωτικής ή εθελοντικής βάσης ε, ε, είναι στον αέρα κάπως. Εγώ πάντοτε θέλω να, πάντοτε λέω πρώτα να δούμε τι δουλεύει, τι λειτουργεί. Γι' αυτό και είπα και επέμεινα στο να, στο να επιμείνουμε στην παρακολούθηση, ποιες εταιρείες ξέρουν τις κατευθυντήριες γραμμές, ποιες τις ακολουθούν, ποιες γνωρίζουν ε, τη, τα σημεία επαφής. Όλα αυτά δεν έχουν εξεταστεί. Και γι' αυτό και το άλμα από το ήπιο στο δίκαιο, στο σκληρό δίκαιο, είναι θέμα τελείως υποκειμενικό για την ώρα. Μάλιστα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εξαντλήσαμε τώρα αυτό το ε, θέμα και την ακρόαση. Ε, Θέλω να ευχαριστήσω τους διακεκριμένους μας ομιλητές που ήταν σήμερα εδώ και μοιράστηκαν μαζί μας την εμπειρία τους. Επίσης, για όσους ήταν εδώ, ήταν πραγματικά ε, πολύ πλούσια η συζήτηση. Σας ευχαριστώ όλους. Και να κλείσουμε και τη συνεδρίασή μας μέσω με μια ανακοίνωση που όπως γνωρίζετε πολύ καλά αύριο έχουμε μια έκτακτη συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο. Το λεωφορείο μας φεύγει στις 7 το πρωί. 7 το πρωί παρακαλώ αναχώρηση. Ε, so I will be looking to meeting you looking forward to meeting you tomorrow morning uh, in, the bus. Uh, λοιπόν, η επόμενη μας τακτική συνεδρίαση, 28 Οκτωβρίου, κοινή συνεδρίαση Γιούρι Αύκο στις 11.45 εκείνη είναι η χρονοθυρίδα της Επιτροπής Αύκο και θα είναι αφιερωμένη στην εφαρμογή και υλοποίηση της Διοργανικής Συμφωνίας για την καλύτερη νομοθεσία και η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας θα γίνει στις 7 Δεκεμβρίου. Χαίρετε, αντίο σας.